Συνάδελφοι, καλημέρα σα. Αν θέλετε να πάρετε τι θέσει να αρχίσουμε τη συνεδρίασή μα. Έχουμε του καλεσμένου μα, οι οποίοι είναι παρόντες. Τον καθηγητή Τωμάζο Πάντο Ασκιώπα, ο οποίο ε, πρέπει να φύγει το πολύ στι 4, γιατί πρέπει να ε, προλάβει το αεροπλάνο, γιατί έχει ένα μεγάλο ταξίδι στην Ιαπωνία. Ehm, λοιπόν, να σα κάνω και ορισμένε ανακοινώσει προηγουμένω, αλλά πραγματικά δεν θα σα ε, κουράσω καθόλου, ε, γιατί θέλω να συνεχίσουμε τι εργασίε μα. Όπω ξέρετε, είχα ζητήσει από τον νέο ειδικό ε, απεσταλμένο αρχηγό τη αντιπροσωπεία τη Ευρωπαϊκή Ένωση στο Αφγανιστάν, τον κύριο Ουσάκα, Είχα ζητήσει λοιπόν μέσω της κυρίας Άστον να έρθει ε, στην Επιτροπή μας για μία ακρόαση και, το ίδιο πράξαμε και προς τον επικεφαλής της αντιπροσωπείας ε, στην Washington, Βάλεντε Αλμέιντα. Και ήθελα ε, αυτό να γίνει πριν να λάβουν τα καθήκοντά τους ε, οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι, ακριβώς για να, υπάρχει, να υπάρξει μια εξέταση, αν θέλετε, από το Κοινοβούλιο των προσωπικών του χαρακτηριστικών, των προσόντων του παρόλο που βεβαίω ε, που ο διορισμό έγινε στην ΥΠΑ το εκπρόσωπο, αλλά ξέρετε ότι και εμεί εκφράσαμε την επιθυμία και αναλαμβάνουμε βέβαια και την ευθύνη τουλάχιστον συμβουλευτικό επίπεδο να συμμετάσχουμε στη διαδικασία αυτή ε, της εκλογής. Ο κύριος Σουζάκας θα έρθει στις 23, Μαρτίου στις 5 η ώρα. Η συνεδρίαση στις 22 το απόγευμα ακυρώθηκε για να μπορέσουμε όλοι να συμμετάσχουμε στη συνεδρίαση της Επιτροπής ε, Ανάπτυξης με προσκεκλημένο τον ε, πρώην ε, Πρωθυπουργό της Βρετανίας, τον Ιμπλερ, για ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό. Και νομίζω ότι έπρεπε να αφήσουμε ελεύθερο το απόγευμα για να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε αυτή τη συνεδρίαση. Στις 23 Μαρτίου λοιπόν, στις 3 η ώρα, σας το υπενθυμίζω, προβλέπεται ανταλλαγή απόψεων με την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και είπα το εκπρόσωπο, την Βαρόνια Άστον. Η συνάντηση αυτή είναι πολύ χρήσιμη γιατί θα μπορέσουμε να συζητήσουμε την πρόταση δημιουργίας της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση, με τον Έλμαρ ε, Μπρόκ, ε, εισηγητή εκ μέρου τη Επιτροπή μα, για να είμαστε έτοιμοι και για το. Και, ε, μάλλον θα ακούσουμε την στο Συμβούλου Εξωτερικών την προηγούμενη ημέρα. Λοιπόν, έχουμε τώρα την έγκριση των πρακτικών συνεδριάσεων 26-27 Ιανουαρίου, 28 Ιανουαρίου και 4 Φεβρουαρίου. Αν έχετε να κάνετε κάποιες παρατηρήσεις, πριν τη λήξη σημερινή συνεδρίαση είμαστε στη διάθεσή σα. Διαφορετικά θα θεωρήσουμε ότι εγκρίθηκαν τα πρακτικά. Περνάμε τώρα στην ανταλλαγή απόψεων με τον ε, Τομάζο Πάντου Ασκιόπα και τον ε, κύριο Ντομινιόν για αυτή την τόσο ενδιαφέρουσα έκθεση με τίτλο «Χάρτης για μια νέα ευρωαμερικανική εταιρική σχέση». Έχουμε και την Νικόλ Γνεζότο, την ε, εισηγήτρια ε, την οποία επίσης καλωσορίζω και την ευχαριστούμε για, το, για την εργασία της. Ο καθηγητής Τομάζο Πάντα είναι πρόεδρος αυτής της ομάδας προβληματισμού υψηλού επίπεδου, του επίπεδου, όπου ανήκει και ο πρόεδρος Μπούζεκ, ο συνάδελφος Φερχόφστατ και άλλες εξέχουσες προσωπικότητες που διαθέτουν μακροχρόνια εμπειρία στην διεθνή πολιτική και έχουν, ε, κατέχουν ή κατήχαν ύψιστα αξιώματα στην κυβέρνησή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θέμα ε, είναι ιδιαίτερα επίκαιρο και πάρα πολύ σημαντικό λαμβάνοντας υπόψη ε, και το γεγονό ότι η συνθήκη τη Λισαβόνα ε, προσδίδει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα νέο, είδος, ένα νέο προφίλ. Ε, πρόκειται λοιπόν για μια αναγέννηση των δραστηριοτήτων μα σε εξωτερικό επίπεδο. Επίσης, η αλλαγή του Πρόεδρου στι Ηνωμένε Πολιτείε δημιούργησε νέε συνθήκε και ένα σενάριο ιδιαίτερα ενδιαφέρον, ακριβώς για να έχουμε αυτή την αναγέννηση των σχέσεων ανάμεσα στις δύο υπήρους. Και νομίζω λοιπόν ότι αυτό το ε, θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι με τον τρόπο αυτό μπορούμε ε, να έχουμε τις νέες προϋποθέσεις διαλόγου και μπορούμε να προτείνουμε, να προτείνουμε ένα καινούριο διάλογο, ένα καινούριο είδος διαλόγου ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα ακούσουμε λοιπόν τους εξέχοντες προσκεκλημένους μας Δεν θα κάνω άλλες εγωικές παρατηρήσεις για να μην στερήσω το χρόνο ε, από του ε, ομιλητές μας. Είναι πολύ ενδιαφέρον ο διάλογο και να δώσουμε το λόγο στον Πρόεδρο Πάντο Ασκιώπα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι μεγάλη χαρά που βρίσκομαι εδώ σήμερα. Φιλοξενούμενος της Επιτροπής σας, και μάλιστα κάτω από τη δική σας προεδρία κύριε Αλμπερτίνη. Αυτό μου θυμίζει την παλιά φιλία η οποία μας συνδέει εδώ και δέκα τουλάχιστον χρόνια. Δεν θα μιλήσω Ιταλικά, θα μιλήσω Αγγλικά για να μην χρειαστεί να προσφύγετε, λέει ο κύριος Πάντουας Σκιώπας στην Διευμηνία. Όπως γνωρίζετε, το Νότρο Ευρώπη είναι παιδί θα έλεγα του Ζακ Ντελόρ. Το δημιούργησε όταν επέστρεψε στη Γαλλία δέκα χρόνια μετά από την παρουσία του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είμαι εδώ και αρκετά χρόνια πρόεδρος της Νότρο Ευρώπη και πρόεδρος της Επιτροπής Προσανατολισμού που αποτελείται από προσωπικότητες υψηλού επίπεδου στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή από πολλές χώρες. Εδώ και ένα χρόνο, όταν ξεκίνησε η Προεδρία Ομπάμα και όταν τα ευρωπαϊκά όργανα έμπαιναν σε μια διαδικασία ανανέωσης λόγω των νέων εκλογών του Κοινοβουλίου, της επιλογής των μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της πιθανότητας επικύρωσης της συνθήκης. Εμείς στην οργάνωση Νότρο Ευρώπη θεωρήσαμε ότι είχε φτάσει πλέον η στιγμή να προσπαθήσουμε να επανεξετάσουμε σε βάθος τις σχέσεις ανάμεσα στις Ηνωμένε Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργήθηκε μια ομάδα εργασίας την οποία συμπροέδρευε ο Γκίφερ Χόστατ και ο Ρωμάνο Πρόντι. Έπαιρνε μέρος και ο Γέρζι Μπούζεκ, ο οποίος μόλις είχε ενταχθεί στην ομάδα Νοτρερόπ, ο Νταβινιόν, ο Φίσερ, ο Λίπομεν και η συγγήτρια ήταν η Νικόλ Νιεζότο. Η οικογένεια λοιπόν η ευρύτερη της Νότου Ευρώπου προχώρησε στην σύνταξη μιας εκθέσεως για το νέο τρόπο αντιμετώπισης των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης και ήπα στην περίοδο την οποία έχουμε μπροστά μας. Η ομάδα συνειδητοποιούσε το ότι μετά από πολλές δεκαετίες κατά τη διάρκεια των οποίων ο κόσμος λειτουργήσε σε διπολική βάση, και η σχέση Ευρώπης-ΗΠΑ βασιζόταν σε μια συγκεκριμένη πολιτική συμμαχία, έπρεπε να υπάρξουν κάποιες αλλαγές γιατί άλλαξε η συγκυρία, άλλαξε το περιβάλλον, περάσαμε σε έναν κόσμο ο οποίος ουσιαστικά θα έλεγε κανείς ήταν μονοπολικός με την ισχύ των Ηνωμένων Πολιτειών ιδιαίτερα έντονη και με μια αντίληψη που έβλεπε ότι η στάση των Αμερικανών απέναντι στον κόσμο ήταν ε, ηγεμονικού τύπου. Η τρίτη φάση είναι ότι τελικά έχουμε περάσει σε μια πολύ πολική κατάσταση στον κόσμο σήμερα και γι' αυτό οι σχέσεις μας θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από την εταιρική, το εταιρικό τους χαρακτηριστικό. Και αυτό υπογραμμίζεται από τις προκλήσεις τις οποίες δημιουργεί η παγκοσμιοποίηση και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και προς τη ΣΥΠΑ υπάρχουν προβλήματα που προέρχονται από την παγκοσμιοποίηση. Έτσι λοιπόν αυτοί οι δύο μεγάλοι πρωταγωνιστές στη διεθνή σκηνή, η Ένωση από τη μία και η ΕΠΑ από την άλλη, δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν κάποιες από αυτές τις προκλήσεις μόνες τους. Και η ανάγκη διαχείρισης της παγκοσμιοποίησης είναι κατεπίγουσα για να αποφύγουμε οι διεθνείς σχέσεις να ακολουθήσουν θα έλεγα ένα παιχνίδι εξουσίας το οποίο μακροπρόθεσμα μπορεί να αποβεί καταστροφικό για τον κόσμο. Η έκθεση περιλαμβάνει μια ανάλυση των προκλήσεων αυτών σε διάφορους τόμεις, περιλαμβάνει μια ανάλυση των αποτελεσμάτων τα οποία δεν θα μπορέσουν να αποφύγουν από μόνες τους η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ΕΠΑ και προτείνει μια κοινή αντίληψη η οποία να εδράζεται στην αποδοχή δύο βασικών έννοιων. Η μία είναι οι πολυμερείς σχέσεις, το πολυμερές χαρακτηριστικό στις διεθνείς, στη διεθνή σκηνή, μία δηλαδή μορφή κατανομής κυριαρχίας θα έλεγα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της α, παγκοσμιοποίησης. Δεν θα σας κουράσω άλλο. Ο Στίβη που κάθεται εδώ αριστερά θα συνεχίσει και εννοεί τον υποκόμη Τιέν Ταβινιό. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα συζητήσουμε αυτά εκ νέου. Το γεγονός ότι εσείς ε, ε, μας ακούτε εδώ σήμερα δείχνει το βάρος που δίνετε στην προσπάθειά μας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Σας είμαστε υπόχρεοι. Ο Νταβινιόν έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ γιατί μας δίνετε την ευκαιρία να μιλήσουμε ενώπιον της Επιτροπής της οποίας προεδρεύεται για το έγγραφο το οποίο καταρτήσαμε από κοινού. Θα επανέλθω πολύ σύντομα στο σημείο εκκίνησης. Πριν από ένα χρόνο περίπου θέσαμε το ερώτημα σχετικά με την προβληματική των σχέσεων είπα, που έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλών συζητήσεων, προβληματισμών και εγγράφων. Θέσαμε λοιπόν και εμείς αυτόν τον προβληματισμό και σκεφτήκαμε ότι θα έπρεπε να ξεκινήσουμε από το μηδέν, σαν να μην υπήρξαν αυτά τα 60 χρόνια σχέσεων ανάμεσα στα δύο μέρη. Ακριβώς γιατί τώρα βρισκόμαστε δεν βρισκόμαστε πλέον στον κόσμο που ε, φεύγει από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο βρισκόμαστε σε έναν κόσμο που έχει εξαφανιστεί ε, η Σοβιετική Ένωση και ε, όπου η παγκοσμιοποίηση έχει γίνει καθημερινή πρακτική. Άρα λοιπόν θεωρήσαμε ότι θα έπρεπε να θέσουμε το ερώτημα τη στιγμή που η συνθήκη της Λισαβόνας προέβλεπε συμπληρωματικά μέσα, μέτρα, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τη μια και από την άλλη ε, αναλάμβανε την εξουσία στις Ηνωμένε Πολιτείε ο Ομπάμα με διαφορετική εντολή από τον προκατόχων του. Άρα λοιπόν άξιζε τον κόπο να ξεκινήσουμε ε, ε, από το μηδέν και να δούμε ε, τι συμφέρον τι και ενδιαφέρον, τι συμφέρον για μας και τι ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάπτυξη σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα, πρώτη διαπίστωση, η αλλαγή σε παγκόσμιο επίπεδο, η παγκοσμιοποίηση, άλλη εξάρτηση, η βούληση μεγάλου ε, ε, αριθμού συμπληρωματικών εταίρων που ε, ως, να συμμετάσχουν στην παγκόσμια οργάνωση, στην οργάνωση του κόσμου το τέλος του 20ου και στις αρχές του 21ου αιώνα. Άρα, πολύ σύντομα να σας πω ότι προβήκαμε στην ανάλυση αυτών των αλλαγών που σας ανέφερα και αυτές οι αλλαγές όσον αφορά τα δύο μέρη που θέλουμε να μελετήσουμε, δηλαδή τις Ηνωμένε Πολιτείε, σίγουρα την πιο μεγάλη υπερδύναμη που υπήρξε ποτέ στην ιστορία και το γεγονός ότι δεν μπορεί όμως από μόνη της να, ε, ε, να πετύχει τους στόχους που θέτει. Είτε καλή είτε κακή είναι αυτή η στόχη. Η εμπειρία στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν, ε, στο Μεσανατολικό είναι λίγα από τα άπειρα παραδείγματα που θα μπορούσαμε να δώσουμε όσον αφορά την εφαρμογή και την εκτέλεση μιας ηγεμονικής πολιτικής που δεν, μπορεί να την εφαρμόσουν, που δεν μπορεί να την εφαρμόσουν από μόνες τους οι Ηνωμένες Πολιτείες. Από την άλλη θεωρήσαμε σκοπό να σταθούμε κριτικά σε αυτό σε αυτό το οποίο αποτέλεσε ε, μία σειρά επιτευμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα επιτεύγματα αυτά είναι πολύ σημαντικά βεβαίως, αλλά ταυτόχρονα οδήγησαν σε μία κατάσταση όπου όπου ε, ε, υστερούμε πολύ σε επίπεδο αποτελεσματικότητας της πολιτικής μας και ε, ενώ επιθυμούμε να κάνουμε μία σειρά από πράγματα, δεν έχουμε τα μέσα για να τα υλοποιήσουμε. Άρα λοιπόν είναι εξίσου σημαντικό να αντιληφθούμε ότι υπήρχαν και υπάρχουν ορισμένες αυταπάτες όσον αφορά τις δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά λοιπόν αυτή τη διπλή διαπίστωση, Δηλαδή ότι οι Αμερικανοί δεν μπορούν από μόνοι τους να πετύχουν τους στόχους τους και ότι εάν δεν προσέξουν οι Ευρωπαίοι θα βρεθούν στο περιθώριο της αρχιτεκτονικής αυτού του νέου κόσμου. Πρέπει λοιπόν να θέσουμε σημαντικές ερωτήσεις και να δούμε το πώς μπορούμε να ε, αντιμετωπίσουμε τα νέα διακυβεύματα. Τρεις διαπιστώσεις λοιπόν κάναμε ως προς την κατεύθυνση αυτή. Πρώτον, ότι παντού υπάρχει κίνδυνος. Το να θεωρούμε λοιπόν ότι βρισκόμαστε σε ένα σταθεροποιημένο κόσμο είναι απολύτως λάθος. Όπου και να στρέψουμε το, το βλέμμα μας θα δούμε ότι υπάρχει πρόβλημα ή κίνδυνος, ότι η οικονομική κατάσταση είναι αυτή που όλοι γνωρίζουμε. Άρα λοιπόν και εδώ ε, ε, απαιτούνται κανόνες ε, και, και διακυβέρνηση και ότι υπάρχει ένας άλλος κίνδυνος που αφορά τη μεθοδολογία που πρέπει να ακολουθηθεί για να απαντήσουμε σε αυτές τις σημαντικές προκλήσεις που θα είναι η επιστροφή ε, σε μια πολιτική ισορροπίας δυνάμεων. Όμως εμείς στην Ευρώπη έχουμε μάθει από την ίδια μας την ιστορία ότι η σταθερότητα δεν προέρχεται από την, ε, από την ισορροπία των δυνάμεων. Άρα λοιπόν, πέραν αυτών των προβλημάτων των αντικειμενικών, υπήρχε και ένα πρόβλημα μεθοδολογίας, το οποίο είναι εξίσου σημαντικό. Επομένως θεωρήσαμε ότι εάν ακολουθήσουμε τις, τις σκέψεις αυτές που αναφέρονται στο έγγραφο, δηλαδή ότι είναι πολυμερείς οι απαντήσεις και ότι μέσα σε αυτές τις πολυμερείς απαντήσεις η Ευρώπη και η ΕΠΑ που από κοινού είναι πολύ σημαντικές οικονομικές δυνάμεις ε, και κατέχουν σημαντικές τεχνολογικές γνώσεις, δεν μπορούμε παρά να ε, ασκήσουμε επιρροή σε αυτή την έρθει Άρα λοιπόν πρέπει να θέσουμε τα ερωτήματα αυτά και αν επιθυμούμε μία πολυμερή δομή, τότε πρέπει να δούμε ποια ερωτήματα πρέπει να αντιμετωπίσει αυτή η νέα δομή και ποιες είναι οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες όλα αυτά μπορούν να επιτευχθούν με το βέλτιστο τρόπο, δυνατό τρόπο. Πολύ σύντομα θα σας πω ότι τα βασικά προβλήματα που φαίνονται έχουν να κάνουν με τη δημοκρατία και την ανάπτυξη, συνδέονται με το πρόβλημα των αξιών γύρω από τις οποίες οικοδομείται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης η κρίση στην διεθνή ασφάλεια, ε, αραβο-ισραηλινή διένεξη, προβλήματα της Ασιατικής Υπήρου, η ο προσδιορισμός σε πολιτική έναντι της Ρωσίας και βεβαίως στη συνέχεια έχουμε τις βασικές προκλήσεις του μέλλοντος, η, η κλιματολογική πρόκληση και βέβαια η κλιματική πρόκληση επιβεβαίωσε αυτό το οποίο η παραδοσιακή προσέγγιση που όπου οι Ευρωπαίοι είχαν μια κανονιστική πολυμερή ε, αντιμετώπιση στην Κοπενχάγη. Αυτή λοιπόν η προσέγγιση ε, απορρίφθηκε από μια σειρά από χώρε που θεωρούσαν ότι δεν έχουν την υποχρέωση να ακολουθήσουν τις, ε, ε τις αντιλήψεις ή τις θεωρίες ή τα διδάγματα τα οποία προέρχονταν από τη Δύση. Φάνηκε με ιδιαίτερα προφανή τρόπο ότι οι Αμερικανοί από μόνοι του δεν μπορούν να τα πετύχουν όλα αυτά, ότι συνειδητοποιούμε ταυτόχρονα και εμείς ότι και οι Ευρωπαίοι από μόνοι τους δεν μπορούν να τα πετύχουν όλα αυτά. Άρα λοιπόν, εάν οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτά τα βασικά ζητήματα και να συμβάλλουν σε μια συνένεση εκτελεστικής φύσεως επί αυτών των βασικών ζητημάτων, τα οποία ξεκινούν από την οικονομική διακυβέρνηση και φτάνουν μέχρι την ασφάλεια μέχρι την εξασφάλιση ε, της ασφάλειας, την εγγύηση ασφάλειας, λοιπόν πρέπει να ρωτηθούμε κατά πόσο στα σημερινά πλαίσια αυτές οι προνομιούχο σχέσεις ανάμεσα στους Ευρωπαίους και στους ε, Αμερικανούς ε, είναι δυνατόν να επιτευθούν. Και προσδιορίσαμε ότι μπορούν να επιτευθούν μόνο αν πληρούνται τρεις προϋποθέσεις. Και εδώ, αν θέλετε, ε, ε, παίρνουμε τις αποστάσεις μας σαν μια απλή, απλή συνέχεια ε, των σχέσεων ΗΠΑ και Ευρώπης σαν να βρισκόμαστε στην προηγούμενη κατάσταση. Καταλήγουμε στο συμπέρασμα λοιπόν ότι είναι απαραίτητη αυτή η σχέση αλλά μέσα σε διαφορετικά πλαίσια. Όλα αυτά λοιπόν μας οδηγούν στο να ορίσουμε αυτές τις τρεις προϋποθέσεις. η στρατιωτική εξάρτηση της Ευρώπης από τη ΣΥΠΑ δεν ε, συνεπάγεται απαραίτητα και οικονομική εξάρτηση. Ναι, άλλο πράγμα είναι η ασφάλεια, αλλά η εξάρτηση σε επίπεδο ασφάλειας δεν συνεπάγεται υποχρεωτικά και εξάρτηση σε πολιτικό επίπεδο. Επομένως, αυτό τι σημαίνει ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε δέχονται την ίδια ευθύνη της Ευρώπης και η Ευρώπη φιλοδοξεί να αναλάβει αυτή αυτέ τις δικές ευθύνες. Αυτή είναι η πρώτη προϋπόθεση. Δεύτερον, δεχόμαστε ότι στα πλαίσια του προσδιορισμού αυτών των νέων πολιτικών θα πρέπει να αντλήσουμε τα διδάγματα που είναι ότι τα κράτη της Ευρώπης από μόνα τους δεν μπορούν να τα πετύχουν όλα αυτά και οπομένως εάν επιθυμούμε να έχουμε ε, αποτελεσματικές πολιτικές, η έννοια ε, του επιμερισμού της κυριαρχίας ε, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και, να, και αποτελεί μάλιστα απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία και τον προσδιορισμό μιας πολιτικής. Αφήνοντας στην αρχή τα ερωτήματα γιατί δεν, πήγε, γιατί δεν θα πάει στη Μαδρίτη ο Ομπάμα, μία από τις ερμηνείες είναι ότι εάν πάει στη Μαδρίτη ο Ομπάμα δεν θα ακούσει τίποτα ενδιαφέρον ε, για αυτόν εκ μέρου των Ευρωπαίων. Δεν λέω ότι αυτή είναι η δική μου ερμηνεία, αλλά πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι τέτοιε καταστάσει δεν, θα ξανα, ε, ε, δεν, θα, ξαναεμφανιστούν ποτέ. Και τρίτη προπόθεση, οι Αμερικανοί να δεχθούν ότι η πολυμερή οδό και μια διακυβέρνηση στην οποία συμμετέχουν πολλοί εταίροι δεν είναι ε, υποχώρηση εκ μέρους τους, αλλά η αποδοχή του ότι η ηγεμονία δεν είναι μια πολιτική που θα πρέπει να ακολουθείτε. Αντίθετα, πρέπει να ακολουθούν μια πολιτική ε, ε και συνεργασίας. Αυτά λοιπόν αναφέρομαι σε αυτή την έκθεση που αφορούν τη μεθοδολογία, την επαλήθευση ε, και, ε, τα, ε, και, και τους οποίους εφαρμοστεί αυτή η πολιτική για σχέσεις προνομιούχες μεν αλλά υπό προϋποθέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τους εξέχοντες ομιλητές και αρχίζουμε τη συζήτηση. Πρώτα απ' όλα να δώσουμε το λόγο στην συνάδελφο Σάρα Λάτφορντ, αντιπρόεδρο της, ε, Επιτροπή, της Αντιπροσωπείας των Σχέσεων με τις Ηνωμένε Πολιτείε και τον, ε, και, ε, τον κύριο Μπρόκο, και ο κύριος Μπρόκ ζητά συγγνώμη για την απουσία του. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ναι, όντως αναπληρώνω και εγώ τον Έλμαρ Μπρόκ, τον πρόεδρο της αντιπροσωπείας με τη ΣΥΠΑ, ο οποίος δυστυχώς είχε ανηλυμένες υποχρεώσεις στο Συμβούλιο αλλά θα ήθελα να πω πως ε, καλωσορίζουμε αυτή την ενδιαφέρουσα έκθεση. Δεν ε, μπόρεσα να τη διαβάσω βεβαίως ε, ολόκληρη, αλλά συμφωνώ με το γενικό πνεύμα. Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, πως θα πρέπει να έχουμε εταιρική σχέση και να μην εξαρτώμεθα από τις ΗΠΑ. Και βεβαίως ε, μια διχασμένη Ευρώπη δεν έχει λόγο. Μόνο αν έχουμε μία φωνή θα ακουστούμε στην παγκόσμια σκηνή. Αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι για το, το τελευταίο κομμάτι πριν τα συμπεράσματα. Μία κάπως έτσι ενδιαφέρουσα πρόταση. Η ευρωαμερικανική εταιρική σχέση θα παραμείνει αναποτελεσματική εάν θεωρείται μόνο μία νέα δικαιολογία ή αφετηρία για κυριαρχία από τη Δύση και εννοούμε εδώ τις είπα. Μήπως ε, έχουμε εδώ πέρα έτσι, κάποια παράνοια. Δηλαδή υπάρχει ένας δισταγμός ε, για το ότι η Ευρώπη είναι ισχυρή και ενωμένη και φοβόμαστε το να έχουμε μια εταιρική σχέση ίσον διατλαντική, μήπως ενισχύσουμε την αμερικανική ηγεμονία. Δηλαδή σαν να διστάζει η Ευρώπη για το ότι είναι αξιόπιστος ε, και αποτελεσματικός σύμμαχος. Και αν είμαστε έτσι διχασμένοι, τόσο το καλύτερο. Γιατί θα αποφύγουμε έτσι το να βασίζονται πάνω μας οι Αμερικάνοι ως ε, εφαλτήριο ως εφαλτήριο για την παγκόσμια κυριαρχία τους. Πράγματι υπάρχουν κάποια τέτοια στοιχεία, δηλαδή όσο πιο ενωμένοι και αποτελεσματικοί είμαστε, τόσο πιο μεγάλος ο κίνδυνος να μας έχουν δεδομένους οι Αμερικάνοι και να πατήσουν πάνω μας και να κυριαρχήσουν στον κόσμο. Ευχαριστώ κυρία Λότφορντ. Αρχίζουμε λοιπόν με την συζήτηση. Έχουμε 8 ομιλητέ και για να ε, τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα σας παρακαλώ να αναπτύξετε τις απόψεις σας και να διατυπώσετε τις ερωτήσεις σας σε 1,5 λεπτό. Πρώτος ομιλητής. Φρανσίσκο Μίλα Φρανσίσκο Μιλανμόν, που ήταν ε, εισηγητή τη Επιτροπή μα για τι διατλαντικέ σχέσει. Έχετε το λόγο για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Ε, κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι ιδιαίτερα που σα ξαναβλέπω σήμερα το απόγευμα. Είχα την ευκαιρία να είμαι στην παρουσίαση τη έκθεσή σα σήμερα το πρωί, όταν σα συνόδευε και ο, ο πρόεδρο Μπούσεκ. Πριν από ένα χρόνο είχαμε μία έκθεση που ενεκρίθηκε, ενεκρίθηκε στο τέλο ε, Μαρτίου του 2009, όπου αναφέραμε ότι ε, είναι πλέον στρατηγική σημασία και ε, οι ε, σχέσει μας με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Πιστεύω, όπω και εσείς, ότι οι σχέσεις αυτές πρέπει να εξεταστούν με προσοχή. Και φαίνεται όμως ότι τα τελευταία δύο χρόνια φάνηκαν τρεις παράγοντες, θα έλεγα, που διευκολύνουν την ενίσχυση αυτών των σχέσεων τη σύσφυξη των σχέσεων. Από τη μια έχουμε τη νέα ε, κυβέρνηση στι ΗΠΑ, ε, τον πρόεδρο Ομπάμα, ε, που είναι πιο ανοιχτό στον πολυμερή χαρακτήρα. Δεύτερον, έχουμε μια νέα Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θέλετε, με τη συνθήκη τη Λισαβόνα, ενισχυμένη, με νέου θεσμού με νέα όργανα. Και τρίτον, νομίζω ότι έχουν συνειδητοποιήσει και τα δύο μέρη ότι, βρισκόμα, ότι σήμερα βρισκόμαστε σε ένα νέο σενάριο, όπω είπατε κι εσεί. Η προκλήση δεν είναι μόνο θεωρητική φύσεω και δεν ε, είναι χρήσιμε μόνο οι στρατιωτικέ συμμαχίε όπω το ΝΑΤΟ, αλλά απαιτούνται παγκόσμιε εταιρικέ σχέσει ανάμεσα σε δύο εταίρου όπω ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένε Πολιτείε. Βεβαίω η σύσφυξη των σχέσεων αυτών περνά όχι μόνο από την πολιτική βούληση των κρατών, αλλά νομίζω ότι αυτό που απαιτείται ναι, βεβαίω από, τα, από τα κράτη, αλλά αφήστε με να σταθώ για λίγο στο ότι εμεί και οι 27 συνειδητοποιούμε ότι μιλώντα με μία φωνή θα είμαστε πιο αποτελεσματικοί στη σχέση μα με, την Ευρωπα... με τι Ηνωμένε Πολιτείε. Πρέπει το συνειδητοποιήσουμε αυτό, παρά να ακολουθούμε μια πολιτική διμερών σχέσεων. Για να ενισχύσουμε λοιπόν αυτέ τι σχέσει, χρειαζόμαστε και τα νέα μέσα τη συνθήκη Λισαβόνα. Σήμερα το πρωί είχα την ευκαιρία να αναφερθώ στο ζήτημα αυτό στην ΥΠΟΤΕΚ εκπρόσωπο. Ένα, ε, έχουμε το μόνιμο πρόεδρο ε, και θα ήθελα να σα ε, σας ρωτήσω. Όσον αφορά τα νέα όργανα από τη Λισαβόνα, δεν πρέπει να έχουμε αρνητική ε, στάση απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κρίση, ε, προβλήματα. αυτά βλέπω στη σελίδα 11 όσον αφορά τη φωτογραφική απεικόνηση αυτή τη στιγμή τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να μου σχολιάσετε αυτό το ζήτημα και αυτέ τι ακραίε θέσει κατά κάποιο τρόπο. Ευχαριστώ. Γκόμε για 1,5 λεπτό. Σα παρακαλώ, 1,5 λεπτό. Thank you for your, um, views. Ευχαριστώ για τι ε, απόψει σα πράγματι πολύ ενδιαφέρουσες. Συμφωνώ με το δεύτερο συμπέρασμά σας πως τα κράτη-μέλη δεν αρκούν, οπότε δεν φτάνει μόνο η διακυβερνητική προσέγγιση και πράγματι έτσι υποβαθμίζεται η δυνατότητα δράσης για να σώσουμε π.χ. την Ελλάδα τώρα ή για να μην αναφέρω και άλλα ζητήματα σοβαρά όπως π.χ το να αντιπαλέψουμε αυτές τις μαύρες τρύπες εγκληματικότητας που είναι οι υπεράκτιες εταιρείε. Συμφωνώ πως ε, πρέπει, είπα, να αποδεχτούν ε, έναν πολύπλευρο κόσμο, αλλά το ίδιο πρέπει να κάνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αντί να πηγαίνουμε προς τους G2, να ενισχύσουμε τον ΟΗΕ και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει κάνει τίποτα στη συνθήκη της Λισαβόνας για να υπάρξει μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ εάν είναι να έχουμε πράγματι αποτελεσματική πολυμερή πολιτική. Και πράγματι αναφέρομαι στο πρώτο σας συμπέρασμα. Η πολιτική ανεξαρτησία δεν σημαίνει στρατιωτική ανεξαρτησία. Εγώ από αυτά που βλέπω στο σημερινό κόσμο νομίζω πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να απέχει από την οικοδόμηση στρατιωτικής ισχύω. Όχι για λάθος σκοπούς, για τους σωστούς σκοπούς, για να υπάρχει σωστή πολυμερής ε, εφαρμογή του δικαίου στο διεθνές επίπεδο. Ευχαριστώ κυρία Γκόμες. Η κυρία Νέιτς, 1,5 λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους ε, της ε, Νότρε Ροπ ε, για την συνεισφορά τους στην αναδιαμόρφωση των σχέσεών μας με τις ΗΠΑ. Είναι βεβαίως η στιγμή περίεργη. Είμαστε ακόμα σε μια μεταβατική φάση όσον αφορά τα θεσμικά όργανα. Θα έχουμε υπηρεσία εξωτερικής δράσης, αλλά ακόμα δεν υπάρχει και ταυτόχρονα ο κόσμος δεν έχει σταματήσει να γυρίζει και δεν μας περιμένει. Δεν περιμένει ο κόσμος να ξεμπλέξουμε εμείς και να κάνουμε είσοδο. Όπως και να έχουν τα πράγματα πρέπει να εκμεταλλευτούμε την κατάσταση. Και να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Θεωρώ πως πρέπει να δούμε τον εαυτό μας έτσι με λίγο μια κριτική ματιά. Πρώτα απ' όλα εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση χρειαζόμαστε έτσι μια παλιά καλή εξωτερική πολιτική που θα αρχίσουμε να ζητούμε λύσεις και όχι να κάνουμε δηλώσεις. Καλά τα πάμε στα λόγια, αλλά όχι τόσο καλά στο να λύνουμε προβλήματα. Οπότε αυτό χρειαζόμαστε. Δεύτερον, όταν ε, προετοιμαζόμαστε για πολυμερείς διαπραγματεύσεις πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πως δεν φτάνει να συμφωνήσουμε εμείς εδώ μεταξύ μας και να πάμε στη διάσκεψη π.χ. στη Κοπεχάγη και να θεωρήσουμε ότι όλοι μας ακολουθούν, γιατί συμφωνήσαμε μεταξύ μας μόνο. Αυτό το οποίο συνέβη στην Κοπεχάγη υπογράμμισε την δυσκολία των διαπραγματεύσεων που έρχονται. Ευχαριστώ και την υπομονή σας. Ευχαριστώ, κυρία Λόιζινγκ. Καταρχήν εγώ δεν έλαβα καν την έκθεση γραπτό. Κάποιοι άλλοι την έχουν, τη διαβάζουν από μέσα. Α, είναι απ' έξω εδώ, εντάξει, ευχαριστώ. Μετά, λέτε για αυτή την διάσταση πολιτικής και στρατιωτικής ανεξαρτησίας να σας υπενθυμίσω πως η πολιτική ανεξαρτησία σχετίζεται με τη νέα στρατηγική του ΝΑΤΟ. Και αναρωτιέμαι πώς θα έχουμε πολιτική ανεξαρτησία εντός ε, του ΝΑΤΟ όταν έχουμε στρατιωτική ε, εξάρτηση και με αυτή την αρχή της ε, συνένεσης εντός του ΝΑΤΟ. Ένα άλλο ερώτημα. Ο αντιπρόεδρος ε, των ΗΠΑ, ο Τζοζεφ Βάιντεν, ξεκαθάρισε πως η Ουάσιγκτον είναι διατεθειμένη να κάνει περισσότερα πράγματα διεθνώς, αλλά να σκεφτούν και οι σύμμαχοι της υποχρεώσεις τους και μιλάει εδώ πέρα βεβαίω και για στρατιωτική ισχύ. Μήπως αυτό είναι ένα deal δηλαδή να δώσει κάποια εξουσία η ΕΠΑ εάν ε, συμμετέχει περισσότερο στρατιωτικά ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε δηλαδή μια στρατιωτικοποίηση της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μας λένε η ΕΠΑ ότι επενδύουμε πολύ λίγο στην άμυνα. Συχνά αναφέρεται ως μήνυμου με ένα 2% του ΑΕΠ. πού βλέπετε εσείς ε, τη διαφορά και το όριο και όλες για να έχουμε και μια καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και τη στόχια στην Ευρώπη. Τελευταία ερώτηση. Πριν περάσουμε στον πρόεδρο Πάντουα Σκιώπα, ο κύριος Μπούτι Κόφερ, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Οι Αμερικάνοι έχουν τον πρώτο ειρηνόφιλο πρόεδρο που ξεκαθαρίζει ένα πράγμα ό,τι και αν κάνει. Δεν βλέπει νοσταλγικά τη σχέση του μαζί μας, αλλά ρεαλιστικά. Εγώ αμφιβάλλω πως οι Ευρωπαίοι με τη νοσταλγική τους στάση μπορούν να επηρεάσουν την Αμερικανική πολιτική ή τον κίνδυνο της περιθωριοποίησής μας. Υπάρχει μια διαλεκτική στην ε, διατλαντική σχέση. Θα αποκτήσει σημασία και θα κερδίσει σημασία και οι δύο πλευρές αποκτήσουν την πρακτική εμπειρία πως είναι αμοιβαία χρήσιμη ο ένας τον άλλον. Γιατί το είπε και μία συνάδελφος εδώ πέρα ότι οι Αμερικάνοι αμφιβάνουν γι' αυτό. Λένε όλο δηλώσεις κάνετε και στην πράξη τίποτα. Δεν συνεισφέρεται σε τίποτα και κάτι το οποίο δεν κατάλαβα εδώ πέρα σε δύο σημείο. Πιθανώς πρέπει πράγματι να έχουμε την ανησυχία πως ε, εάν συνεργαζόμαστε καλύτερα θα επιβάλλουν την ατζέντα τους Είπαμε πως έχει περάσει πια ο καιρός της μονομέρειας και μετά λέτε η Δύση δεν θα αναλάβει την ηγεσία. Το ερώτημα είναι απλό. Πρώτον, πρέπει να υπάρχει ηγεσία. Και δεύτερον, εάν ναι, ποιος θα την ασκήσει. Θα δώσω το λόγο τώρα στον πρόεδρο Παντό Θα πρέπει να φύγει πριν από τον Etienne Νταβινιόν από τη συνεδρίασή μας. Θα αναφερθώ... αναφερθώ σε κάποια από τα σχόλια και ο Ετιέν θα απαντήσει στα υπόλοιπα. Ένα από τα θέματα που τέθηκαν περιλαμβάνεται στην ανάλυση της έκθεσης σχετικά με την αυξανόμενη ακαταλληλότητα και την αυξανόμενη ανεπάρκεια των δράσεων που βασίζονται αποκλειστικά στην έννοια θα έλεγα που έχουμε για το ε, κράτος έθνος. Η παγκοσμιοποίηση δημιουργεί ένα παράδοξο. Από τη μία υπονομεύει την εξουσία που έχουν τα κράτη μεμονωμένα να αντιμετωπίσουν και τη δύναμη που έχουν σε μεμονωμένο επίπεδο να δώσουν απαντήσεις και από την άλλη αυξάνει κάποια θα έλεγα αισθήματα και κάποιες ανησυχίες για την προάσπιση της ακαιρεότητας και της κυριαρχίας των χωρών. Βλέπουμε το τι δείχνει η εμπειρία της τελευταίας δεκαετίας βλέπουμε ποια ήταν η πορεία της πιο ισχυρής και ταυτόχρονα της πιο πλούσιας χώρας στον κόσμο και αναφέρομαι φυσικά στη ΣΥΠΑ και γι' αυτό ακριβώς προσπαθούμε να βρούμε κάποια νέα στοιχεία στις ε, σχέσεις αυτές. Να έρθω στην παρατήρηση την οποία έκανε η κυρία Γκόμες για την ακαταλληλότητα την οποία επιδεικνύει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια της προώθησης της μεταρρύθμισης του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Και ταυτόχρονα της προσπάθειας αποφυγής από πλευράς των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων Τη ευθύνη την οποία έχουν να αναλάβουν μόνοι τους υπεύθυνα την υπεράσπισή τους ή την άμυνά τους. Νομίζω ότι αυτά τα δύο στοιχεία είναι καθοριστικά η Ευρώπη. Θα πρέπει να προσπαθήσει να καλύψει κάποιες παραλήψεις οι οποίες χαρακτηρίζουν τις πολιτικές της, αλλά και οι Ηνωμένε Πολιτείες από την αντίθετη αν θέλετε κατεύθυνση θα πρέπει να αναθεωρήσει το όνειρο της αυτάρκειας και της πλήρους ανεξαρτησίας. Αν θέλετε εδώ έχουμε να κάνουμε με δύο αντιλήψεις καθρέφτη, με δύο αντιλήψεις παραπληρωματικές, οι οποίες θα πρέπει να διορθωθούν. Συμφωνώ λοιπόν με τις παρατηρήσεις της κυρίας Γκόμες. Δεν θα σας κουράσω εγώ άλλο. Ευχαριστώ κύριε Πάντο Ασκιώπα. Μετά από την συμπλήρωση όλων των ερωτήσεων θα δώσω το λόγο στον δόκτωρα Νταβινιό. Αλλά δεν θα πρέπει όσοι είναι εγγεγραμμένοι να ξεπερνούν το ένα λεπτό. Ο κύριος Κέλαμ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και αναφέρομαι στους δύο ομιλητές να εκφράσω το θαυμασμό μου για την προσπάθεια την οποία έκανα να αντιμετωπίσουν αυτές τις δύο δύσκολες, ε, αυτά τα δύσκολα θέματα. Δείχνεται το πώς μπορούμε να, να αυτά τα μειονεκτήματα τα οποία μας χαρακτηρίζουν σήμερα να τα μετατρέψουμε σε πλεονεκτήματα σχετικά. Ίσως η μία γνώση της υπερεθνικής εικόνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία κάποτε ήταν χρήσιμη στο παρελθόν, ίσως θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί εκ νέου στα πλαίσια της αντιμετώπισης των συνεπειών της παγκοσμιοποίησης. Πάντως Κάποιοι υποστηρίζουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένε Πολιτείε μοιάζουν σαν ένα κουρασμένο, γερασμένο και γρουσούζικο ζευγάρι. Είναι έτσι τα πράγματα. Θα συμφωνήσετε με αυτά τα οποία είπε ο Αλεξάνδερ Στούμπο, Υπουργός Εξωτερικών της Φιλανδίας ότι θα πρέπει να υπάρξει μια νέα πράξη αλληλεγγύης ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένε Πολιτείε. και ότι θα πρέπει επίσης να προωθήσουμε ακόμα περισσότερο όπως έχει ζητήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ιδέα της υπερατλαντικής αγοράς. Τάλερ, ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και τους ε, δύο προσκεκλημένους μας για την έκθεση αυτή. Νομίζω ότι η έκθεση αυτή ήρθε την κατάλληλη στη χρονική στιγμή. Η πράγματι είναι μια σημαντική χώρα. Άρα αν λάβουμε υπόψη το ΑΕΠ ε, μπορούμε να πούμε ότι η ε, Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πιο, κατά 30% μεγαλύτερη χώρα εντό εισαγωγικών. Να σα ρωτήσω το εξή Για το, για το είναι το πλέον σημαντικό παγκόσμιο πρόβλημα και εδώ η ΕΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσαν να κάνουν πολύ περισσότερο από κοινού από ό,τι έχουν κάνει μέχρι στιγμή. Ενώ πιστεύω ότι ε, το πρόβλημα αυτό ε, είναι η βασική πηγή δημιουργίας αστάθειας στο παγκόσμιο, σε παγκόσμιο επίπεδο ε, και δημιουργεί τα περισσότερα αντιευρωπαϊκά και αντιαμερικανικά αισθήματα. Ρωτώ λοιπόν, Πώς, ε, πιστεύετε ότι θα μπορέσουμε να καταφέρουμε την επίτευξη ε, μακροχρόνιας ειρήνης ε, στο Μεσανατολικό ή θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το ΝΑΤΟ. Ευχαριστώ. Βαν Μπάλεν, για να τελειώσει η συζήτηση για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Γεγονό είναι ότι αν εξετάσετε την ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική θα δείτε ότι έχουμε δύο μέλη που είναι μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας που έχουν, κατέχουν μια θέση την οποία δεν πρόκειται να, ε, την οποία δεν πρόκειται να υποχωρήσουν. Πρέπει να δούμε λοιπόν πώς οι Γάλλοι, οι Βρετανοί και η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να συνεργαστούν και πώς βλέπετε αυτό το ζήτημα. Δεύτερον, μιλήσατε για στρατιωτική ανάμειξη. Προσωπική μου άποψη είναι αν δεν μπορεί να στείλει θέματα, για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Αφγανιστάν, ποτέ δεν θα έχουμε ε, σχέση σε ισότιμο επίπεδο με τι ΗΠΑ. Πρέπει ε, να μην ασχοληθούμε μόνο με την soft power, με την ήπια εξουσία, αλλά και με το στρατιωτικό σκέλο. Ποια είναι η άποψή σα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σα παρακαλώ, κύριε Νταβινιόν, να απαντήσετε Μέχρι τις 4 και 4 πρέπει να έχουμε ολοκληρώσει τη συζήτηση. Τώρα εσείς απαντήστε ε, για όσο χρόνο έχετε στη διάθεσή σα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα είμαστε εδώ πιο σύντομος. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά αυτά τα φαλτήρια για τα οποία με ρωτήσατε, αυτό που προσπαθούμε να πούμε είναι ότι αυτή η καρικατούρα των σχέσεών μας με τη ΣΥΠΑ, εάν δεν στηρίζεται ε, σε συγκεκριμένες προσπάθειες, τότε πραγματικά θα μας βλέπουν σαν καρικατούρα. Σαν να προσπαθούμε να αυτή τη δεσπόζουσα θέση να την καλύψουμε. Αυτό είναι ο φόβος, δεν είναι στόχος. Η ολόκληρη έκθεση στηρίζεται σε αυτό το θέμα. Και τώρα όσον αφορά τις άλλες ερωτήσεις, τις συναφείς ερωτήσεις, να σας πω το εξής. Ένας ε, κόσμος πολυμερής απαιτεί συνεισφορές από τους άλλους. Και σημαίνει ότι πρέπει οι συμβολές αυτές, οι συνεισφορές αυτές να λαμβάνονται υπόψη από τους υπόλοιπους. Δεν ε, δεν υπάρχει κανένα ισχυρό που να πετύχει τη δέσμευση και των υπολείπων. Και αν μου επιτρέπετε, να ξαναγυρίσω και λίγο στην Κοπενχάγη. Η συνδιάσκεψη της Κοπενχάγης δεν θα μπορούσε να είχε γίνει χωρίς τη συμβολή και τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά πήγαμε στη διάσκεψη της Κοπενχάγης έχοντας την άποψη ότι το αποτέλεσμα θα ήταν ανάλογο με τις προηγούμενες προσπαθίες μας, δηλαδή συλλογική συμφωνία με συλλογική δέσμευση και αξιολόγηση του πώ έχουν αντιμετωπιστεί μέχρι στιγμή αυτέ οι συνολικέ υποχρεώσει. Φάνηκε όμω στην Κοπενχάγη ότι η πλειονότητα των άλλων χωρών δεν συμφωνούσαν με αυτή την προσέγγιση και ήθελαν μια διαφορετική προσέγγιση με βάση τη διαπραγμάτευση των δικών του συμφερόντων. Δεν δέχονταν λοιπόν σαν δεδομένο ότι το πολυμερές φόρουμ είναι η σωστή αντιμετώπιση. Άρα λοιπόν πρέπει να αντιληφθούμε ότι ίσως θα πρέπει να πείσουμε και τους υπολείπους να ακολουθήσουν την οδό του πολυμερούς, της πολυμερούς μεθοδολογίας. Θα πετύχουμε όμως μόνο εάν συμβάλλουν και οι υπόλοιποι στους κανόνες αυτής της πολυμερούς φιλοσοφίας και να μην κάνουμε αυτό το οποίο κάνουμε εδώ και χρόνια. Μα αυτή είναι ακριβώς η αλλαγή. Και εδώ πρέπει να προσέξουμε το συγκεκριμένο αυτό σημείο. Επομένως, ε, η βασική ε, ιδέα σε ολόκληρη την έκθεση είναι ότι κανείς σήμερα δεν μπορεί να υποστηρίζει τους άλλους τι πρέπει να κάνουν. Από την άλλη όμως, αν δεν υπάρχουν ορισμένοι κανόνες, δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα βασικά προβλήματα. Άρα θα πρέπει να δούμε ε, την πλατφόρμα και τη μεθοδολογία συζητήσεων για να μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Και στα πλαίσια αυτά η φιλοδοξία των Ευρωπαίων είναι να μην βρεθούν στο περιθώριο. Η ανάγκη των Αμερικανών είναι να αναπτύξουν όλε τι δυνατότητε και το ρόλο του και αν συμφωνήσουμε ε, οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί σε μία σειρά στόχων που θα αποτελέσουν τη δική μα συνεισφορά αλλά όχι το συμπέρασμα των διαφόρων συνδιασκέψεων, τότε αυτός είναι ένας πολύ χρήσιμος τρόπος για να προχωρήσουμε. Ναι, στενές σχέσεις με τη ΣΥΠΑ, αλλά να συμφωνήσουμε σε τι θα προσδώσουν, τι θα προσδώσουν όλες αυτές τις σχέσεις και να εγκαταλείψουμε ε, την ε, σκέψη του παρελθόντος. Και σε σχέση με αυτό, Έχουμε το ερώτημα για τη Μέση Ανατολή. Πρέπει τα δύο μέρη να κάνουν περισσότερα και καλύτερα ε, στη, στη, Μέση Ανατολή. Η απάντηση είναι σαφώς ναι. Σήμερα υπάρχει ένα είδος καταμερισμού εργασίας όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση συμβάλλει μαζικά στην ε, ε, οικονομική βοήθεια και ενίσχυση των Παλαιστινίων και εδώ δεν έχουμε κανένα πρόβλημα και η αναλαμβάνουν το καθήκον να προσπαθούν να πείσουν τους Ισραηλινούς ότι πρέπει να υπάρχει συμφωνία. Μα ε, εδώ όμως μιλάμε για δύο διαφορετικές προσπάθειες. Άρα, κανείς δεν αξιοποιεί ε, τα αποτελέσματα του άλλου μέρους και των προσπαθειών του άλλου μέρους. Και εδώ πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Και συμφωνώ επίσης σε μεγάλο βαθμό και με την εξή παρατήρηση, ότι οι συνέπειες του συνεχιζόμενου αδιεξόδου στη Μέση Ανατολή οδηγούν σε ε, ε, σημαντική μείωση της δημοτικότητας οποιοδήποτε οποιασδήποτε προσπάθειας προέρχεται από τη Δύση. Είτε δίκαια είτε άδικα. Ε, φαίνεται όμως και το ξέρουμε όλοι ότι η αντίληψη και η εικόνα που έχουν οι άλλοι είναι πιο σημαντική. Άρα και άλλοι ανησυχούν για την έλλειψη της ειρήνης, αλλά ε, δυστυχώς λόγω αυτού του καταμερισμού εργασίας έχουμε αυτή την αρνητική εικόνα. Και αυτό το σημείο λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, και το λέμε άλλωστε στην έκθεση, ότι η ρητορική μας ε, είναι εξαιρετικής ποιότητας, αλλά δεν αρκεί αυτό. Δεν μπορούμε να πείσουμε με λόγια, πρέπει να πείσουμε με πράξεις, με στόχους και αποτελέσματα. Και τώρα που έχουμε το μέσον, έχουμε τα μέσα που μας έδωσε η ίδια συνθήκη της Λισαβόνας, δεν έχουμε πλέον καμία δικαιολογία. Τώρα δεν μπορούμε να πούμε ότι θα θέλαμε να κάνουμε κάτι αλλά δεν έχουμε τα εργαλεία για να το πράξουμε. Όχι. Τώρα έχει φτάσει η στιγμή της αλήθειας. Έχουμε τα εργαλεία και τι θέλουμε να κάνουμε τώρα με τα εργαλεία αυτά. Τα εργαλεία θα είναι έγκυρα και αποτελεσματικά εάν οδηγούν σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Σε αυτή την κατάσταση βρισκόμαστε τώρα και πρέπει να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε και τι δεν θα κάνουμε. Και γι' αυτό αναπόφευκτα, αναπόφευκτα το τονίζω, η αποτελεσματικότητα σημαίνει καταμερισμό, επιμερισμό. Δεν είναι δυνατόν να ορίσουμε μία θέση που, ε, και η θέση αυτή να είναι το άφρισμα των θέσεων των 27 κρατών μελών. Αυτό δεν είναι πλέον θέση. Ε, είναι απογραφή και δεν πρόκειται να οδηγήσει σε πράξεις. Άρα λοιπόν πρέπει να αρχίσουμε να αποδεχόμαστε ότι ε, στην ε, πρώτη γραμμή των πολιτικών μας και διπλωματικών δραστηριοτήτων μας για να πετύχουμε αποτελέσματα σε, στην ευρωπαϊκή σφαίρα θα πρέπει ε, να χρησιμοποιήσουμε και μέσα από τη σφαίρα αυτή. Να είμαστε λοιπόν έτοιμοι να μοιραστούμε μέρος της εθνικής μας καριερχίας διότι οι επιμέρους δράσεις δεν αρκούν πλέον. Το θέμα δεν είναι κατά πόσον φοβόμαστε τη μονομερή δράση, αλλά τη μονομερή έλλειψη αποτελεσματικότητας. Διότι με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται μεγάλη ασάφεια και αυ... όσον αφορά τους στόχους μας. Δεν φοβάμαι ε, τη, τη G2, δεν νομίζω ότι υπάρχουν κοινά, αρκετά κοινά στοιχεία ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και στην Κίνα ώστε να οδηγηθούν σε μια μακροχρόνια σχέση, αλλά φοβάμαι ότι αν δεν, δεν εκφράσουν τι δικέ του επιθυμίε οι Ευρωπαίοι, δεν πούν τι μπορούν να δεχθούν και τι δεν μπορούν να δεχθούν και δεν είναι έτοιμοι να δεσμευθούν, τότε φοβάμαι για το αποτέλεσμα. Και τελειώνοντα, το, το συνολικό ζήτημα τη ασφάλεια, ε, των δαπανών κτλ. Εδώ να σα πω το εξή. Αυτό το οποίο προσπαθούμε να πούμε στην έκθεση και θα το διαβάσετε, ε, προσπαθώ αυτή τη στιγμή να συνοψίσω όλες αυτές τις ιδέες, είναι το εξή πάντως. Επειδή υπάρχει εξάρτηση ασφάλειας από τις Ηνωμένε Πολιτείες, αυτό δεν σημαίνει ότι αυτόματα πρέπει να δεχθούμε και πολιτική εξάρτηση από τις ΗΠΑ. Αυτό είναι μια συγκεκριμένη δήλωση. Στη συνέχεια πάμε ένα βήμα περαιτέρω. Πρέπει να δεχθούμε στρατιωτική εξάρτηση από τις Ηνωμένε Και εδώ λέμε όχι. Αλλά όταν ε, ε, καταρτίζει κανείς κάποιες εκθέσεις, ξεκινά από το που βρίσκεται και μετά ε, περιγράφει, περιγράφει την κατάσταση και λέει που θέλουμε να πάμε. Γιατί αν μιλήσουμε μόνο για τις επιθυμίες μας, τότε καταλαβαίνετε ότι θα υπάρξει μια αντίφαση σχέση με την πραγματικότητα ως τον αναγνώστη. Λέμε πώς έχουν τα πράγματα. Δεν λέμε ότι θα πρέπει να είμαστε πολιτικά εξαρτώμενοι ή εξαρτώμενοι στο θέμα της ασφάλειας. Και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος με την πάροδο του χρόνου. Δηλαδή πριν από πέντε χρόνια θα βρισκόμασταν εδώ, κανείς δεν θα, μας, δεν θα πίστευε ότι οι γερμανικές δυνάμεις θα βρίσκονται σε, σε άλλες χώρες, λαμβάνοντας υπόψη την παλιά παράδοση του ΝΑΤΟ, εκτός ε, της ε, ζώνης επιρροής ε, της Ατλαντικής Συμμαχίας στο Αφγανιστάν, δεν ξέρω, στα Βαλκάνια ίσως θα μπορούσε κανείς να το συζητήσει. Άρα έχει σημειωθεί πρόοδος. Όχι αρκετή, αλλά αρκετή αν θέλετε για να μην α, ε, δημιουργούμε ψευδεστήσεις με την έκθεσή μας. Εμείς με την έκθεσή μας αναφέρουμε τι πιστεύουμε θα μπορούσε να επιτευχθεί ε, ρεαλιστική. Δεν είναι περιγραφή του τι θα έπρεπε να γίνει σε κάθε περίπτωση, αλλά περιγραφή του γιατί. Δηλαδή, αν θέλουμε να παίξουμε ένα ρόλο στον μεταβαλλόμενο αυτό κόσμο, τότε υπάρχει η εταιρική σχέση με τη ΣΥΠΑ αλλά το βασικό, και που θα βοηθήσει, αλλά το βασικό σημείο είναι το πώς θα οργανώσουμε αυτήν την εταιρική σχέση. Αυτά τα στοιχεία προσπαθήσαμε να βάλουμε στην έκθεση αυτή και νομίζω ότι απάντησα όσο καλύτερα μπορούσα στις διάφορες ερωτήσεις και να σα πω για άλλη μια φορά ότι αισθανόμαστε μεγάλη ευγνωμοσύνη που μα δώσατε την ευκαιρία να έρθουμε εδώ και να μιλήσουμε για το κείμενό μα. Ευχαριστούμε. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συνάντηση και οι απαντήσει. η ανταπόκριση των συναδέλφων μαρτυρεί άλλωστε το ενδιαφέρον ε, όλων μας. Συνοψίζω τα τρία βασικά επιχειρήματα και αυτό που βγαίνει από την έκθεση είναι ότι η Ευρώπη ε, θα πρέπει να, ε, να δει ε, και, το, και το κατά πόσο το ΝΑΤΟ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως ένα μέσο για να υποστηρίξει τη συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης και είπα πρέπει να υπάρξει σύσφυση των σχέσεων θα πρέπει όμως να δούμε το πώς και η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα είναι ένα απλό άθροισμα των θέσεων των 27 κρατών μελών αλλά θα πρέπει να εκφράζει το σύνολο τέλειωσε η εποχή του West and West και θα πρέπει τώρα να εργαστούμε όλοι προς προ την κατεύθυνση μια πολυμερού φιλοσοφία τη διεθνή σχέση. Σα ευχαριστώ για την παρουσία σα και συνεχίζουμε τώρα τι εργασίε μα. Και πάμε αυτή εξ αρχή στι ψηφοφορίε, την ψηφοφορία μάλλον. Για την πρόταση απόφαση Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για τη μακροοικονομική βοήθεια για την Ουκρανία. Σας προτείνω να βγάλετε τα δελτία σας, αν δεν τα έχετε κάνει ήδη, βγάλετε τις κάρτες, γιατί θα αρχίσουμε την ψηφοφορία εντός ολίγου. Qualcuno l'ha dimenticata, qualche secondo di tempo per farla Κάποιος έχασε την κάρτα του, ε, ένα λεπτό. Bene, allora possiamo cominciare. Αρχίζουμε. Αιτιολογική σκέψη 1, τροπολογία 1, εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία 2. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτή. Περνάμε τώρα Θέλετε να υπάρξει ηλεκτρονικός έλεγχος. Καλώς λοιπόν. Για την τροπολογία 2 ξεκινάει η ψηφοφορία. Βλέπω ότι δεν δεχόμαστε πιστοτικές κάρτες όπως American Express λοιπά. Καλώς, 60 ψήφισαν, 38 είναι υπέρ, γίνεται δεκτή. πίπτη η 10, ψηφίζουμε την 3, ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές, δεκτή. 4, ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές, δεκτή. 5, ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή, η 6, υπέρ κατά αποχές δεκτεί. Η 7 υπέρ κατά αποχές δεκτεί. Η 8 υπέρ κατά αποχές δεκτεί. Η 11 υπέρ κατά αποχές δεκτεί. Καλώς. Πάντα με ηλεκτρονικό τρόπο. Έχουμε τώρα την τελική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Τέλος της ψηφοφορίας ψηφίζουν 61, 57 υπέρ, 4 αποχές, κανένας κατά. Συγχαρητήρια. Τελείωσε η ψηφοφορία. Συνάδελφοι, συνεχίζουμε. Ξεκινάμε τη δεύτερη συζήτηση. Τη δεύτερη συζήτηση λοιπόν της εκθέσεως Αλαφράγκα για τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις σχέσεις της με τη Λατινική Αμερική. Η πρώτη ανταλλαγή απόψεων έγινε στις 4 Φεβρουαρίου του 2010 και θα ψηφίσουμε αύριο. Χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις, γνωρίζω ότι βιάζεται και ο συνάδελφος Σαλαφράνκα, θα του δώσω αμέσως το λόγο και μετά σε όλους τους άλλους συναδέλφους που θα τον ζητήσουν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι διάβασα με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή ξαναρχίζει ο κύριος Σαλαφράγκα. Λοιπόν, μελέτησα με την μέγιστη δυνατή προσοχή τις 100 περίπου τροπολογίες οι οποίες κατατέθηκαν στην έκθεσή μου. Προσπάθησα να δω αν οι τροπολογίες αυτές ήταν συμβατές με το έγγραφο το οποίο έχω ετοιμάσει, το οποίο όπως σας είπα δεν είναι ένα κείμενο αυτόνομο, πρωτότυπο εντελώς, αλλά εμπνέεται ουσιαστικά από, τις προηγούμενες, από τα προηγούμενα ψηφίσματα που έχουν γίνει δεκτά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από τη συνάντηση κορυφής. Δέχτηκα σχεδόν όλες τις τροπολογίες της σοσιαλιστικής ομάδας. Ο κύριος Μενέντες Δεβάγε, σε ορισμένες τουλάχιστον περιπτώσεις, προσπάθησε να αναπροσανατολίσει θα έλεγα το κείμενο, αλλά παρόλα αυτά ε, προσπαθήσαμε να διατηρήσουμε τις βασικές κατευθύνσεις ε, της εκθέσεως Δέχτηκα πολλές τροπολογίες επίσης και της ομάδας των φιλελευθέρων και από τις υπόλοιπες τροπολογίες ε, δεν δέχτηκα θα έλεγα αυτές οι οποίοι θα ενίσχυαν κατά τη γνώμη μου την συγκεκριμένη έκθεση. Ίσως να επανέλθω σε αυτές τις τροπολογίες οι οποίες ήθελα να καλύψουν κάποια ε, κενά τα οποία παρουσιάζει η έκθεση Λόγω της έλλειψης χώρου όμως, ε, ε, την οποία αντιμετωπίζουμε, δεν μπορούμε να γράφουμε δεκάδες σελίδες. Υπάρχουν θέματα στα οποία θα μπορούσαμε να ε, συμφωνήσουμε στα θέματα της περιφερειακής συνεργασίας, στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι πλευρές αυτές συμπλήρωσαν την έκθεση μέσω των τροπολογιών τις οποίες κατέθεσαν οι συνάδελφοι αλλά και εγώ ίδιος. Θα ήθελα να επιμείνω σε τρία βασικά σημεία. Πρώτον, η πολυμερή συμφωνία την οποία προωθούμε με την Κολοβία και το Περού. Βρίσκεται σε τεχνική φάση, ήδη έχουν ξεκινήσει δηλαδή αναλυτικότερα συζητήσεις με τους χιώδεις συζητητές, με την κυρία Βέμπερ, με τον κύριο Μενέντες Δεβάγε και με τους συντονιστές της ομάδας των Πρασίνων επίσης ήρθα σε επαφή αλλά η συντονίστρια των Πρασίνων δεν έχει ακόμα καταλήξει σε μια αποφασιστική συνεισφορά θα έλεγα και απλά παραπέμπουμε σε μια πρώτη φάση στην έκθεση Αλμπερτίνη. Δέχομαι τις τροπολογίες οι οποίες έχουν κατατεθεί σχετικά με την ύπατη εκπρόσωπο. Τίθεται και από άλλες τροπολογίες το θέμα της ισότητας των φύλων Υπάρχει ένα θέμα το οποίο παρουσιάζει προβλήματα, είναι το Ευρωλατινικό Ίδρυμα, Ευρωπαϊκό Λατινικό Ίδρυμα. Κάποιοι πιστεύουν ότι θα πρέπει να είναι δημόσιος ο χαρακτήρας του Ιδρύματος αυτού, κάποιοι άλλοι ότι θα έπρεπε να είναι ιδιωτικός. Εν πάση περιπτώσει εδώ υπάρχουν διστάμενες απόψεις. Για να αποφύγουμε αυτές τις διαφορές εγώ είμαι διατεθειμένος να προτείνω κάποιες συμβιβαστικές τροπολογίες οι οποίες θα έχουν σαν στόχο να μην διευκρινίζουν με επαρκώς το χαρακτήρα αυτού του Ιδρύματος αλλά τουλάχιστον να παίρνουν τις βασικές αποφάσεις που απαιτούνται για την δημιουργία του. Εδώ έρχεται και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία είναι ιδιαίτερα εύθετη. Υπάρχουν βέβαια κάποιοι οι οποίοι από κάποιες πολιτικές ομάδες θεωρούν ότι είναι ανεπαρκής η δήλωση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εκεί υπάρχει μια επιπλέον διαφορά η οποία συνεχίζει να μένει, να παραμένει και ελπίζω ότι μέχρι τη στιγμή που θα φτάσουμε στην ψηφοφορία Ίσως να μπορέσουμε να έχουμε καταλήξει σε μια καλύτερη συμφωνία όπως έχει συμβεί και σε προηγούμενες περιπτώσεις. Επαναλαμβάνω ότι και σε συνεργασία με τον Λούκατσεκ ε, προσπαθήσαμε να προωθήσουμε κάποιες τροπολογίες, αλλά είμαι στη διάθεσή του για να του εξηγήσω ό,τι ακριβώς έχει ανάγκη για να συμφωνήσουμε σε κάποια φάση. Καταβάλουμε λοιπόν κάθε προσπάθεια γιατί η, η, η αυτή η έκθεση ε, ε, χρειάζεται σαν τον περισσότερο υποστήριξη ακριβώς για τη στρατηγική σημασία. Ευχαριστώ κύριε Σαλαφράγκα για την ε, παρέμβασή σας και για το γεγονός ότι είσαστε έτοιμος να συνεργαστείτε με τους υπόλοιπους συναδέλφους. Ε, Μενέντες Δενβάλε ζήτησε το λόγο να τοποθετηθεί. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βεβαίω, εγώ ήδη έχω συγχαρεί τον εισηγητή. Έχουμε μακροχρόνια εμπειρία σε αυτέ τι εργασίε. Να μην ε, καθυστερήσω καθόλου σαν αφορά τι ε, τροπολογίε μου, γιατί ήδη έχουν ε, ληφθεί υπόψη. Απλά και μόνο να εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία για να υπενθυμίσω σε όλους τους συναδέλφους που είναι παρόντες ότι αυτή η έκθεση είναι μέρος των προσπαθειών που καταβάλει η Επιτροπή μας αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδώ και καιρό έτσι ώστε να είναι όλο και πιο ορατό το θέμα της Λατινικής Αμερικής και η στρατηγική εταιρική σχέση, η διαπεριφερειακή εταιρική σχέση ε, στην κοινή γνώμη αλλά και στις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιμένω, πρόκειται για μία μόνιμη ε, προσπάθεια που έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό και νομίζω ότι εξακολουθεί να είναι απαραίτητο να συνεχιστεί η προσπάθεια αυτή. Διότι ούτε η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη ε, στο σύνολό τη, αλλά ούτε και όλε οι κυβερνήσει των χωρών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά την άποψή μου, είναι ενημερωμένοι στον επαρκή βαθμό για την πραγματικότητα στη Λατινική Αμερική. Ταυτόχρονα, πιστεύω, δεν έχουν συνειδητοποιήσει ε, το πόσο σημαντικά είναι ορισμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει η συγκεκριμένη περιοχή. Προβλήματα που, κατά την άποψή μου, έτσι, προβλήματα που με την απαραίτητη βοήθεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μόνο θα μπορέσουν να εξελιχθούν, αλλά θα μετατραπούν σε ευκαιρίες. Και τέλος, για να μην καθυστερήσω πολύ, θα ήθελα να πω ότι υπάρχει κι άλλος ένας λόγος έτσι ώστε η Ευρώπη, οι κυβερνήσεις και η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη ε, πρέπει να απασχολούνται όλο και περισσότερο ε, με το πρόβλημα της Λατινικής Αμερικής. Γιατί για λόγους κουλτούρας, πολιτισμού, ιστορίας και κοινών αξιών, κατά την άποψή μου, δεν υπάρχει άλλη περιοχή στον κόσμο που να ε, βλέπει τόσο ευνοϊκά τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα θέλω να πω πρόεδρο και ευχαριστώ. Grazie, Κυρία Γιαννάκου, παρακαλώ. Πολύ κύριε Πρόεδρε, θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή μας, ο οποίος άλλωστε είναι και έχει εργαστεί πάρα πολύ στο θέμα των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Λατινική Αμερική. Θεωρώ ότι η έκθεση του είναι εξαιρετική, δεν χρειάζεται να είναι πολύ μακρά. Ήθελα να κάνω μία μόνο επισήμανση. Δεν έχω υποβάλει τροπολογίες, αλλά το ζήτημα των πολιτιστικών σχέσεων ε, νομίζω ότι είναι μεγάλης αξίας για τη σχέση με τη Λατινική Αμερική και δεν έχει αναφερθεί αρκετά βέβαια. Η εταιρική σχέση αντιλαμβάνομαι ότι περιορίζεται από τα όσα μέχρι σήμερα έχουν συμβεί και από τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά ίσως θα είχε κάποια αξία ε, να γίνει μία αναφορά από τον ίδιο τον εισηγητή ε, διατροπολογίας και να δοθεί έμφαση Ζήσαμε στη δεκαετία του 80 τη σχέση, εγώ τότε είχα αρμοδιότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη Λατινική Αμερική, σε μια εποχή που οι χώρες αυτές είχαν δικτατορία. Και η μεγαλύτερη έμφαση που δινόταν τότε ήταν ακριβώς το να αλλάξει το πολιτικό σύστημα, να γίνουν δημοκρατίες. Σήμερα νομίζω ότι μπορούμε ε, να διευρύνουμε πολύ περισσότερο τη σχέση μας με τη Λατινική Αμερική, ακριβώς σε αυτό το πεδίο, διότι πράγματι, όπως είπε και ο προηγούμενος συνάδελφος, δεν υπάρχει καμία άλλη περιοχή του κόσμου που να είναι τόσο κοντά από πλευράς αξιών και πολιτισμού δύο ήπειροι, όπως είναι η Ευρώπη με τη Λατινική Αμερική. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριο Στάνοκ, έχει το λόγο. Um, Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, πρώτα απ' όλα να, συγχαστώ, να συγχαρώ τον Ιγνάσιο Σαλαφράγκα για την εξαιρετική έκθεση. Τώρα διαβάζω τις συμβαστικές τροπολογίες που είναι πάρα πολλές. Νομίζω πως είναι πολύ εύκολο εδώ μέσα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ξεχνάμε ή να αφήνουμε κατά μέρο τη στρατηγική σχέση που πρέπει να έχουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Λατινική Αμερική. Ε, ειδικά την τελευταία δεκαετία με τη διεύρυνση και τις προκλήσεις που έχουμε με τις σχέσεις ε, με τη Ρωσία, Κίνα, Νότια Ασία κτλ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε λοιπόν την Λατινική Αμερική που μας απασχόλησε περισσότερο στη δεκαετία του 80 και 90 πιο πολύ από ότι μετά τη διεύρυνση. Και βεβαίως πρέπει να εστιάζουμε και στους δύο στρατηγικούς παίκτες, Βραζιλία και Μεξικό, αλλά υπάρχουν και άλλες δυνάμεις, ειδικά η Κολομβία, η Χιλή και η Αργεντινή, την πολιτική δυναμική των οποίων πρέπει να παρακολουθούμε στενά. Και νομίζω πως είναι σημαντικό να ενισχύσουμε καλύτερες εμπορικές και πολιτικές σχέσεις μεταξύ των υπήρων και ειδικά πρέπει να αντισταθούμε στις πιέσεις που υπάρχουν εδώ μέσα να σταματήσουμε τις συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου, ειδικά όσες μελετάμε αυτή τη στιγμή η Κολομβία με τις κατηγορίες αυτές περί παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την κυβέρνηση για τις οποίες δεν υπάρχει βάση. Εγώ θεωρώ πως μοιραζόμαστε ένα κοινό πολιτισμό με βάση κοινέ αξίες με τη Λατινική Αμερική και πρέπει να προσπαθήσουμε να προστατεύσουμε τις εύθραυστες ε, παραδόσεις κοινοβουλευτικής δημοκρατίας σε αντίθεση με τους διάφορους ε, καοτήγιο που υπάρχουν σε αυτές τις ε, χώρες την άνοδο του τσαβισμού στη Βενεζουέλα που συνεργάζεται με το καθιστός Κάστρο στην Κούβα για να εξαγάγουν αυτή τη, τη μορφή διακυβέρνησης σε χώρες με πλουραλιστικές δυτικές δημοκρατικές παραδόσεις και προσπαθούν να επιβάλλουν εν σοβιετικού τύπου αυταρχικό καθεστώς, κάτι στο οποίο η ομάδα μου θα αντιταχθεί. Έχω πρόβλημα με κάποιες ε, τροπολογίες ε, που θέλουν να θέσουν και ζητήματα δικαιωμάτων ή προβλημάτων λατινοαμερικανικής μετανάστευσης ως ένα ζήτημα πολυμερές. Σε κάποια κράτη-μέλη και ειδικά στο δικό μου, οποιαδήποτε πολιτική ανοιχτών θυρών για τη μετανάστευση με αφετηρία την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απαράδεκτη και κατά την άποψή μου αποτέλεσμα θα έχει μόνο περισσότερη αντιπάθεια για την Ευρωπαϊκή Ένωση και μεγαλύτερη δημοτικότητα των ακροδεξιών κομμάτων. Οπότε εμείς θα καταψηφίσουμε αυτές τις τροπολογίες. Συνάδελφο Βέμπερ, που είστε και σκιώδη συγγήτρια εξ ονόματος της Ομάδας Φιλελευθέρων. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα επιτρέψτε μου να συγχαρώ ε, τον εισηγητή. Είναι πολύ καλή και ολοκληρωμένη έκθεση και για να ε, για καταλάβουμε ε, τι εκπροσωπεί αυτή η προσπάθεια, καταλάβουμε ότι ε, τυποποιήθηκαν πάνω από 120 τροπολογίες και πραγματικά δεν ήταν εύκολο να εργαστεί κανείς με τόσες πολλές τροπολογίες. Εδώ έχουμε μία έκθεση που αφορά τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις σχέσεις με τη Λατινική Αμερική. ε, πολλές τροπολογίες ε, που αναφέρονται στις λεπτομέρειες μιας τέτοιας στρατηγικής και που δεν πρέπει να γίνουν δεκτές. Ταυτόχρονα όμως να πω ότι ε, λαμβάνοντας υπόψη τις ε, αρχές ε, των φιλελευθέρων για την υποστήριξη των ανθρωπινών δικαιωμάτων, για τα ισότιμα δικαιώματα, θέλω να πω ότι ενώ υποστηρίζουμε ιδιαίτερα τη φιλοσοφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. για, προς την κατεύθυνση των περιφερειακών διαπραγματεύσεων, ε, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να μην αφήσουμε στην άκρη μία χώρα και να μην τους απομονώσουμε. επειδή ε, ε, συμβαίνουν ορισμένα γεγονότα στη συγκεκριμένη περιφέρεια και μπορεί να μην θέλουν όλε οι χώρε να αναπτύξουν σχέσει σχέση στον ίδιο βαθμό με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πράγματι, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εξετάσει με πολύ μεγάλη προσοχή ε, τη Λατινική Αμερική. Και όσον αφορά αυτό το ευαίσθητο θέμα, για παράδειγμα, τη μετανάστευση. από τη μια μεριά έχουμε ε, την Κεντρική και την Νότια Αμερική που ζητά ε, μια ειδική ρύθμιση στον αφορά τη μετανάστευση. Και από την άλλη έχουμε αυτή την ε, ε, πολιτική που περιέγραψε ο συνάδελφος ω πολιτική ε, κλειστής πόρτας. Ε, το θέμα είναι ότι δεν θα πρέπει να κλειστούμε τη μία την άλλη οδό με απόλυτο τρόπο, αλλά να δούμε το θέμα της καλύτερης εκπαίδευσης στη Λατινική Αμερική, της περισσότερης απασχόλησης, της ε, δυνατότητας για μια αξιοπρεπή ζωή εκεί, ε, τότε αν αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα, τότε ίσως να μην έχουμε και τόσο πολλοί μετανάστες στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Για μια φορά το λέω ότι η συνεργασία ήταν ιδιαίτερα επικοδομητική και με την ομάδα του Σοσιαλιστών και με τον εισηγητή. ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Συνάδελφο ε, Λούνατσεκ από τους Πράσινους, επίση και ο εισηγητή. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να αρχίσω με ε, τη διαδικασία όσον αφορά τις τροπολογίες. Κάτι που με ανήσυχε ιδιαίτερα. Στη συνέχεια θα αναφερθώ στην ουσία. Εδώ και ένα χρόνο έχω αναλάβει τα καθήκοντά μου ως μέλος του Κοινοβουλίου. Για δέκα χρόνια ήμουν στο Κοινοβούλιο της Αυστρία και έχω διαπραγματευτεί πολλές εκθέσεις. Αυτή τη φορά πρέπει να σας πω ότι περίμενα ο εισηγητής, ο κύριος Ελαφράνκα, να συνεργαστεί και να πλησιάσει όχι μόνο τις δύο μεγάλες ομάδες, σοσιαλδημοκράτες και τους φιλελεύθερους, αλλά και τους πράσινους. Δεν έγινε όμως κάτι τέτοιο και θέλω να εκφράσω τη λύπη μου για το θέμα αυτό ε, δημόσια. Το είπα κατηδίαν ε, στον κύριο Σαλαφράγκα. Χθε εγώ τον πλησίασα για να τον ρωτήσω τι γίνεται με, τις, με τους συμβασμούς κτλ. ε, ο κύριος Μίλαν Μον ε, μου, ε, μου, μου, έδωσε τους, ε, τις συμβαστικές προτάσεις του κύριου Μενέντες και του ίδιου του συγκητή. Η διαδικασία αυτή με, δεν με ικανοποιεί καθόλου. Θα ήθελα λοιπόν να μα είχε δοθεί η δυνατότητα διαπραγμάτευση με τον εισηγητή για να δούμε τι δεσμεύσει, τι συμβασμού θα μπορούσαμε να έχουμε πετύχει. Ε, και όχι σήμερα έτσι πολύ ε, βεβαιασμένα να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε κάποιε συμφωνίε. Αυτό το λέω ε, εν είδη εισαγωγή. Και εκφράζω τη λύπη μου για το γεγονό ότι ακολουθήθηκε αυτή η διαδικασία. Γιατί κατά την άποψή μου και κατά την άποψη τη ομάδα των Πρασίνων, οι σχέσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση με την ε, ε, Λατινική Αμερική και με την Καραϊβική ε, είναι ουσιώδου σημασία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ζήτημα αυτό. Και προσωπικά πρέπει να σα πω ότι έχω μακρά εμπειρία σε πολιτικό επίπεδο και επαφών με την κοινωνία των πολιτών στη Λατινική Αμερική. Μα ανησυχεί πολύ το ζήτημα αυτό και θα ήθελα ε, η έκθεσή μας πραγματικά να αντιπροσωπεύει ολόκληρο το Κοινοβούλιο ή τουλάχιστον όσο, την ώστε να δουν ευρύτερη πλειοψηφία και όχι μόνο τις βασικές πολιτικές ομάδες. Φαίνεται ότι εδώ ε, προσπαθείτε να, να, δείξετε ότι είστε πλειοψηφία, μα είστε πλειοψηφία. Αλλά πραγματικά θέλω να ζητήσω από όλους στι μελλοντικέ διαπραγματεύσει να συμπεριλαμβάνετε, να συμπεριλαμβάνετε και τι άλλε πολιτικέ ομάδε. Αυτό εν είδη αγωγή, όπω σα είπα. Και, το, και τώρα να αναφερθώ σε ορισμένε λεπτομέρειε. Χαίρομαι γιατί ο κύριο Σαλαφράγκα συμπεριέλαβε ορισμένα από τα θέματα τα οποία ε, προτείναμε εγώ και η ομάδα μου. Για παράδειγμα, την αναφορά ε, στην ευρωπαϊκή προσέγγιση στο χάρτα, στη Χάρτα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στο θέμα της βίας κατά των γυναικών, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο αυτό. Επίσης, το θέμα της ατιμορρησίας που κυριαρχεί σε πολλές χώρες της Λατινική Αμερικής η καταπολέμηση της ε, κλιματικής αλλαγής ε, και δεχθήκατε να το διατυπώσετε με περισσότερη ισχύ. Αυτά είναι πράγματα που μας ε, ικανοποιούν. Θα ήθελα όμως να έχουμε πετύχει περισσότερους συμβασμούς. Αυτή τη στιγμή όσον αφορά αυτά που βλέπω και δεν είχα το, το χρόνο να διαβάσω τους συμβασμούς που μας μοιράστηκαν μόλις πριν από λίγο, ίσως ορισμένα πράγματα στα οποία θα μπορούσαμε να βρούμε κάποια συμφωνία είναι για παράδειγμα σε ένα συγκεκριμένο σημείο όπου εμείς θέλαμε να μιλήσουμε για πηγές ανανεώσιμης ενέργειας. Αλλά βλέποντας επίσης και με κριτικό μάτι τα, τις, μεγάλα υδροελεκτρικού, τους μεγάλους υδροελεκτρικούς σταθμούς που γίνονται σε ορισμένες χώρες ε, της Λατινικής Αμερικής, όπως παράδειγμα η Βραζιλία. Ε, έργα που προέρχονται από άλλες εποχές και που είναι, και που είναι επικίνδυνα και για, το, και το περιβάλλον αλλά και για τους αυτόχθονες. Άρα λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει ε, ώστε να τον ευρύτερη συνένεση και να δούμε κατά πόσο αξίζουν τον κόπο αυτά τα έργα. Αλλά δεν ε, βλέπω τίποτα για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά για ενέργειες ε, που μολύνουν λιγότερο. Εσείς μπορεί να θεωρείτε ότι αυτό είναι λεπτομέρεια, αλλά γνωρίζουμε ότι αυτοί που υποστηρίζουν την πυρηνική ενέργεια ως πηγή καθαρή εντός εισαγωγικών, ακριβώς προτιμούν αυτήν την ορολογία, να μιλάμε για λιγότερο ρηπαίνουσες μορφές ενέργειας. Εγώ όμως θα το ξεκαθαρίσω. Η πυρηνική ενέργεια μπορεί να μην ρηπαίνει, μπορεί να μην μολύνει το περιβάλλον και να μην συμβάλλει στην αλλαγή του κλίματος, αλλά κοιτάξτε, πρόκειται για ε, ιδιαίτερα ρηπαίνουσα πηγή ενέργειας. Κάτι άλλο Μα ενδιαφέρει και εδώ κύριε Ρεσαλαφράνκα έχω μια ερώτηση. Γιατί στι κατηδίαν συνομιλίε μα μου είπε ότι και ο κύριο Ρεσαλαφράνκα θα προτιμούσε να ε, έχουμε ε, μια αναφορά ε, σε αυτά τα οποία γίνονται στη Γουατεμάλα, στο Μεξικό και αλλού. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε κατά πόσο θα συμπεριλάβετε για αυτά τα θέματα. Κάτι το οποίο είναι δύσκολο για μας, τους πράσινους, κάτι που είναι δύσκολο να δεχθούμε, αφορά το σημείο 16, εκεί όπου αναφέρει τις διαπραγματεύσεις για τη Συμφωνία Σχέση Σχέσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Κεντρική Αμερικής. Να ολοκληρωθεί πριν από τη διάσκεψη κορυφή τη Μαδρίτη. Κοιτάξτε, ε, εδώ ε, να σας πω το εξή και συμφωνούν πολύ όχι μόνο από την ομάδα μου η κατάσταση ε, στην Οδούρα ε, και πώς τη χαρακτηρίζουμε. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν ότι ότι όταν έχουμε μια κυβέρνηση η οποία βρίσκεται παράνομα στην εξουσία μπορούμε να εξακολουθούμε να έχουμε διαπραγματεύσεις με μια τέτοια κυβέρνηση μια τέτοια χώρα. Για τη Συμφωνία ιταλικής Σχέσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Κεντρικής Αμερικής. Και τέλος, ο κύριος Σελαφράκα αναφέρεται στο ότι στην ε, ικανοποιητική ολοκλήρωση της Συμφωνίας Πολυμερούς Εμπορίου ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις χώρες της κοινότητας των Άνδεων. Ξέρουμε ότι εδώ πρόκειται μόνο για την Κολομβία και το Περού. Αλλά για να το δεχτούμε αυτό, για μας είναι σημαντικό να πούμε ότι εκφράζουμε τη λύπη μας για το ότι η ιδέα ε, μιας ευρύτερης συμφωνίας ε, ε, σύνδεσης με ολόκληρη την κοινότητα των Άνδεων εγκαταλείφθηκε, τα μέλη δηλαδή της κοινότητας των Άνδεων. Αυτά προς στιγμή και ελπίζω πραγματικά να υπάρξουν άλλες διαπραγματεύσεις. Ξέρω ότι αύριο το πρωί έχουμε την ψηφοφορία και ελπίζω στο μέλλον πραγματικά να καταφέρουμε να έχουμε μια έκθεση που να συμπεριλαμβάνει τις απόψεις και τις ιδέες όλων των ομάδων του Κοινοβουλίου για να βελτιωθούν πραγματικά οι σχέσει ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Λατινική Αμερική. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ, συνάδελφε Λούνατσεκ. Ο Βίλι Μάιερ είναι ο επόμενο ομιλητή. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να πω στον κύριο Σαλανφράκα ότι οι συμβαστικέ τροπολογίε ε, έφτασαν σε μένα μόλι τώρα. Οπότε για μένα είναι πολύ δύσκολο να το πιστεύω. Πάνω σε αυτές Κοιτάξτε, πραγματικά καταβάλει σημαντική προσπάθεια και το αναγνωρίζω αυτό ο κύριο Αλαφράγκα για να αποφευθούν οι πλέον ε, δύσκολες ε, ζώνες. Από την προοπτική της Λατινικής Αμερικής και, της, ε, και των χωρών της Καραϊβικής. Υπάρχει ένα, και εδώ υπάρχει μια κεντρική, ένα κεντρικό σημείο το οποίο το ξεπέρασε ε, χωρίς να επισέλθει στην ουσία. Εφείς! αναφέρομαι σε αυτή την αιμονή της Ευρωπαϊκής Ένωσης να θεωρεί ότι τα πάντα πρέπει να μετατραπούν σε συνθήκη ελεύθερου εμπορίου. Και άλλες φορές ε, είχαμε σκληρές συζητήσεις και διαπραγματεύσει για το θέμα αυτό. Με ευφύη τρόπο λοιπόν πέρασε ξαπαλώνων ήχων το θέμα αυτό. Ο εισηγητής. Και άλλωστε εμείς οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να δούμε ότι ε, να αποφεύγουμε κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το κάνουμε. Να ε, υπαγορεύουμε και να δίνουμε μαθήματα για το πώς πρέπει ε, να επιτυγχάνεται η περιφερειακή ολοκλήρωση. Εγώ ζω στο, σε επίπεδο Eurolat και πραγματικά πρέπει να σας πω ότι βλέπω τα... Ε, βλέπω τι γίνεται. Εμεί είμαστε έτοιμοι να διδάξουμε του πάντε, για το πώ πρέπει να ε, κάνουν το α ή το β. Και ταυτόχρονα τολμάμε να λέμε στου γείτονε γείτονες Αμερική και στην Καραϊβική για το πώ πρέπει να πετύχουν την ολοκλήρωσή του. Ε, κοιτάξτε, πραγματικά όλα αυτά δημιουργούν μια κατάσταση ιδιαίτερα περίπλοκη όσον αφορά τις σχέσεις ε, που, που, που λέμε ότι είναι στρατηγική σημασία. Για παράδειγμα, εγώ θα έλεγα στον κύριο Σαλαφράγκα το εξή. Όταν ε, προβαίνουμε σε κριτικέ για παράδειγμα, όσον αφορά τι θα δαπάνε, σε βάσιμε κριτικέ. Αυτέ τι κριτικέ να τι απευθύνουμε και στην Ευρώπη. Δηλαδή λυπούμαστε για την αύξηση των δαπανών στη Λατινική Αμερική και στην Καραϊβική, ενώ ταυτόχρονα ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δαπανά 8 φορές περισσότερα σύμφωνα με το ΣΥΠΡΙ. Επομένως, καταλαβαίνετε θέλω να πω, αν εγώ είμαι μια χώρα τη Λατινική Αμερική ή τη Καραϊβική και ακούω αυτέ τι κριτικέ από του Ευρωπαίου, θα, θα, σκεφτώ, μα αυτοί τι κάνουν. Δηλαδή, εσεί πάτε σε ένα συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο και ταυτόχρονα εσεί ε, και κάνετε αυτή την κριτική και ταυτόχρονα εσεί κάνετε αυτέ τι θετικέ δαπάνε, μάλιστα και σε όπλα μαζική καταστροφή. Και μα λέτε σε εμά, θα έλεγα εγώ, ότι εμεί είμαστε κακοί. Ε, τι να σα πω. Άρα λοιπόν πρέπει να αποφεύγουμε τα μαθήματα στου άλλου. Για την ομάδα μα λοιπόν είναι σαφέ ότι δεν μπορούμε να περνάμε έτσι επιφανειακά ορισμένα ζητήματα, όπως για παράδειγμα η, καθαρά αρνητική αξιολόγηση της συμφωνίας σύνδεσης με την Κολομβία. Γιατί στο τμήμα που αναφέρεται στον πολιτικό διάλογο, το γεγονό ότι μια χώρα όπω η Κολομβία δολοφονεί ε, συνδικαλιστέ ηγέτε, ότι ανακαλύφθηκε πρόσφατα ένα ε, κοινό τάφο με πάνω από το 2.500 θύματα, ότι ε, ε, κυριαρχούν παραστρατιωτική διαφθορά κτλ. Ε, τι να σα πω, νομίζω ότι μπορούμε όλα αυτά να τα παραγνωρίζουμε. Καταλαβαίνω βεβαίω ότι υπάρχουν ε, εδώ άνθρωποι στο Κοινοβούλιο που όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα ακολουθούν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Εγώ όμω δεν συμφωνώ. Και γι' αυτό νομίζω ότι είναι πολύ λεπτό το ζήτημα αυτό. Όπω όπως επίση και το θέμα τη de facto αναγνώριση των βουλευτικών και προεδρικών εκλογών στην Ονδούρα. Επρόκειτο για στρατικό πραξικόπημα και οι συνέπειες αυτού του πραξικοπήματος ε, ήταν τρομερές, ε, θάνατοι, δεινά και τώρα ε, γίνεται προσπάθεια νομοποίησης μια κυβέρνησης, κυβέρνησης που ανήλθε στην εξουσία με στρατιωτικό πραξικόπημα. Όπως είπα στην αρχή λοιπόν, ε, σας λέω και τώρα, ότι υπάρχουν βαθιές ανησυχίες από την Λατινική Αμερική και την Καραϊβική. Δηλαδή όταν μιλάμε για εμπόριο, πάντα μιλάμε για ελεύθερο εμπόριο. Πάντως βλέπω θετικά την προσπάθεια του κ. Σαλαφράγκα να αποφύγει ε, να θέσει αυτό το δίλημα και γιατί, και γιατί υπάρχουν χώρες όπως το Εκουαδόρ που στην τελευταία συνταγματική μεταρρύθμιση απαγόρευσαν την υπογραφή μια συνθήκη ελευθέρου εμπορίου. Απαγορεύεται έτσι από το Σύνταγμα του Εκουαδόρ με βάση ε, την κακή εμπειρία του παρελθόντος και τις προηγούμενες συνθήκες ελεύθερου εμπορίου. Άρα είναι κατακλείδη. Η ομάδα μου σημειώνει την προσπάθεια του κ. Σαλαφράκα για να αποφύγει μία έκθεση ε, που να περιέχει πάρα πολλά φιλοκόμενα σημεία. Όσον αφορά πάντως ε, ε, την διαπεριφερειακή αυτή στρατηγική σχέση. Εμείς απέχουμε πολύ από την προσέγγιση που ακολουθεί εδώ. Εμείς θέλουμε μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη με προώθηση των δημοσίων υπηρεσιών, του εργατικού δικαίου, των, δικαιωμάτων των ε, αυτοχθόνων, ε, την καταπολέμηση της ανεργίας, συγκεκριμένα μέτρα για την, για την επίτευξη των στόχων της χιλιετίας. Δηλαδή έχουμε μια εναλλακτική θεώρηση αυτό όμως το οποίο, ε, στο οποίο στέκομαι και στο οποίο στέκεται η ομάδα μου είναι αυτή την προσπάθεια ε, που κατέβαλε ο κύριος Αλαφράγκα για να αποφύγει τα διάφορα επικίνδυνα σημεία. Όσον αφορά τις διμερείς σχέσεις μεταξύ των χωρών της περιοχής και την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να σας πω ότι πάντα το θέμα της μετανάστευσης και με βάση και την οδηγία ε, για την επιστροφή, ορισμένη την ονομάζουμε οδηγία της ντροπή πάντως, εδώ πρέπει να δούμε ότι αποτελεί ένα πολύ, σοβαρό, πολύ μεγάλο εμπόδιο για, την, ε, για τις ομαλές σχέσεις ανάμεσα στις δύο περιοχές. Γιατί είναι αλήθεια ότι δεν μπορεί να καταλάβει κανείς το γεγονός ότι παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ε χρειάζεται μετανάστευση, λαμβάνοντας, για, για την ίδια μας την ύπαρξη, λαμβάνοντας υπόψη ε, το βαθμό γύρανσης του πληθυσμού, ταυτόχρονα τους μετανάστες ε, τους αντιμετωπίζουμε σαν εγκληματίες, ε, που βρίσκονται στη φυλακή χωρίς καν να έχουν περάσει από δίκη. Άρα εδώ νομίζω ότι η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική θα εξακολουθεί να ζητά την παρέκκληση και την υπέρβαση αυτή τη οδηγία για την επιστροφή. Αυτά ήθελα να πω και ευχαριστώ. Οι δύο τελευταίε ομιλίε πριν πάρει το λόγο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή εκπρόσωπος, ο κύριος Μονιές Δεοκίσα και αμέσως μετά ο κύριος Αγκουράκης. Ευχαριστώ και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Σαλαφράκα και του ε, σκιώδει ηγητέ ε, των ομάδων για την έκθεση και για τι συμβαστικέ τροπολογίε. έτσι ώστε να έχουμε μια εκθέση που να χαρακτηρίζεται από ισορροπία και να αντικατοπτρίζει το ποιε είναι και ποιε θα έπρεπε ε, να είναι οι στρατηγικέ στη σχέση μα με την Δυτική Αμερική. Θα ήθελα όμω. Βεβαίω δεν είχα το χρόνο για να δω με την ησυχία μου τι συμβαστικέ τροπολογίε, αλλά θα ήθελα να σα πω ότι αν δεν συμπεριληφθεί η προφορική τροπολογία στην οποία αναφέρεται η χιλή και ο σεισμός στη χιλή. Πρέπει. Α, έχει συμπεριληφθεί. Α, ωραία, τότε. Εντάξει. Μια και έχω το χρόνο, λοιπόν, να, ευχαριστή, να σα ευχαριστήσω που συμπεριλάβατε το θέμα τη Χιλή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και στο, όσον αφορά το μέλλον. Τόσο η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, όσο και η πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τι προσπάθειε ανασυγκρότηση στη Χιλή. Και όσον αφορά τη συμφωνία, την πολυμερή συμφωνία με την, με την Κολομβία και με το Περού, σήμερα ε, πήραμε μια ανακοίνωση επίσημη από τον, ε, ε, από τον οργανισμό της Λατινικής περιοχής, τον Οργανισμό Ιβερομερικών Κρατών, Κρατών, για, και να λάβουμε υπόψη την πρόοδο που έχει, την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε διεθνές επίπεδο. Δεν υπάρχει αμφιβολία για το ότι έχει σημειωθεί πρόοδο στις χώρες αυτές όσον αφορά τα διάφορα δικαιώματα. Γιατί ε, ε, μερικές φορές υπάρχουν επικρίσεις. Όσον αφορά την Κολομβία, σίγουρα υπάρχει πρόοδος και έχουμε την επίσημη επιστοποίηση από τον Οργανισμό Ιβυροαμερικανικών Κρατών για το ότι υπήρξε η πρόοδος αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σαγκουράκης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα το συντομότερο δυνατόν να επισημάνω τα εξή. Κατά την ε, γνώμη μου και μιλάω ως Κομμουνιστικό Κόμμα, όχι ως ομάδα της ε, αριστεράς. Η έκθεση που παρουσιάζει ο κύριος ε, Σαλαφράνκα ε, πάει σε δύο κατευθύνσεις ε, άσχημες. Το πρώτο είναι η ιδιωτικοποίηση των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Λατινική Αμερική και επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο διότι δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεται συζήτηση το ίδρυμα που θα παρακολουθεί την υλοποίηση της συμφωνίας να είναι ημιδιωτικό, να χρηματοδοτείται από εταιρείε κτλ. κτλ. Διότι όπω γνωρίζουμε όποιο πληρώνει ελέγχει. Δεν θα μπορούσε δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει μηχανισμούς, γραμματείε για να ελέγχει την ε, υλοποίηση της συμφωνίας χρειάζεται αυτό το ίδρυμα, η Δεύτερον, στρατιωτικοποίηση των σχέσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Λατινική Αμερική, διότι τα όσα αναφέρονται στο άρθρο που έχουν σχέση για τη δημιουργία μιας ε, σχέσεις για ζητήματα ειρήνης και ασφάλειας κτλ. Ε, μάλιστα είναι το άρθρο 11. Ακριβώς επειδή γίνεται λόγος για αντιμετώπιση κοινών απειλών και γνωρίζουμε, εν πάση περιπτώσει, πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση διατυπών τις απειλές, φαντάζομαι ότι το ίδιο θα απαιτούν και από τους Λατινοαμερικανούς. Την εποχή που στη Λατινική Αμερική έχουμε μια φοβερή διείσδυση ξανά των Ηνωμένων Πολιτειών, με τις βάσεις που όπως γνωρίζετε έχει στην Κολομβία, με αυτά που συμβαίνουν στην Αϊτή και όπου κατά τη γνώμη μου η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κάνει τίποτα άλλο από ότι να βοηθεί του Αμερικανού στο έργο αυτό. Εξάλλου για την ιδιαίτερη σχέση τη Ευρωπαϊκή Ένωση με ΗΠΑ τα ακούσαμε και πριν. Τρίτο ζήτημα, κοινή θέση. Δεν είναι δυνατόν να συζητάμε για ένα τέτοιο πράγμα και να μην θίγεται το θέμα τη απαράδεκτη κοινή θέση τη Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στην Κούβα. Και όσο βεβαίω διατηρείται αυτή η κοινή θέση, Αφενός, όσο όμως από την άλλη πλευρά αυξάνει η επιρροή της Κούβας στη Λατινική Αμερική και ας λένε μερικοί διάφορα πράγματα εδώ, τόσο σε χειρότερη θέση θα βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τέλος, είναι απαράδεκτη η θέση όσον αφορά τη μετανάστευση. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό το πρόβλημα να λυθεί με αυτόν τον τρόπο. Ε, χρειάζεται να υπάρχει ε, νομοποίηση των μεταναστών και τέλος ή θα είναι σε ισότιμη βάση η σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη Λατινική Αμερική ή δεν θα υπάρχει καθόλου. Αυτά που λέγονται στην έκθεση, ότι να προωθηθούν σχέσεις ε, ε, μεταβλητής γεωμετρίας, τριγωνικά σχήματα κτλ. δεν θα τα δεχτούν οι Αμερικανοί. Ευχαριστώ πολύ. Κάστρο Καστρίο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να προσθέσω και τη φωνή της Επιτροπής στα συγχαρτήρια προς τον κύριο Σαλαφράκα για το σχέδιο έκθεσης και για τις προσπάθειες που καταβάλει για να βρεθούν συμβαστικές λύσεις στα διάφορα σημεία τα οποία ετέθησαν από τα υπόλοιπα μέλη του Κοινοβουλίου. για άλλη μια φορά συμβάλλει με βοηθητικό τρόπο, όπως και στο παρελθόν, για την ενίσχυση των σχέσεων ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Λατινική Αμερική. Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλει ε, ιδιαίτερα στο, στο στόχο στον εξή στόχο, να γίνει η περισσότερο γνωστή η Λατινική Αμερική και στι κυβερνήσει και στου πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπω ήδη ελέγχθη και στην έκθεση αναφέρεται πολύ σωστά, πρόκειται για δύο περιοχέ που από κοινού ε, έχουν πάνω από ένα δι κατοίκου, 60 κράτη, ε, το 1 τρίτο ή το 1 τέταρτο των κρατών των Ηνωμένων Εθνών. Άρα λοιπόν είναι απολύτως απαραίτητο για την Ευρώπη να έχει ε, αυτή τη στρατηγική σχέση με τη Λατινική Αμερική. Επίσης αναφέρθηκε εδώ ιδιαίτερα και αυτό το αναφέρεται και στην ανακοίνωσή μας η της αξιών και κοινή ιστορίας που μας συνδέει με την Λατινική Αμερική. Και πρόκειται λοιπόν για ένα κεκτημένο μέσο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να αξιοποιηθεί σε πολυμερές επίπεδο με ιδιαίτερα σημαντικό τρόπο. Το μόνο που θα ήθελα τώρα είναι να κάνω ορισμένε επιμέρους παρατηρήσεις για το θέμα της περιφερειακής ολοκληρωσής και για τις διαδικασίες που έχουν ξεκινήσει ήδη και βρίσκονται να εξελίξει. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι η πολιτική διαδικασία με την κοινότητα των Άνδρων δεν έχει ολοκληρωθεί, είναι ανοιχτή και πριν από δύο εβδομάδες είχαμε μία συνεδρίαση της Μικτής Επιτροπής, της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Κοινότητας των Άνδεων που διεξήχθη σε ιδιαίτερα επικοδομητικό πνεύμα με τη συμμετοχή των τεσσάρων μελών. Επίσης γνωρίζουμε ότι το Εκουαδόρ υπέβαλε αίτηση για να προσθεθεί σε αυτή την διαπραγματευτική διαδικασία. Όταν ολοκληρώθηκαν οι τεχνικές διαπραγματεύσεις με την Κολομβία και με το Περού. Επίσης θα να σας πω ότι οι συνεδριάσεις με την Κεντρική Αμερική γίνονται με τη συμμετοχή ε, της Ονδούρας και με την υποστήριξη των χωρών της περιοχής. Προφανώς, ε, να σας πω και το εξής, ότι αύριο θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε για τη Χιλή και για το σεισμό και επειδή εγώ είμαι υπεύθυνο και για τη σχέση με τη Χιλή, εάν η έκθεση αυτή θα μπορούσε να εκπέμψει ένα μήνυμα αλληλεγγύης, προφανώς ε, ε, αυτό θα το βλέπαμε ιδιαίτερα θετικό πνεύμα. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, e ευχαριστώ να δώσουμε τέλος ε, ε την δυνατότητα δευτερολογία στον κύριο Σαλαφράγκα. Χαίρομαι ιδιαίτερα για την έκθεσή σα και σα συγχαίρω για την εξαιρετική εργασία. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλου του συναδέλφου για τι παρεμβάσει του και για αυτόν τον ε, γενικά θετικό και επικοδομητικό τόνο που θέλησα να δώσω στη συζήτηση. Που βεβαίω, γιατί βεβαίω περί αυτού πρόκειται. Νομίζω ότι ο κύριο Μέγερ το είπε πολύ καλά. Νομίζω ότι όταν θέλουμε, όταν στόχο είναι να προωθήσουμε μια στρατηγική σχέση ε, με μια περιοχή του κόσμου όπω η Λατινική Αμερική, πρέπει να έχουμε ε, όραμα και να προσπαθήσουμε να αφήσουμε στην άκρη τα θέματα που μας διαχωρίζουν. Ε, εμείς ε, είμαστε ε, ένα κοινοβούλιο στο οποίο επικρατούν διάφορες ιδεολογίες και διάφορες απόψεις όσον αφορά τα ζητήματα αυτά. Πρέπει να έχουμε λοιπόν την απαραίτητη διάβγεια πνεύματος έτσι ώστε να αφήσουμε στην άκρη τις διαφορές και να προσπαθήσουμε να δούμε ε, πώς μπορούμε να πετύχουμε τη μέγιστη συνένεση σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο όπου θέλουμε να δώσουμε κοινέ απαντήσεις στα κοινά προβλήματα που αφορούν όλους μας. Όταν ε, ήμουν εισηγητή ε, ε, στο κοινοβούλιο αυτό, και αυτό έχει γίνει αρκετά συχνά και πριν από τι διασκέψεις κορυφή, ξεκινώ ήδη από το παγιοποιημένο δόγμα του κοινοβουλίου, λαμβάνω υπόψη ότι οι θέσει εξελίσσονται και λαμβάνω υπόψη και τι θέσει και την εργασία των άλλων συναδέλφων. Έχουμε εδώ τον πρόεδρο της Επιπροσωπής για το Μεξικό, που προετοίμασε για την Eurolat μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα κατά την άποψή μου έκθεση, με πολλέ πρωτοβουλίε, που εγώ θα, θα, θα, θα δεχόμουν χωρίς καμία δυσκολία σχολεία. Επίσης η κυρία Ντεκάιζερ ε, ε, προετοίμασε μια έκθεση για, μια, για ένα χάρτη ανάμεσα σε δύο περιοχέ για την ειρήνη και για τη σταθερότητα. Όλα αυτά αποτελούν και μέρο του δόγματο του Κοινοβουλίου και με βρίσκουν σύμφωνο. Τώρα, να απαντήσω ε, στι συγκεκριμένε ερωτήσει και πολύ σύντομα και στι ανησυχίε που εκφράστηκαν μέσα από τη συζήτηση. Στην κυρία Γιαννάκου, την οποία ευχαριστώ για τα σχόλιά τη και για του επένου τη, ε, μα ε, ρωτά για το εξή, γιατί δεν προσπαθούμε να συμπεριλάβουμε με βάση μια προφορική τροπολογία, γιατί δεν υπάρχει χρόνο για κάτι άλλο την ενίσχυση της πολιτιστικής διάστασης αυτής της, της εταιρικής σχέσης. Πολύ καλή ιδέα. Κρίμα που δεν μας ε, ε, υπέβαλε τροπολογία συγκεκριμένη ε, μέσα στο χρονικό διάστημα υποβολής τροπολογιών, αλλά θα προσπαθήσω να δώσω συγκεκριμένη απάντηση στις, στο αίτημά της. Και συνέχεια. Όσον αφορά την κυρία Λούνατσεκ η οποία εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της γιατί θεώρησε ότι εγώ άσκησα διακριτική μεταχείριση κατά των πράσινων. Προ Θεού, Πρόεδρε, δεν ήταν κάτι τέτοιο καθόλου η πρόθεσή μου. Αυτό το οποίο είπα και στην αρχή και νομίζω ότι το αποδεικνύει και η εμπειρία μου μέσα στο Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι ο κύριο Μέγερ ε, το ανέφερε. Αυτό προσπαθώ είναι να πετύχω το, τη μέγιστη δυνατή συνένεση όχι, κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι είναι λάθος να αγνοούμε ε, τις ε, μειοψηφούσες ομάδες. Άλλο πράγμα είναι όταν, ότι όταν κάποιος αναλαμβάνει τη σύνταξη μιας έκθεσης πρέπει ε, να ε, συντάξει την έκθεση με απόλυτη αυστηρότητα εάν παίρναμε όλες τις τροπολογίε όλων των πολιτικών ομάδων, στην ουσία θα είχαμε ένα μοσαϊκό ε, και επαναλήψεων χωρίς καμία συνοχή. Άρα νομίζω ότι πρέπει ε, ε, όλοι να ξεκινάμε με βάση τον εξή στόχο. Ε, εκθέσεις ε, συνοπτικές, ε, ποιοτικές για να βγαίνουμε και γελοί ενώπιον των πολιτών. Γιατί για μένα είναι πολύ εύκολο να πω σε όλου βεβαίω και τη δική σου τροπολογία ομόφωνα όλα. Χωρί να με απασχολεί το θέμα τη συνοχή και τη ε, παρουσία τη έκθεση. Βεβαίω θέλω θέλω να πω στην κυρία Λούνατσεκ ότι ε, μοιράστηκαν ε, αργά οι συμβασμοί γιατί οριστικοποιήθηκαν σήμερα το πρωί καθυστερημένα. Και υπήρξαν και άλλε σκιώδει συγκητέ και άλλε πολιτικέ ομάδε, στου οποίου δεν ε, απευθύνθηκα. Αυτοί ήρθαν και με βρήκαν. Όταν ήρθατε και με βρήκατε το βράδυ, σα ε, εξέφρασα την προθυμία μου να ακούσω τα προβλήματά σα και τι υποδείξει σα. Και προσπάθησα να κρατήσω το, το, το ουσιώδε από τι τροπολογίε τη ομάδα σα. Όσον αφορά το 64 και τις λιγότερο ρηπαίνουσες ε, ε, μορφές ενέργειας, νομίζω ότι είναι η πιο λογική λύση που καλύπτει και τις ανησυχίες σας. Γιατί εσείς στην τροπολογία σας, ε, στην 64, αναφέρεστε σε, ε, μεγα, σε μεγάλα υδροελεκτρικά έργα. Καταλαβαίνω τις ανησυχίες σας, αλλά ταυτόχρονα νομίζω ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μία γλώσσα και μία ορολογία που να είναι επαρκής. Γι' αυτό δεν, θεωρεί, ότι είναι σκόπιμο να Ε, Θεωρήσα ότι είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη διατύπωση χωρίς να κάνουμε απαραίτητα μία σύνδεση με την πυρηνική. Το θέμα τώρα ε, των, ε, αυτών των ε, των δολοφονιών και έχουμε την 82 που αναφέρεται στην καταπολέμηση αυτού του φαινομένου που αφορά την ακρογωνιά, τον ακρογωνιαίο λίθο των σχέσεών μας. Ναι, ναι. Λοιπόν, όσον αφορά τη βία κατά των γενικών ε, και τη δολοφονία των γυναικών ω ακραία έκφραση διακριτική μεταχείριση ενάντια στι γυναίκε, ότι αυτό αποτελεί ακρογωνιαίο λίθος στη σχέση μα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα. Είμαι διατεθειμένο να παραπέμψω στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τι ε, ε, ε γυναικοκτονίε. Αλλά το να πούμε τώρα ότι αυτό είναι ακρογωνιαίο λήθο, νομίζω ότι είναι υπερβολικό. Ε, γι' αυτό, αυτό που σα προτείνω ε, και το προτείνω και σε άλλε πολιτικέ ομάδε, είναι στα πλαίσια αυτή τη στρατηγική εταιρική σχέση, όπω αναφέρεστε και στο δεύτερο μέρο τη τροπολογία σα, ε, οι αρμόδιε ε, οργανώσει με την κατάλληλη πολιτική και οικονομική υποστήριξη να ασχοληθούν με το θέμα τη προστασία των γυναικών και τη μετώπιση του φαινομένου τη βία. Όσον αφορά αυτό το θέμα, αλλά και πολλά άλλα, πρέπει να αποφύγουμε ένα κάποιο πατερναλισμό. Κοιτάξτε, όταν μιλάμε για στρατηγικέ δαπάνε, έχετε δίκιο κύριε Μέγερ. Έτσι και εμεί θα πρέπει να επαγρυπνούμε και να κοιτάμε κοιτάμε τι γίνεται στον οίκο μα, ε, όπου πραγματικά οι στρατιωτικέ δαπάνε βεβαίω είναι περισσότερε από ό,τι στη Λατινική Αμερική. Αλλά κύριε Μέγερ, το, το μόνο που θέλησα και αυτή που υπέβαλε η τροπολογία είναι να χαμηλώσουμε κάπως τη θερμοκρασία και να ε, μην, να μην δημιουργήσουμε την εντύπωση ενός ε, πατερναλισμού. Όσον αφορά την κυρία Λούνατσεκ και την ε, σχετική παράγραφο, για τι συμφωνίε που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευση, περιορίστηκα στο να ακολουθήσω αποκλειστικά ε, την, ε, αυτό που ενέκρινε και στην ολομέλειά του το προηγούμενο, ε, στην προηγούμενη ολομέλειά του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε σχέση με την έκθεση Αλμπερτίν. Όπου δηλαδή σημειώνουμε ότι ε, ολοκληρώθηκαν σε τεχνικό επίπεδο, όμως, όπως μας εξέφρασε και η εκπρόσωπος της Επιτροπής, ε, τα θέματα αυτά των διαπραγματεύσεων και ότι παραμένουν ανοιχτά τα πολιτικά ζητήματα. Ήδη ενεκρίθη στο, ε, στο Κοινοβούλιο και υπήρξε ευρεία συνένεση στην τροπολογία όπως την πρότειναν οι σοσιαλιστές στην προηγούμενη ομολομέλεια. Γιατί τώρα να ξεφύγουμε από τη συνένεση αυτή και να ακολουθήσουμε άλλες, άλλες οδούς. Επίσης να σας πω, και στον κύριο Μέγερ απευθύνομαι, ότι όσον αφορά την αρνητική αξιολόγηση της συμφωνίας με την Κολομβία είναι κάτι το οποίο μας διαιρεί. Εμείς πιστεύουμε ότι η Κολομβία ωφελείται από το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων, από ένα σύστημα πολιτικού διαλόγου και συνεργασία και θεωρούμε ότι θα ε, οδηγούσαμε την πλειοψηφία ε, τη κοινωνία τη Κολομβία και του λαό τη Κολομβία σε τιμωρία, ακριβώ επειδή ε, βεβαίω υπάρχουν αυτά τα φρικτά εγκλήματα τα οποία όλοι τα καταδικάζουμε. Αλλά δεν μπορούμε να καταδικάσουμε ολόκληρο τον Κολομβιανό λαό. Κοιτάξτε, αυτή ε, για τη συμφωνία της ε, σύνδεσης ε, συμφωνούμε. Μακάρι να είχαμε συμφωνία σύνδεσης με το σύνολο των χωρών της κοινότητας των άντων. Δυστυχώς, όπως θύμισε και ο κύριος ε, Μέγερ, ε, υπάρχει μια χώρα ε, που, από την κοινότητα των άντων που δεν δέχεται ούτε στο Σύνταγμα ούτε στην πολιτική φιλοσοφία αυτές τις συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου που είναι τέταρτης γενιάς και που οδηγούν σε σταδιακή απελευθέρωση των σχέσεων, των εμπορικών σχέσεων. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να αναφερθώ στο θέμα αυτό και να πω ότι πραγματικά εμεί θα θέλαμε να έχει ολοκληρωθεί, να έχει συναυθεί συμφωνία ε, τέτοια φύση με όλε τι χώρε κοινότητα των Άνδεων. Όσον αφορά τον κύριο Αγκουράκη, ο οποίο μα μίλησε για αποστρατητικοποίηση. Ειλικρινά, διάβασα με πολύ μεγάλη προσοχή την 11, την παράγραφο 11 της έκθεσης και τι ζητάμε να υπάρξει ένας ε, χάρτης ε, ε, για την ασφάλεια με βάση τον καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ και τη συναφή διεθνή νομοθεσία να περιλαμβάνει κοινέ στρατηγικές και κατευθύνσεις πολιτικές δράσεις και ασφάλειες για την αντιμετώπιση των κοινών απειλών που σκιάζουν τους εταίρους της διπεριφερειακής στρατηγικής εταιρικής σχέσης. Με όλο το σεβασμό. Δεν βλέπω πουθενά τη στρατηγική διάσταση. Είναι μια έκθεση, όπως είπα και προηγουμένως, ήταν η η κυρία που δεν νομίζω ότι πρέπει να την υποψιάζεστε για στρατιωτικοποίηση των σχέσεων και για τέτοιε προσπάθειε. Και ειλικρινά πιστεύω ότι η διατύπωση αυτή είναι ιδιαίτερα λογική και δεν παρουσιάζει πρόβλημα. Όσον αφορά τα θέματα τη μετανάστευση, βεβαίω είναι ευαίσθητο το θέμα αυτό, το καταλαβαίνω. Είναι ένα θέμα ε, το οποίο πραγματικά ε, είναι αμφιλεγόμενο, ξέρετε όλοι, ότι η πράσινη βίβλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το θέμα αυτό αναφέρει στο ότι ε, είμαστε οι μόνοι που θα χάσουμε ενεργό πληθυσμό μέσα σε 30-35 χρόνια ε, με, με, με, ανισχυτικά στοιχεία ε, για τη γύραση του πληθυσμού, για το πώς θα είναι αν των 80, αν των 60 και θα πρέπει λοιπόν να καταβάλουμε όλη κάθε προσπάθεια για να βρούμε κάποιες λύσεις που θα μας επιτρέψουν να ξεπεράσουμε αυτά τα προβλήματα και αυτές τις ελλείψεις πάντα στο πλαίσιο του σεβασμού του νόμου. Ε, όσον αφορά την οδηγία για την επιστροφή ήταν ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο σημείο, αλλά σα υπενθυμίζω ότι το κοινοβούλιο μα ήταν το πρώτο που ξεκίνησε αυτό το προβληματισμό και το διάλογο για να, για να ακούσουμε και να εξηγήσουμε ποιοι είναι οι λόγοι για του οποίου ε, ε, ε, υπήρξαν οι κανόνε αυτοί. Σα υπενθυμίζω, ακρο, με τον κύριο Μπαρόν, τον αντιπρόεδρο τη Επιτροπή ε, και με την κυρία Φεραίρο που είχαν την ευκαιρία να μα εξηγήσουν ποιο ποια ήταν η αρχή που οδήγησε στην έμπνευση αυτών των κανόνων. Ε, κύριε Πρόεδρε, τελειώνω λέγοντα, όπω και είπα και στην αρχή, ότι αύριο θα ψηφίσουμε την έκθεση αυτή. Νομίζω ότι ε, οι περισσότερε πολιτικέ ομάδε καταβάλαμε ιδιαίτερα ε, σκληρή προσπάθεια για να ε, δούμε τις, και να αντιμετωπίσουμε τι ανησυχίε όλων, να δούμε πού συμφωνούμε και όχι πού διαφωνούμε. Και το μόνο που μπορώ να πω στην κυρία Νούνετσεκ είναι ότι ε, μέχρι την ψηφοφορία αύριο το πρωί στι 9 η ώρα εμεί στη διάθεσή τη για να δούμε πώ μπορούμε να ξεπεράσουμε τα εμπόδια, για να καταβάλουμε όλη κάθε προσπάθεια έτσι ώστε να συμπεριλάβουμε και τι δικέ σα απόψει, πάντα βεβαίω εφόσον είναι συνεπεί με τη βασική φιλοσοφία τη έκθεση και βεβαίω τονίζοντα ότι σε μια διαπραγμάτευση δεν υποχωρεί μόνο ο εισηγητή, αλλά υποχωρούν ο, λίγο και όλε οι πολιτικέ ομάδε. Σα ευχαριστώ όλου για τι προσπάθειέ σα και κατά ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την ευκαιρία που μου δώσατε και για τη ε, συμβολή όλους για αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον συνάδελφο Σαλαφράγκα. Σας θυμίζω ότι αύριο από τις 9 θα ψηφίσουμε με ηλεκτρονικό τρόπο. Σας καλώ όλους να έχετε μαζί σας την κάρτα ψηφοφορίας. Θα περάσουμε στο επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη τις λεγόμενες θεσμικές πλευρές της ε, προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Θα δώσω αμέσως το λόγο στον κύριο Πρέντα, τον εισηγητή, για να μας παρουσιάσει την γνωμοδότησή του και να μας περιγράψει επίσης και τις τροπολογίες τις οποίες έχει μέχρι τώρα λάβει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λίγα εισαγωγικά. Γνωρίζετε όλοι ότι σύμφωνα με το άρθρο 6.2 της Συνθήκης το θέμα της ένταξης της Ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης, αν θέλετε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στη Σύμβαση είναι σε φάση υλοποίησης όπως ακριβώς το περιγράφει το συγκεκριμένο άρθρο, η ε, ένταξη αυτή είναι και μία προτεραιότητα της Ισπανικής Προεδρίας στα πλαίσια της θέσης σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας. Από πλευράς ε, του Συμβουλίου της Ευρώπης, η ένταξη στο πρωτόκολλο 14 έχει σαν στόχο να διευκολύνει την ε, ένταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την άλλη είναι ευκταίο μια γρήγορη ένταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να γίνει πραγματικότητα, γιατί κάτι τέτοιο είμαι πεπισμένος θα βελτιώσει την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη και την αξιοπιστία της Ένωσης στη διεθνή σκηνή. Σχετικά τώρα με τους τρόπους ε, αυτής της ένταξης δεν έχουν ρυθμιστεί ακόμα. Τίθενται είναι αλήθεια ορισμένα προβλήματα γιατί στη συνθήκη Υπάρχουν κάποιες πρώτες ενδείξεις. Υπάρχει το άρθρο 218 το οποίο καθορίζει την διαδικασία. Υπάρχει επίσης και το πρωτόκολλο υπαρίθμ 8 όπως επίσης και τη δήλωση υπαρίθμ 2 που ορίζουν τις βασικές γραμμές οι οποίες πρέπει να γίνουν σεβαστές, αρμοδιότητες της Ένωσης, αρμοδιότητες των οργάνων, διατήρηση της θέσης την οποία έχουν από μόνα τους τα κράτη-μέλη, όπως επίσης και το μονοπόλιο του δικαστηρίου για τις διαφορές ανάμεσα στα κράτη-μέλη σχετικά με την ερμηνεία. Κάποια περίπλακα θεσμικά θέματα λοιπόν τίθενται. Τα θέματα αυτά έχουν αντιμετωπιστεί ήδη σε έκθεση του Κοινοβουλίου για την Επιτροπή ΑΦΚΟ. και κάποια από τα θέματα περιλαμβάνονται και στην δική μου γνωμοδότηση. Έχει ήδη γίνει μία πρώτη συζήτηση στις 22 Φεβρουαρίου αν θυμάμαι και υπάρχουν τρία θέματα στα οποία επιμένω. Καταρχάς το θέμα της εμβέλειας της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Ε, θα γίνει προσχώρηση μόνο στη σύμβαση ή και στα πρωτόκολλα τα συμπληρωματικά γιατί δεν έχουν επικυρώσει όλες οι χώρες το συμπληρωματικό πρωτόκολλο. Το δεύτερο είναι η εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στα όργανα ελέγχου. Καταρχάς θα πρέπει να ορίσουμε ένα δικαστή ε, στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που να εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Ένωση η κοινοβουλευτική συνέλευση όταν ορίζει τους συγκεκριμένους δικαστές δίνει τη δυνατότητα και στο Υπουργικό Συμβούλιο να ελέγχουν τη διαδικασία αυτή. Και θα πρέπει επίσης και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να διατηρηθεί θα έλεγα και πριν την προσχώρηση και μετά την προσχώρηση και θα πρέπει να διευκρινιστεί γενικά η συνεργασία και συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τώρα να σχολιάσω λίγο αν μου επιτρέπετε τις τροπολογίες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που κατέθεσαν τροπολογίες. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω αυτούς οι οποίοι δέχτηκαν τις συμβιβαστικές προτάσεις τις οποίες κάνω Σχετικά με την εμβέλεια της προσχώρησης, προτείνω κάποιες συμβιβαστικές προτάσεις οι οποίες αντικατοπτρίζουν τη γενικότερη συνένεση. Η προσχώρηση στη σύμβαση αυτή λέγεται στις συμβιβαστικές προτάσεις πρέπει να συμπληρωθεί και με την ένταξη σε άλλα θέματα, σε άλλους τομείς όπως το σύστημα του Στρασβούργου και στα συμπληρωματικά πρωτόκολλα. Θα πρέπει να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας με το Συμβούλιο της Ευρώπης, συμμετέχοντας στην Επιτροπή για την ε, πρόληψη των βασανιστήριων, σαν παράδειγμα. Παράλληλα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει κατά τη διάρκεια αυτή της διαδικασίας, ήδη από την πρώιμη φάση καθορισμού της εντολής μέχρι την πλήρη κατάληξη της συμφωνίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επαναλαμβάνω, θα πρέπει να εμπλέκεται πλήρως. Μια άλλη συμβιβαστική πρόταση είναι η επιβεβαίωση των αρχών σύμφωνα με τον οποίο θα πρέπει να διατηρηθεί πλήρως το δικαστικό σύστημα της σύμβασης αυτής το οποίο έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα θετικό και λειτουργικό. Και η ένταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα πρέπει να δημιουργήσει προβλήματα σε σχέση ιδιαίτερα με το βάρος, τον όγκο των εργασιών του δικαστηρίου και όπως σας είπα στην αρχή η τελευταία συμβιβαστική πρόταση αφορά τη χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Εδώ θα πρέπει να υπάρξει μια διατύπωση θετικότερη της αρχικής, υπογραμμίζοντας ότι είναι απαραίτητο ότι η χάρτα αυτή θα πρέπει να εφαρμόζεται πλήρως και με ενιαίο τρόπο σε επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από όλα τα κράτη-μέλη. Θα σταματήσω εδώ ευχαριστώντας όλους τους συναδέλφους οι οποίοι με βοήθησαν και κατέθεσαν τροπολογίες και δέχτηκαν μερικές φορές τις συμβιβαστικές τροπολογίες. Ευχαριστώ κύριε Πρέντα. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, Ατόντο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Προφανώς θα προσπαθήσω να σχολιάσω κι εγώ τις τροπολογίες τις οποίες συζητάτε. Βεβαίως, ε, στην ε, Επιτροπή μας δεν θα αποφασίσω εγώ ποια θα πρέπει να είναι η άποψη. Βεβαίως, η έκθεση της ΑΦΕΤ θα αποτελέσει τμήμα του κεκτημένου και του συνόλου των εγγράφων, τα οποία την κατάλληλη στιγμή θα υποβληθούν στην Ολομέλεια. Τώρα, τούτου λεχθέντος και με όλο το σεβασμό, θα ήθελα να σας δώσω την άποψή μου για αυτό το που θα αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης ε, από εσάς. για τις τροπολογίες στο έγγραφο της Άφετος όσον αφορά την έκθεση αυτή. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομο. Τονίζω, με όλο το σεβασμό. Για παράδειγμα, επανειλημμένα, σας λέω, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι πολλές φορές οι τροπολογίες έχουν ως στόχο να τελειοποιήσουν, να ολοκληρώσουν ένα έγγραφο της ΑΦΕΤ που συμπεριλαμβάνει, που συμπεριλαμβάνουν ιδέες που ήδη βρίσκονται στη βασική έκθεση. Αυτό ισχύει όσον αφορά, για παράδειγμα, την πρώτη τροπολογία, που κατά την άποψή μου πάλι δεν ε, ε, φέρνει κάτι το καινούριο, ούτε κάποια σημαντική ιδέα. Και αυτά τα οποία προτείνεται, προτείνει είναι στην καλύτερη περίπτωση ε, πράγματα που αναφέρονται και στην βασική έκθεση. Δεν συμβαίνει το ίδιο και με την τροπολογία 2 της κυρίας Γιαννάκου που ε, ακριβώς εδώ η, η, η σκιώδης εισηγήτρια ε, στην τροπολογία 2 ε, νομίζω ότι ε, τα, θέτει τα πράγματα πολύ σωστά. Δεν θα κρίνω τώρα τις συμβαστικές τροπολογίες που μας μοίρασε ο κύριος Πρέντα γιατί δεν μπόρεσα να τις κρίνω. Αλλά θα σχολιάσω τις τροπολογίες μία-μία. Λοιπόν, όσον αφορά την τρία της κυρίας Χαουτάλα και της Μπάρμπαρα Λόχμπιλερ, εδώ έχουν το πρόβλημα το εξής ότι αναφέρονται σε μία εντολή που νομίζω δεν είναι σωστό να θεσπιστεί. Γιατί αναφέρεται. Αναφέρει ότι η προσχώρηση θα πρέπει να γίνει χωρίς να αλλάξει τίποτα. Εντάξει, στη σύμβαση. Είναι προφανές ότι η σύμβαση, όσον αφορά το ουσιώδες του τμήμα, θα παραμείνει αυτή που είναι. Γιατί εμείς είμαστε που προσχωρούμε στη σύμβαση. Αλλά ορισμένε πτυχές που αποτελούν μέρος ε, του κεκτημένου της σύμβασης θα αλλάξουν. Για παράδειγμα, η οικονομική συνεισφορά στη σύμβαση. Να, ε, ε, δευτερεύουσε πτυχέ. Αλλά γιατί εδώ να πούμε δεν θα αλλάξει τίποτα και να δώσουμε αυτή την εντολή. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό και, και σόφρον. Στην τέσσερα. Εδώ και δυστυχώς, το λέω από προσωπική άποψη, δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε αυτό το οποίο αναφέρει. Γιατί είναι σαφέ ότι η προσχώρηση στη Σύμβαση, η προσχώρηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, έχει να κάνει με, με ένα δρόμο που μπορεί να έχει να κάνει και με την ένταξη στην κοινωνική χάρτα, αλλά έχουμε και το, χάρτα, και το, και το χάρτη του, του, Τωρίνο. Που δυστυχώ, το ξαναλέω, δεν είναι αποδεκτή ε, συνολικά από, το νομικό, από την νομοθεσία των κρατών μελών και δεν μπορούμε να συνδέουμε άμεσα την προσχώρηση στη σύμβαση με, την, ε, με το χάρτη, τον κοινωνικό χάρτη. Δυστυχώς. Το λέμε πιο σαφώ στην έκθεση Τσάφκο, ότι στο 13, που στο 13, στη 13 παράγραφο αναφέρεται ο προβληματισμό αυτό σε σχέση με, με την κοινωνική χάρτα, δεδομένη προσχώρηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Από την άλλη, όσον αφορά αυτό το οποίο αναφέρεται, ότι η, πρόσβαση, ότι η προσχώρηση πρέπει να γίνει σε όλα τα πρωτόκολλα. Α, εδώ προσοχή, γιατί η εντολή ε, του, της, του Ευρωπαϊκού Συντάγματος δεν μας επιτρέπει να αλλάξουμε αυτό που θα ονομάζαμε status quo κάθε χώρα απέναντι στη σύμβαση. Δηλαδή, να το πω διαφορετικά, να το πω διαφορετικά. Οι 27 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν μέρος της σύμβασης, βεβαίως. Αλλά οι 27 δεν έχουν προσυπογράψει όλοι τα πρωτόκολλα, τα οποία μεταγενέστερα αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασία με βάση τη σύμβαση. Η συνθήκη τη Λισαβόνα τι μα λέει, ότι η προσχώρηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να αλλάξει το status quo σε κάθε χώρα. Άρα πρέπει να δούμε τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπραγματεύεται με τη σύμβαση και σε ποια πρωτόκολλα προσχωρά το σύνολο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούμε αυτή τη να δώσουμε εντολή ότι μια εντολή που να αλλάζει τα πράγματα και το status quo, και τότε παραβιάζουμε μια συνθήκη, την αρχή τη συνθήκη Λισαβόνα, συγγνώμη, που αναφέρεται ότι θα πρέπει να σεβαστούμε τι αρμοδιότητε, ε, τι εξουσίε και την ουδετερότητα των χωρών. Αυτό δυστυχώ δεν μπορούμε να το αλλάξουμε και δεν μπορούμε να το κάνουμε με μια εντολή όπω αυτή που αναφέρεται εδώ. Πέντε τώρα, τροπολογία 5. Εγώ νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να δούμε συνδυασμό με την 22. Και είδα, και είδω ότι ο κύριος Πρέντα εργάζεται προς την κατεύθυνση αυτή. Να δούμε, να δούμε. Για να ξεκαθαρίσω κάπως τα πράγματα. Ε, η κυρία Μεργιάτ μας προτείνει το εξή. Ε, εντασσόμενη η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Σύμβαση εντάσσεται ταυτόχρονα και σε μία σειρά από οργανισμούς που απορρέουν από τη σύμβαση. Αλλά κοιτάξτε, προσοχή. Η σύμβαση έχει τρεις βασικού οργανισμούς. Την Υπουργική Επιτροπή που ασχολείται με την εκτέλεση των αποφάσεων, το Δικαστήριο του Στρασβούργου και την ε, Κοινοβουλευτική Συνέλευση. Μετά υπάρχει μια Επιτροπή για τα Βασανιστήρια, μια Επιτροπή για τη Μετανάστευση ε, κτλ. Αλλά κοιτάξτε, δεν είναι σαφές ότι όλες οι χώρες ανήκουν σε αυτούς τους οργανισμούς. Ούτε είναι σαφές ότι μπορούμε να υποχρεώσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να ενταχθεί σε όλους αυτούς τους οργανισμούς. Και κάτι άλλο. Και νομίζω ότι αυτό ε, είναι και η σύσταση της ΑΦΕΤ. Να συμπεριλάβουμε στη βασική έκθεση της ΑΦΚΟ την δυνατότητα αυτή οι διαπραγματεύσει να εξετάσουν τη δυνατότητα ένταξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση στου τρει βασικού οργανισμού, σε τρία βασικά όργανα και ίσω και σε άλλα. Και θα δούμε. Αλλά να μην θέσουμε τόσο σαφή εντολή και άκαμπτη για ένταξη σε, σε μία σειρά επιτροπών που από την άλλη, προσοχή, δεν είναι και ε, οργανισμοί του Συμβουλίου της Ευρώπης. Τώρα, στην επόμενη. Next. Και εδώ το ίδιο. Εκφράζουμε τη λύπη μας για το ότι έχουν επιφυλάξει το Ηνωμένο Βασίλειο ε, η Πολωνία και η Δημοκρατία της Τσεχίας που δεν προσυπόγραψαν το χάρτη. Αλλά αυτό πρέπει να γραφτεί σε μια έκθεση προσχώρηση για την προσχώρηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τι να πω. Από την άλλη, δεν είναι σωστό αυτό το στο τέλο αυτή τη ολομέλεια που αναφέρεται ε, στην ύπαρξη τριών εξαιρέσεων αποδυναμώνει τη θέση προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως Ένωσης. Α, προσοχή. Το ότι οι τρεις αυτές χώρες δεν προσυπέγραψαν το χάρτη δεν σημαίνει ότι στις χώρες αυτές δεν είναι απαιτητή ε, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μα είναι. Διότι αυτές οι τρεις ε, χώρες ε, είναι μέρος της σύμβασης. Γιατί λοιπόν τις αναφέρουμε ως εξαίρεση από την εφαρμογή της σύμβασης, δεν το καταλαβαίνω, δεν είναι σωστό. Και από την άλλη να σας πω και το εξή. Όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση στις πράξεις της ε, ε, ε, ε, χρησιμοποιεί το δίκαιο το οποίο προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπόκειται και στη σύμβαση και στο χάρτη, πέραν του γεγονότος ότι τρεις χώρες δεν έχουν προσπρογράψει το χάρτη. Όταν μιλάμε για την Ένωση, δηλαδή για τα κοινοτικά όργανα και για το κοινοτικό δίκαιο, τότε αυτό το κοινοτικό δίκαιο υπόκειται στο χάρτη. Ανεξάρτητα με το ότι οι τρει χώρε δεν έχουν προσπογράψει το συγκεκριμένο έγγραφο. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί εδώ υπάρχει μια κάποια νομική ασάφεια. Νομίζω λοιπόν ότι η τροπολογία προκαλεί σύγχυση και τίποτα άλλο. Συμφωνώ ιδιαίτερα με την τροπολογία του κυρίου Τοκέ και τη κυρία Μπερτζίατ στις ε, 7 ε, και 8. Νομίζω ότι είναι δύο ε, τροπολογίες που θα μπορούσαμε κάλλιστα να συμπεριλάβουμε. Γιατί πραγματικά εδώ αναφέρουν την πολιτική αρχή του. Τι σημαίνει δηλαδή η ένταξη. Ιδίω όσον αφορά τι τρίτε χώρε, τι λεγόμενε τρίτε χώρε. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και πολλά χρόνια με τις ε, υπόλοιπες 20 ε, χώρες ε, που συνδέονται με την Ένωση. Δεν ξέρω, μακρυγορό πρόεδρε, να τελειώσω έτσι. Ωραία, τελειώνω. Ήθελα να πω λοιπόν ότι όσον αφορά τις τροπολογίες 7 και 8 είναι πολύ σημαντικές γιατί σχολιάζουν και αναφέρονται στην σημασία που έχει η ενίσχυση της αξιοπιστίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι των χωρών που ενώ δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνδέονται στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Σύμβασης. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό να συμπεριλάβουμε την εννέα. Το είπαμε και προηγουμένως. Δεν, ανήκουν σε, δεν έχουν προσπογράψει όλα τα πρωτόκολλα όλες οι χώρες. Όσον αφορά τώρα την τροπολογία 10. Νομίζω ότι δεν είναι ορθή αυτή η δήλωση του ότι από την ένταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη συνέχεια νομικά δεσμεύεται. Α, κοίταξε με, με το χάρτη ήδη δεσμευόταν. Μην ξεχνάμε ότι ο χάρτη ενεκρίθη στο Μάστριχ και στην, και πριν από πολλά χρόνια. Και ενώ η συνθήκη Λισαβόνα, της Λισαβόνα αναφέρεται ε, με δεσμευτικό τρόπο στις πράξεις, στην πρώτη παράγραφο του 6, ε, αυτό δεν σημαίνει ότι ο χάρτη δεν αποτελούσε ήδη πηγή έμπνευση για το κοινοτικό δίκαιο. Αντίθετα, μεγάλο μέρο τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του Λουξεμβούργου ε, προέρχεται ακριβώ από την εφαρμογή του χάρτη, που αποτελεί το βασικό προσανατολισμό για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τι θεμελιώδει ελευθερίε που θεσπίζονται από το χάρτη που όπω σα είπα ενεκρίθη στην οίκια πριν από 10 χρόνια. Κατανοώ βεβαίω ότι μπορεί να υπάρξει μια λύση σε σχετικά με την 11. Ίσως συνδυασμού με την 23. Σε σχέση με τις πράξεις που αφορούν τις εξωτερικές σχέσεις. Α, τελειώνω, τελειώνω, ναι, ναι εντάξει. Η 12 δεν έχει κανένα πρόβλημα και η 13 θα τη συνδυάσουμε με την 21. Νομίζω ότι ο κύριος Πρέντα ήδη το, το πράττει. Τελειώνω, τελειώνω γιατί ο πρόεδρος μου λέει ότι μακρηγόρησα και το φοβόμουν αυτό. Σας λέω λοιπόν το εξή. Δεν συμφωνούμε με το 14, ούτε με το 15, ούτε με το 16. Δυστυχώς δεν μπορώ να συμφωνήσω με τις τροπολογίε αυτές, ούτε με το 17. Ε, αν και ναι, ναι, θα μπορούσαμε να δεχτούμε το πρώτο τμήμα, όχι το δεύτερο. Συμφωνούμε με το 18 και με το 19 και με την 20 και με την 21. Τη κυρία Γιαννάκου Μεργία και του κύριου Πρέντα και στην 22 να ε, τη συνδυάσουμε με αυτό που σας είπα προηγουμένως για την δυνατότητα η εντολή να λάβει υπόψη τη δυνατότητα ένταξη σε ορισμένους οργανισμούς ε, στα πλαίσια του Συμβουλίου της Ευρώπης. Και για την 23 θα εξετάσουμε την ε, ε, εξέβρεση μια πιθανή λύση σε συνδυασμό με μια άλλη που σα είπα και προηγουμένω, που είχε παρόμοιο περιεχόμενο. Λυπάμαι, τα πάω πολύ γρήγορα τώρα. Ε, αυτή είναι η άποψή μου. Πρόεδρε, αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ, αλλά δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Είχε πολύ ενδιαφέρον αυτό που μα είπατε παρόλα αυτά. Η κυρία Γκάλ έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε θα είμαι σύντομη. Εγώ είμαι η συντάκτης της ε, γνωμοδότησης στον ε, φάκελο αυτόν ε, που αφορά την ενισχυμένη συνεργασία με την Επιτροπή Ελευθεριών. Θα οφείλω να συγχαρώ τον εισηγητή γιατί δεν είναι κάτι το εύκολο, το γνωρίζω και από η δική μου τη δουλειά το να αποφύγει κανείς να αγγίξει ζητήματα που θεωρούνται αρμοδιότητα της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων ή εδώ πέρα της Επιτροπής Ελευθεριών. Είναι αναπόφευκτο τα ζητήματα αυτά να ανακύπτουν συνεχώς και δεν μπορεί να διαχωρίσει κανείς αυστηρά τις αρμοδιότητες και είναι σημαντικό αυτό το οποίο έκανε ο κύριος ε, Πρέντα και συμφωνώ με τις ε, τροπολογίες του γιατί νομίζω πως ένα από τα βασικά θέματα της ε, ένταξης προσχώρησης Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να δημιουργηθεί μια πανευρωπαϊκή ζώνη ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να ενισχυθούν οι σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ευρύτερης Ευρώπης και θα υπάρξει μια δυναμική στα ανθρώπινα δικαιώματα ευρύτερα στην Ευρώπη. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το οποίο προτείνεται από την Επιτροπή, μας και πράγματι είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η προσχώρηση αλλά βεβαίως τα υπόλοιπα θα τα πω αύριο στην Επιτροπή Ελευθεριών. Ευχαριστώ. Η κυρία Ουτάλ, πρόεδρος Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Πρέντα για το εξαιρετικό έργο του. για να συζητήσουμε αυτή την έκθεση θα ήθελα εγώ τώρα να πω το εξής. Η Επιτροπή μας μπορεί να θίξει πολιτικές ε, προοπτικές ε, που ανοίγει αυτή η προσχώρηση στην ε, Σύμβαση και βεβαίως η Επιτροπή συνταγματικών θεμάτων δικαίως είδε την νομική πτυχή, αλλά νομίζω πως ο συγητής εδώ είναι πολύ αυστηρός, γιατί προφανώς δεν αντιλαμβανόμαστε ακόμα όλες τις ε, συνέπειες της ε, προσχώρησης και αυτό το οποίο είδε ο κύριος Πρέντα και εγώ και η κυρία Λοχμπίλερ είναι να δούμε περαιτέρω σημεία που θα άνοιγαν λίγο το να δούμε το τι αντίκτυπο θα έχει αυτή η συνθήκη στην εξωτερική δράση και τις ε, διεθνείς σχέσεις ε, της Ένωσης και λυπούμε λίγο για το ότι ο εισηγητής δεν έκανε δεκτές τροπολογίες 11 και 12 που τονίζουν πως σύμφωνα με το άρθρο 1 της Ένωσης οποιοδήποτε άρθρο μπαίνει εντός της ε, επικράτειας της δικαιοδοσίας της Ένωσης θα μπορεί να επικαλεστεί την ε, σύμβαση. Δεν ξέρω, θέλω να μας το διευκρινίσει αυτό η Κομισιόν. Δεν ξέρω εάν η συνθήκη, η σύμβαση ισχύει μόνο για επικόους της Ένωσης. Και είναι κάτι το ενδιαφέρον εδώ πέρα, αυτό που λέμε στις τροπολογίες 11 και 12 πώς. Η προσχώρηση της Ένωσης ισχύει και για οποιοδήποτε άτομο που υπόκειται στην δικαιοδοσία της Ένωσης και εκτός της επικράτειάς της π.χ. αντιπροσωπείας της Ένωσης. Θα ήθελα να γνωρίζω αν την Κομισιόν αν ισχύει αυτό ή όχι και αν ισχύει δεν νομίζω πως η Επιτροπή Εξωτερικών δεν θα πρέπει να κάνει τέτοιες δηλώσεις. Οπότε εγώ είμαι υπέρ των τροπολογιών 11 και 12. Τώρα ο εισηγητής της Επιτροπής Συνταγματικών Θεμάτων φαίνεται πως είναι κάπως επιφυλακτικός για την τροπολογία 8 που αφορά την εμπιστοσύνη των πολιτών στην επία της προσχώρησης. Θα ήθελα να επισημάνω πως η δική μας τροπολογία 10 πηγαίνει προς την ίδια κατεύθυνση. Είτε λοιπόν η 8 είτε η 10 αναφέρουν αυτή την ιδέα ότι η προσχώρηση δηλαδή στην σύμβαση είναι πάρα πολύ σημαντική για την αξιοπιστία και της Ένωσης ε, και της ε, εξωτερικής πολιτικής της. Ε, λυπούμε που δεν έγιναν κατανοητές αυτές οι τροπολογίες γιατί όπως ξέρετε η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει τρίτες χώρες όλο και περισσότερο όσον αφορά τον διάλογο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίες μας λένε δείτε πρώτα τα, δικά σας και μετά έλατε να μας κάνετε κήρυγμα. Οπότε νομίζω πως έχουμε εδώ πέρα μια προσθέμενη αξία της προσχώρησης στην σύμβαση και δεν νομίζω πως τίποτα πρέπει να μας να το πούμε. Είτε θέμε να επισημάνουμε τα δύο μέτρα και δύο σταθμά, είτε ε, να μιλήσουμε για την αξιοπιστία της Ένωσης. Πρέπει να αναφερθεί τέλος. Κατάλαβα πως ο εισηγητής της Επιτροπής Θεμάτων είναι κατά του να κάνουμε πολύ έντονες δηλώσεις για τυχόν άλλες προσχωρήσεις για την κοινωνική χάρτα, για την Επιτροπή πρόληψη των βασανιστήριων και καταπολέμησης του ρατσισμού και της μη ανεκτικότητα. Ε, με συγχωρείτε, αλλά μπορεί να κάνει μια πολιτική δήλωση η Ευρωπαϊκή Ένωση πως ε, θα είναι χρήσιμο τα κράτη-μέλη να αναγνωρίσουν αυτά τα πρωτόκολλα και να διευκολύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ μπορώ να πω πως ε, η πρόληψη των βασανιστήριων είναι απόλυτη προτεραιότητα και αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να συνεργαστούμε με το Συμβούλιο τη Ευρώπη με τον ΟΗΕ. Νομίζω λοιπόν πως η προσχώρηση θα είναι πάρα πολύ χρήσιμη για να αυξήσουμε και να ενισχύσουμε την διεθνή δικαιοσύνη σε συνεργασία με τους σημαντικούς αυτούς διεθνείς παίκτες τέλος ε, ο έχει είχε ένα πρόβλημα με την τροπολογία 3 που μιλάει για τα χαρακτηριστικά της σύμβασης αυτής κατά τη στιγμή της ε, προσχώρησης. Ε, νομίζω πως η σύμβαση αυτή είναι ένας θησαυρό αν θέλετε και αν είναι να προτείνουμε αλλαγές και αν να προτείνουμε αλλαγές χάνουμε το, το νόημα και νομίζω επίσης πως ξέρω πως η συγητής εδώ πέρα της Επιτροπής Δραματικών Θεμάτων μιλάει για ένα νέο δικαστικό φορέα για να δει τις διαφωνίες μεταξύ του Δικαστηρίου του Στρασβούργου και του Λουξεμβούργου, εγώ δεν είμαι πολύ υπεπισμένη. Γι' αυτό λέμε εδώ πέρα πως αλλαγές στο δικαστικό σύστημα της ΣΥΜΑΣ πρέπει να παραμείνουν ελάχιστες. Αυτά. Και χαίρομαι για το ότι οι εισηγητές Επιτροπής Νομικών και εξωτερικών δέχτηκαν πολλές από τις τροπολογίες μας. Ευχαριστώ. Τελευταία παρέμβαση κύριε Γεννακού. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, η έκθεση του κυρίου Πρέντα από πλευράς ε, Επιτροπής ε, Εξωτερικών Υποθέσεων πραγματικά καλύπτει το ζήτημα που αφορά στους υπηκόους τρίτων χωρών και στο πώς θα αντιμετωπιστεί στο εσωτερικό της Ένωσης η τυχόν προσφυγή Απ' την άλλη πλευρά γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και νομίζω το μνημόνευσε και ο κύριος ο εισηγητής ότι η σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες με βάση τα, ε, τις αποφάσεις και το δεδικασμένο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του Στρασβούργου στην ουσία έχουν ευρύτερη ισχύ και δικαιοδοσία από ό,τι έχει ο χάρτης ε, των θεμελιωδών δικαιωμάτων που προσαρτήσαμε στη συνθήκη της Λισαβόνας. Έτσι λοιπόν έχει και λογική η προσχώρηση της Ένωσης, της ίδιας, στη σύμβαση ε, του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ε, όχι διότι η σύμβαση αυτή καθ' αυτή ως κείμενο είναι ευρύτερη, αλλά γιατί οι δικαστικές αποφάσεις που έχουν εν συνεχεία εκδοθεί από το Στρασβούργο πραγματικά δημιουργούν ένα ευρύτερο πλαίσιο προστασίας. Στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων βεβαίω έχουμε συζητήσει αρκετά. Θα γίνει και μία ακρόαση με προσωπικότητες που θα δώσουν τις ανάλογες κατευθύνσεις. Έχει ενδιαφέρον βέβαια να δούμε με τα πρωτόκολλα τι θα γίνει αν η προσχώρηση συνιστά και προσχώρηση στα πρωτόκολλα, αλλά κύριε Πρόεδρε είναι μια περίπλοκη υπόθεση, δεν είναι απλή. Έχει όμως ιδιαίτερη αξία, διότι με τη συνθήκη της Λισαβόνας η Ένωση αποκτά ενιαία και ιδία νομική προσωπικότητα. Και με την έννοια αυτή η προσχώρηση στη Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών και η υπαγωγή κατά κάποιο τρόπο στο Δικαστήριο του Στρασβούργου θα προσφέρει πολύ μεγάλες δυνατότητες στους πολίτες της Ευρώπης αλλά και στα κράτη-μέλη, ε, στην ίδια την Ένωση για να τροποποιήσει ε, πολύ συγκεκριμένα πράγματα και σε πολιτικό επίπεδο και σε ουσιαστικό ε, και νομίζω πως όλοι πρέπει να συμβάλλουμε στην προσπάθεια αυτή η οποία γίνεται τώρα για τον χάρτη των κοινωνικών δικαιωμάτων κλπ. Είναι ζητήματα τα οποία μπορούμε να κουβεντιάσουμε και θα συζητήσουμε στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Πάντως, η υπόθεση αυτή είναι αρκετά περίπλοκη, όχι μόνο στο επίπεδο της εκπροσώπησής μας στο Συμβούλιο της Ευρώπης, δηλαδή στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ε, ή στο Συμβούλιο Υπουργών κτλ., ε, αλλά κυρίως στην γνωμοδοτική δυνατότητα ε, που ανοίγεται για τα ίδια τα κράτη-μέλη και τους πολίτες της Ευρώπης θα είμαστε περισσότερο σίγουροι νομίζω να δώσουμε την τελική μας θέση και να συνεννοηθούμε μέσω του συντονισμού που μπορεί να κάνει ο εισηγητής μας αφού γίνει η ακρόαση στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων και ακούσουμε διακεκριμένους νομικούς και τη δική τους προσέγγιση ώστε να μην γίνουν λάθη στην τελική απόφαση του Κοινοβουλίου και να έχει η απόφαση αυτή την ευρύτητα που χρειάζεται. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχουν άλλοι δύο ζητήσει το λόγο. Γκέρζεμπ και η κυρία Βερζά. Παρακαλώ να είστε πολύ συνοπτικοί. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή της ε, γνωμοδότησης και να πω βεβαίως πως ε, αυτή είναι μία από τις συνέπειες του ότι η Ένωση απέκτησε νομική προσωπικότητα με την Λισαβόνα, οπότε μπορεί τώρα να προσχωρήσει στην ε, σύμβαση, η οποία όπως ξέρετε υπάρχει εδώ και δεκαετίες και μέχρι στιγμής η Ένωση δεν είχε προσχωρήσει σε αυτή την ε, σύμβαση. Οπότε μιλάμε για την ε, νομολογία του δικαστηρίου, μεν, αλλά βεβαίως δεν ίσχυε άμεσα. Τα κράτη-μέλη ήταν συμβαλόμενα μέρη οπωσδήποτε η δε Πολωνία πολύ πριν γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει εξοικειωθεί με την συνθήκη και τα πρωτόκολλα που ακολούθησαν. Θα ήθελα τώρα να ευσύρω την προσοχή σας στην παράγραφο 3 της Επιτροπής Δημοτικών Θεμάτων που λέει πως η προσχώρηση δεν αλλάζει την κατάσταση όσον αφορά το καθεστώς των κρατών μελών που έχουν ήδη ενταχθεί στην ε, συνθήκη. Νομίζω πως αυτό αναφέρεται στην τροπολογία 5 όπου μιλάμε για τα τρία κράτη-μέλη που έχουν διαφορετική στάση όσον αφορά τη χάρτα θεμελιωδών ε, δικαιωμάτων και ήθελα να περάσει στη κύριο μέρος τη συνθήκη της ε, Λισαβόνας. Και μπορεί να πει κανείς πως ε, το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καθίσταται συμβαλόμενο μέρος δεν αλλάζει τίποτα ως ε, προς αυτό. Η συμβαστική λύση η οποία προτείνεται εδώ, η συμβαστική τοπολογία 5 και παράγραφος 5, με συγχωρείτε, τροπολογία 6, είναι πολύ ε, καλύτερη. Δεν είναι μόνο θέμα ορολογίας, πρέπει να δούμε και το εάν ε, οι προτάσεις αυτές έχουν μια κοινή λογική. Αν δούμε παραδείγματο χάρη το ενδεχόμενο του opt-out της ε, αυτοεξαίρεσης. Δεν είναι επιθυμητό κάτι τέτοιο και δεν ε, είναι και ιδιαίτερα θετικό για την αξιοπιστία της Ένωσης εάν έχουμε κράτη-μέλη Τέλο πάντων, τόσο άλλο, τα κράτη-μέλη έχουν όλα προσφογράψει την, ε, τη σύμβαση. Τέλος, νομίζω πως όλοι ξέρουμε όσοι έχουν εμπειρία της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Συμβουλίου της Ευρώπης ξέρουν πως υπάρχουν κάποια προβλήματα όταν μιλάμε για το έργο του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων γιατί υπάρχουν ε, αμφισβητήσεις ε, και διαφωνίες και αν τηρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση την ε, σύμβαση τότε θα μπορέσουμε να επιλύσουμε τις συγκρούσεις αυτές και ελπίζω η ένταξη ενός ε, ακόμα μέλους να μην ενισχύσει τις ε, δυσκολίες αυτές στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου. Πρέπει να, να δούμε τα, τα ζητήματα αυτά, προσπαθήσουμε να τα επιλύσουμε ε, έτσι ώστε να μην γίνει μια δύσκολη κατάσταση ακόμη δυσκολότερη. Ναι, νομίζω κανείς να το θέλει αυτό. Ευχαριστώ. Κύριε Βεωσά, θα είμαι πολύ σύντομη. Η γνωμοδότηση αυτή έχει πολύ μεγάλη σημασία. Εν πολλής ολοκληρώνει αν θέλετε ή μάλλον προσπαθεί να συμπληρώσει και να φέρει πέρας μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό. μπορούμε να καταλήξουμε νομίζω σε μια συνένεση η οποία έχει ευρία βάση και οι συμβιβαστικέ προτάσεις τις οποίες έκανε ανταποκρίνονται πολύ στις ανησυχίες του εισηγητή της ΑΦΚΟ. Ίσως κάποια θέματα που άπτονται των δικών μου τροπολογιών τα γενίκευσε κάπως θα έλεγα, καθιστώντας τα όμως παράλληλα νομικά βιώσιμα και, πιο ευκολότερα, και ευκολότερα αποδεκτά. Έχω δύο ανησυχίες όμως δεν αφορούν τα σημεία στα οποία κατέθεσα τροπολογίες, αλλά σχετικά με τις συμβιβαστικές προτάσεις 1 και 5. Για την 1. Δύσκολα κατανοεί κανείς την έκφραση η οποία λέει θα πρέπει να ενοχληθεί το λιγότερο δυνατόν το σύστημα. Νομίζω ότι η έκφραση αυτή δεν είναι πολύ σωστή. Είναι πολύ προτιμότερο να πούμε να γίνουν οι ελάχιστες δυνατές τροποποιήσεις. Είναι προτιμότερο οι ελάχιστες δυνατές τροποποιήσεις του συστήματος για το 5. Και εγώ διαρωτώ με τι ακριβώς πρέπει να γίνει με τις εξαιρέσεις, τις ειδικέ εξαιρέσεις για την χάρτα. Αλλά δεν θα συμφωνήσω απόλυτα με τις προτάσεις τις οποίες κάνει ο κύριος Πρέντα Καλώς, ευχαριστώ. Πάρα πολύ σύντομα, κύριο Τόντο, για να ακούσουμε τον εισηγητή και να κλείσουμε. Θα ήθελα να πω ότι σέβομαι απολύτως την πρόταση την οποία κάνει η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων Ίσως εγώ να ήμουν περισσότερο συγκεκριμένος από όσο θα έπρεπε. Εσείς είσαστε αυτοί που θα πάρετε αποφάσεις. Κάποιες όμως από τις τροπολογίες οι οποίες έχουν κατατεθεί έγιναν δεκτές και το λέω αυτό και την κυρία Χάουταλα. Η τροπολογία 11 επίσης είναι μια τροπολογία η οποία θα πρέπει να ουσιαστικά να ενοποιηθεί με την αριθμόν 23. Υπάρχει και η 22 που αφορά τους οργανισμούς και τις επιτροπές τις οποίες θα συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ λογικό το να γίνεται συγκεκριμένη πρόταση για τη συμπερίληψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους οργανισμούς αυτούς. Το θέμα είναι να προσπαθήσουμε να διευκρινίσουμε ποιοι είναι αυτοί οι οργανισμοί, ποιος είναι ο κατάλογος αυτός των οργανισμών. Υπάρχουν, εν πάση περιπτώσει, κάποια επιπλέον σημεία στα οποία θα πρέπει να σταθούμε. Υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες οι οποίες θα πρέπει να αλλάξουν γιατί σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να θεωρηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια της συμμετοχής της σε αυτή την σύμβαση σαν ένα επιπλέον κράτος. Οι συζητήσεις που προηγήθηκαν ήταν πολύ ενδιαφέρουσες. Λίγα λόγια μόνο να μου επιτρέψετε να κάνω σχολιάζοντας την τροπολογία 3 και στρέφομαι στον εισηγητή της Επιτροπής ΑΦΚΟ. Η συμβιβαστική πρόταση την οποία εμείς προτείνουμε επί τη βάση της τροπολογίας 3 και της δικής μου τροπολογίας 7 περιλαμβάνεται έτσι και αλλιώς στην παράγραφο 9 της έκθεσής σας. Αυτός είναι ο στόχος μου. Να προσπαθήσει να γίνει ε, ε, συμβατό το κείμενο με το κείμενο 9 της δικής σας εκθέσεως. Σχετικά με την ε, τροπολογία 6 για την οποία μίλησε ο κύριος Γκρίσμπ. Τον ευχαριστώ που δέχθηκε τη συμβιβαστική πρόταση υπαριθμών 5 που είναι η μοναδική μορφή με την οποία μπορεί να περάσει το συγκεκριμένο κείμενο. Τελειώνω λέγοντας ότι αυτό το οποίο είπε η κυρία Ουτάλα έχει πολύ μεγάλη σημασία βέβαια. Νομίζω όμως ότι θα πρέπει να μην προκαταλάβουμε το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων. Και δεν θα πρέπει να προκαθορίσουμε τους τομείς αρμοδιοτήτων σε αυτή τη φάση. Το δικαστήριο είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να προχωρήσει σε τέτοιου είδους ρυθμίσεις και δεν θα πρέπει εμείς όπως είπα να προκαταλάβουμε οτιδήποτε όπως είπε ο Κίνγκα Γκάλ, όπως είπε η Κίνγκα το νόημα της συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το να έρθει η Ευρωπαϊκή Ένωση πιο κοντά στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό είναι ο πολιτικός στόχος. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο, με ηλεκτρονικό τρόπο. Πρέπει να έχετε τις κάρτες μαζί σας. Περνάμε στην επόμενη έκθεση. για την παρακολούθηση των βουλευτικών εκλογών στο Τατζικιστάν δίνει το λόγο στην κυρία Γέγκελ αμέσω. Δεν έχουμε χρόνο πολύ στη διάθεσή μας δυστυχώς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. 20, από 26 Φεβρουαρίου μέχρι 1η Μαρτίου είχα την τιμή να πάω με μία αποστολή πολλών συναδέλφων στο Τατζικιστάν και μάλιστα να είμαι επικεφαλής. Ήμασταν εκεί πέρα για να παρακολουθήσουμε τις εκλογές για την κατοβουλή του Τατζικιστάν. Το Τατζικιστάν είναι μια πολύ φτωχή χώρα η οποία μεταξύ του 1992 και 1997 είχε έναν αιματηρότατο εμφύλιο πόλεμο που τελείωσε με μια συμφωνία για να μοιραστεί η εξουσία στην χώρα. Το Λαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα παρέμεινε στην εξουσία, η ιδέα αντιπολίτευση που συμπεριλάμβανε και το μετρεοπαθές κόσμα της Ισλαμικής Αναγέννησης και ορισμένα άλλα κόμματα, αναγνωρίστηκε. Πήγαμε λοιπόν στην ε, Ντουσάνμπεϊ πριν από τις εκλογές, με τις εκλογικές αρχές, με πολιτικά κόμματα, με τον τύπο, μη κυβερνητικέ οργανώσεις και με τις ε, διπλωματικές ε, αρχές. Εκεί πέρα γνωρίσαμε τον κρατικό μηχανισμό και τις ε, την ατμόσφαιρα που επικρατούσε. την ίδια την ημέρα των εκλογών επισκεφθήκαμε διάφορα εκλογικά κέντρα από την έναρξη της ε, ψηφοφορία μέχρι και το κλείσιμο των εκλογικών κέντρων και την καταμέτρηση των ψήφων. Ήμασταν στο κέντρο και στην περιφέρεια της ε, Ντουσάνμπεϊ αλλά και στην πόλη Κουργαντούμπε και στην περιοχή μέχρι τα αφγανικά σύνορα. Η αντιπροσωπεία μας ήταν τμήμα της μεγάλης ε, αποστολής παρατήρησης των εκλογών του ΟΑΣΕ, της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΟΑΣΕ, σε συνεργασία με το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΑΣΕ. Είχαμε εξαιρετική συνεργασία και εξαιρετικό κλίμα. Η δε σχέση με τον δόκτωρα Πάντριξ, επικεφαλή του ΟΝΤΙΡ και τον πρέσβηνο κύριο Λάτσιξ ήταν αποτελεσματικότατη και η αντιπροσωπεία εργάστηκε πολύ επικοδομητικά πλην ορισμένων μικρών περιπτώσεων και καταλήξαμε γρήγορα σε μια κοινή θέση διαφορετική ήταν η σχέση με την κοινοβουλευτική συνέλευση του ΑΣΕ από την αρχή έως το τέλος ήταν τεταμένη η κατάσταση και είχαμε αρνητική διάθεση κάτι το οποίο μας δυσκόλεψε στη δουλειά μας. Ο λόγος ήταν πιθανός η δύσκολη σχέση μεταξύ των δύο οργάνων του ΑΣΕ. Σύμφωνα με τις ε, παρατηρήσεις μου, η Υπηρεσία Δημοκρατικών Θεσμών ε, και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατέβαλε κάθε προσπάθεια. Η δε κοινοβουλευτική συνέλευση δεν τα θεώρησε αυτά επικοδομητικά. Τώρα κάποιες παρατηρήσεις για το πώς κύλησαν οι εκλογές. Όσον αφορά την ε, ειρηνική και επικοδομητική ατμόσφαιρα, εντυπωσιαστήκαμε και κατά τη διάρκεια της εκστρατείας και κατά την ημέρα της ψηφοφορίας. Αυτό νομίζω είναι ένα θετικό βήμα για την εθνική συμφιλίωση και ενότητα. Από την άλλη όμως νομίζω αποτελεί και απόδειξη της έλλειψης πολιτικού διαλόγου για το πως πρέπει να αντιληφθεί το κοινό ότι οι εκλογές είναι κάτι περισσότερο από έναν σκέτο εκλογικό αγώνα και για το πώς θα υπάρξει μια κατανομή εξουσίας πέρα από την ήδη υπάρχουσα. Επίσης παρατηρούμε πως οι αρχές του Τατζικιστάν αμέλησαν να αναθεωρήσουν το εκλογικό δίκαιο μετά τις συμβουλές που δόθηκαν από την αντιπροσωπή του 2005. Οι δε συμβουλές αυτές αφορούσαν τη σύσταση εθνικού εκλογικού μητρώου των ε, περιορισμών τον περιορισμό των πολύ υψηλών τελών που πρέπει να πληρώσουν κόμματα και ανεξάρτητοι υποψήφοι και το τι γίνεται ε, με ψηφοφόρους οι οποίοι δεν είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους. Παρατηρήσαμε λοιπόν κάποιες παρατυπίες όπως οικογενειακές ψηφοφορίες ή το ότι δεν ήταν τελείως μυστική η ψηφοφορία αλλά δεν υπήρχε νομίζω κάποιο σημάδι προφανούς νοθείας ή παρατυπίες αυτές ε, παρατηρήθηκαν και από τους υπόλοιπους διεθνείς ε, παρατηρητές και αναφέρονται στις εκθέσεις τους. Τώρα, για το πολιτικό πλαίσιο, σημαντικό είναι να σημειώσουμε πως η αντιπροσωπεία μας υποστηρίζει τα προσωρινά αποτελέσματα της εκλογικής ε, επιτροπής και επιπλέον είχαμε μία ημέρα μετά τις εκλογές την δυνατότητα να δούμε τι γίνεται με την ε, καταμετρήση και την ε, κατανομή και υπογραμμίζουμε το ότι κατά την ημέρα των εκλογών δεν παρατηρήσαν πίεση στους ψηφοφόρους ή βία. Επιπλέον δεν είδαμε κάποια δυσαρέσκεια μεταξύ των ψηφοφόρων για τον τρόπο διεξαγωγής των εκλογών. Τονίσαμε την σημασία της σταθερότητας για το Τατζικιστάν και τους πολίτες του. Η σταθερότητα αυτή θα πρέπει να διατηρηθεί και ταυτόχρονα θα πρέπει να οικοδομηθούν περισσότερες δημοκρατικές διαδικασίες και θεσμικά όργανα και εδώ πρέπει να συνεισφέρουμε εμείς. Είμαστε υπέρ με ενός ε, ισχυρότερου πολιτικού διαλόγου που θα συμπεριλαμβάνει και νέους και γυναίκες και ενθαρρύνουμε το νέο κοινοβούλιο του Τατζικιστάν να γίνει ένα νέο δημοκρατικό φόρουμ όπου θα λαμβάνουν τις σημαντικότερες πολιτικές αποφάσεις της χώρας. Σημειώνουμε πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσω της αντιπροσωπείας του για την Κεντρική Ασία είναι διατεθειμένο να ενισχύσει τη συνεργασία με το Τατζικιστάν και απευθύνουμε πρόσκληση, απευθύναμε πρόσκληση στο νέο κοινοβούλιο να επισκεφθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης ε, Είδαμε και εμείς τα αποτελέσματα της νέας νομοθεσίας που ετέθη ισχύ από 1η πρώτου 2010 επίσης. Ε, τα αποτελέσματα νομίζω ανταποκρίθηκαν τελικά στις ε, προσδοκίες. Το Λαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα υπό την Προεδρία του Προέδρου Ραχμάν ε, έλαβε γύρω στο 72% των ψήφων και 53% από τις 63 ε, έδρες. Το ΔΕ Ισλαμικό κόμμα, το οποίο είναι το μόνο νόμιμο Ισλαμικό κόμμα της Κεντρικής ε, Ασίας, ε, έλαβε δεύτερη θέση με 7,7% και δύο έδρες. Και άλλα μικρότερα κόμματα εκπροσωπούνται στο Κοινοβούλιο. Το ΔΕ κόμμα της Ισλαμικής Αναγέννησης και το Σοσιαλδημοκρατικό κόμμα προσέφηκαν στα δικαστήρια κατά του αποτελέσματος καθώς δεν ε, κέρδισαν ε, έδρες στην, ε, στον πρώτο γύρο και βεβαίως είχαμε 13 Μαρτίου τον δεύτερο γύρο τον οποίο δεν παρατηρήσαμε. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω ολόκληρη την ομάδα, τον κύριο Χαντούτσι και από την γραμματεία των αντιπροσωπιών για την, αντιπροσω... για την προετοιμασία και την υποστήριξη. Ήταν εξαιρετική εργασία τους. Θα ήθελα επίσης να υπενθυμίσω εδώ πέρα την σημασία του Τατζικιστάν και για εμάς. Στο ίδιο το Τατζικιστάν ζουν 7,6 ε, εκατομμύρια άνθρωποι Τατζίκοι Ουσμπέκοι. Στο Αφγανιστάν ζουν 10 εκατομμύρια Τατζίκοι. Γι' αυτό πρέπει να σκεφτούμε πόσο σημαντική είναι αυτή η χώρα για μας. Σε ολόκληρη την Κεντρική Ασία μιλάμε για την προβληματική του νερού και εκεί πέρα το Τατζικιστάν είναι ίσως ο σημαντικότερος παίκτη. Οπότε εγώ προτείνω να πάρουμε στα σοβαρά αυτή τη συμφωνία εταιρική σχέσης και να βασιστούμε σε μια σωστή βάση για τη συνεργασία μας με το Τατζικιστάν. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Γέγκελ για την έκθεσή σας. Κανονικά θα έπρεπε να πάρει το λόγο ο κύριο Πέτερλε, ο οποίο είναι απόνομο οπότε δεν έχει ζητήσει κάποιο άλλο το λόγο, περνάμε στο επόμενο θέμα. Ένωση για τη Μεσόγειο. Ο κύριος Πεγιό είναι εισηγητής. Πρώτα θα πάρει το λόγο ο συνάδελφος Πεγιό. Είναι η πρώτη συζήτηση, η πρώτη ανταλλαγή απόψεων γύρω από την υπόθεση αυτή. Γνωρίζουμε το θέμα, το Κοινοβούλιο το Φεβρουάριο του 2009 μέσω της εκθέσεως της ε, κυρίας Πασκουαλίνα Ναπολιτάνο εξέφρασε τις θέσεις της ε, μετά από τις συναντήσεις κορυφής του Παρισιού και της Μασαλίας. Κάποια στοιχεία από την έκθεση αυτή ήταν ιδιαίτερα χρήσιμα και τα λάβαμε υπόψη μας. Το πλαίσιο έχει αλλάξει βέβαια αρκετά. Υπάρχουν κάποια βήματα προόδου, μετά από δύο χρόνια μπλοκαρίσματος φαίνεται ότι τα πράγματα ξεκίνησαν πάλι και σκοπεύουμε τον μήνα Ιούνιο να οργανωθεί η συνάντηση κορυφής αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων στη Βαρκελόνια. Πρόκειται για ένα πρώτο θετικό βήμα. Για λόγους χρονοδιαγράμματος αλλά και για στρατηγικούς λόγους που αφορούν τον πολιτικό προσανατολισμό της Ευρώπης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να εκφραστεί είδαμε όταν συζητούσαμε τις σχέσεις ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις Ηνωμένε Πολιτείε, μετά όταν συζητούσαμε τις σχέσεις της Ένωσης με τη Λατινική Αμερική, μιλάμε για έναν κόσμο με πολλούς πόλους πλέον και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σαφές ότι θα πρέπει να καταστήσει προτεραιότητα και τις σχέσεις της με τις χώρες του Νότου και τις Λεκάνης της Μεσογείου. Υπάρχουν οικονομικές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν, υπάρχουν δημογραφικές προκλήσεις, γεωστρατηγικές, οι οποίες βαρύνουν την διαδικασία. Είναι μια ζώνη η οποία θα μπορούσε να είναι μια ζώνη ευημερίας για μας. Είναι κάτι το οποίο προφανώς θα έχει και δημοσιονομικές συνέπειες. Θα πρέπει να πω προς το σύνολο των συναδέλφων τους ευχαριστώ για τις ήδη αποφόρες συζητήσεις που είχα μαζί τους, ότι η έκθεση κανονικά θα πρέπει να ψηφιστεί στην Ολομέλεια του μηνός Μαΐου και έτσι θα μπορέσει να εκφραστεί το Κοινοβούλιο πριν από τη συνάντηση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Μεσογείου. Σε αυτή την πρώτη φάση λοιπόν καταλήξαμε καταρχάς σε ορισμένες βασικές αρχές έχοντας τις εμπειρίες ιδιαίτερα και από τα δύο τελευταία χρόνια γύρω από την οργάνωση της έκθεσης αυτής και την πολιτική της γραμμή. Η πρώτη βασική αρχή, η συνάδελφος ε, Φλότρο η οποία έπρεπε να φύγει, συζητούσε το θέμα αυτό με μένα και αναφέρθηκε σε αυτά που συζητήθηκαν το Σαββατοκύριακο και στο Αμάν. Η διαδικασία αυτή δεν είναι κάτι το οποίο ξεκίνησε εκ του μηδενός, αλλά είναι καρπός μιας διαδικασίας η οποία γεννήθηκε με τη διαδικασία της Βαρκελόνης ήδη από το 1985. 95, συγγνώμη. Η δεύτερη βασική αρχή και βλέποντας ποιες είναι και οι εβδομάδες οι τελευταίες που είναι αρκετά δύσκολες, δεν θα πρέπει να καταστεί όμοιρος η διαδικασία αυτή της πολιτικής συγκυρίας. Για λόγους διαφορών και συγκρούσεων ανάμεσα σε ορισμένους από τους εταίρους. Πιστεύουμε ότι η ολοκλήρωση συγκεκριμένων προγραμμάτων οικονομικών, εκπαιδευτικών, κοινωνικών θα μπορέσει να λειτουργήσει σαν ένας παράγων προώθησης της ειρήνης και ότι δεν θα πρέπει στα πλαίσια της Μεσογειακής Ένωσης να στοχεύουμε ε, στην επίλυση ε, του Μεσανατολικού. Θα πρέπει λοιπόν εμείς να πιέσουμε προς την υλοποίηση όλων αυτών των μεγάλων προγραμμάτων. Τρίτον, θα πρέπει στα πλαίσια του τρόπου λειτουργίας αλλά και στα πλαίσια του τρόπου λήψης αποφάσεων της μεσογειακής αυτής διαδικασίας να εισαγάγουμε θα έλεγα δημοκρατία και διαφάνεια. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωμεσογειακή διάσκεψη θα πρέπει να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε και σε επίπεδο κοινοβουλευτικού ελέγχου στα πλαίσια της Ένωσης για τη Μεσόγειο. Σχετικά τώρα με τις δημοσιονομικές προοπτικές 2014-2020 και είναι κάτι το οποίο θα συζητηθεί ήδη τον μήνα Ιούνιο, θα πρέπει να διασφαλίσουμε τις χρηματοδοτήσεις που απαιτούνται. Διότι τη στιγμή κατά την οποία η Ευρώπη βρίσκεται σήμερα σχετικά πίσω θα έλεγα σαν επενδύτρια περιοχή, στην περιοχή Ακούγονται πολλά λόγια, προχωρούμε σε πολιτικές συνεργασίες, προχωρούμε σε θεσμικές συνεργασίες, αλλά δεν ακολουθούν τα χρήματα και οι πιστώσεις. Τότε στην περίπτωση αυτή τα αποτελέσματα θα είναι περισσότερο αρνητικά από όσο θα μπορούσαμε να φανταστούμε και θα υπάρξει μια βαθύτατη απογοήτευση για το ρόλο μας. Λοιπόν αυτές είναι οι βασικές γραμμές της έκθεσης. Τρει είναι οι βασικές απαιτήσει και τρία είναι τα βασικά μηνύματα τα οποία θα πρέπει να απευθύνουμε σε αυτούς που θα ασχοληθούν με την δημιουργία αυτής της μορφή συνεργασία. Καταρχά θα πρέπει να υπάρξει ένα θεσμικό μήνυμα. Θα πρέπει να διασφαλιστεί η δημοκρατική νομιμότητα στα πλαίσια της διαδικασίας λειτουργίας της Ένωσης αυτής. Και έτσι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωμεσογειακή Διάσκεψη που θα έχουν ε, μια γραμματεία και θα χρηματοδοτηθούν κατάλληλα και με αυτό ασχολήθηκε ο συνάδελφος Πιτέλα. Θα πρέπει να συνδεθούν με τη διαδικασία αυτή, να εμπλακούν στη διαδικασία αυτή και θα πρέπει οι δύο γενικοί γραμματείς να έχουν την δυνατότητα εργασίας. Είναι ένα από τα θέματα τα οποία τίθενται εδώ. Αυτό το σχήμα που θα δημιουργήσουμε θα είναι θα έλεγα ένα σχήμα ανευπεριεχομένου ή θα δώσουμε τα μέσα στη Γενική αυτή Γραμματεία να μπορέσει να φέρει εις πέρα στην πολιτική. Τρίτον θα πρέπει να εμπλέξουμε εδώ και την κοινωνία των πολιτών όπως επίσης και την Επιτροπή των Περιφερειών και η οποία σαφώς και θα πρέπει να ε, συμμετέχει με κάποιο τρόπο στις εργασίες και της ΑΠΕΜ και της Ένωσης γενικότερα. Λοιπόν, αυτά είναι τα πρώτα στάδια τα οποία θα πρέπει να διανύσουμε. Χρήζουν διευκρινήσεων. Αυτό θα πρέπει να γίνει ε, με συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το δεύτερο στάδιο είναι τα προγράμματα. Υπάρχουν έξι προγράμματα τα οποία έχουν ήδη γίνει αντικείμενο επιλογής εξ αρχής. Τα έξι αυτά προγράμματα θεωρούνται ενδιαφέροντα από όλους, δεν δημιουργούν προβλήματα, βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια υλοποίησης. Θα πρέπει το ταχύτερο δυνατόν να προσθέσουμε και άλλα προγράμματα στον τομέα των εκπαιδευτικό, ανταλλαγής φοιτητών, πολιτιστικά προγράμματα, και να ασχοληθούμε και με τον γεωργικό τομέα, να μπορέσουν να υπάρξουν κάποιες ανταλλαγές εμπειριών οικονομικές σχετικά με την εμβέλεια θα έλεγα δράσης της Ένωσης για τη Μεσόγειο. Και ένα τελευταίο σημείο. Ίσως μαζί με το θεσμικό ένα άλλο θέμα να είναι εξίσου επίγον. Είναι οι εξελίξεις ε, μέσω της συνθήκης της Λισαβόνας οι εξελίξεις σε επίπεδο δημοσιονομικών αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί έτσι ώστε να αποφασίσουν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων τις χρηματοδοτήσεις που απαιτούνται ήδη τον μήνα Ιούνιο. Θα πρέπει επίσης τα χρήματα τα οποία θα δοθούν για την πολιτική αυτή μέχρι το 2013 να μην αφαιρεθούν από άλλες πολιτικές όπως την πολιτική γειτονίας θα πρέπει επίσης να γίνει σεβαστός ο στόχος ή μάλλον η αρχή λειτουργίας 2 τρίτα 1 τρίτο και θα πρέπει επίσης όλα αυτά να συνοδευτούν από συγκεκριμένες υποχρεώσεις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες και αυτό θα πρέπει να φανεί στις δημοσιονομικές προοπτικές 2014-2020. Ήδη λοιπόν από τον Ιούνιο θα πρέπει οι κυβερνήσεις να προχωρήσουν σε δεσμεύσεις οι δεσμεύσεις αυτές ε, να ακολουθηθούν από επίσημες προτάσεις. Έχουμε ακούσει κάποιες πρώτες τέτοιες προτάσεις, όπως ε, η ιδέα μιας ε, χάρτας διασφάλισης των επενδύσεων και κάποιες άλλες αποφάσεις οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν για να διασφαλιστεί η οικονομική εγκυρότητα της συγκεκριμένης προσπάθειας. Λοιπόν, κλείνοντας, Μιλάμε για μια έκθεση η οποία θα πρέπει να είναι έκθεση του συνόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Χαρακτηρίζεται από ένα πνεύμα ανοίγματο και από μένα προσωπικά. Ευχαριστώ ήδη τους ε, εισηγητές γνωμοδότες από τις άλλες αρμόδιες επιτροπές. Την επόμενη εβδομάδα θα συγκεντρωθούν και οι υπόλοιπες τροπολογίες όλες θα γίνουν, ε, είναι καλοδεχούμενες από πλευράς μου. Βέβαια έχουμε κάποιες επιφυλάξεις ε, σχετικά με το μέγεθος της έκθεσης, αλλά περιμένουμε ακόμα περισσότερες τροπολογίες. Θα υπάρξει μια σε περισσότερο βάθος συζήτηση πάρα πολύ σύντομα. Σας ευχαριστούμε. Έχουμε ένα μακρύ κατάλογο μιλητών, όμως έχουμε ε, χρονικούς περιορισμούς. Σας παρακαλώ λοιπόν 1,5 λεπτό το πολύ 2 λεπτά ο καθένας. Πρώτος μιλητής. Συνάδελφος Μίλαν Μον, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστούμε τον εισηγητή συγχαρτήρια όχι μόνο για την έκθεσή σας αλλά ε, για την καρτεσιανή θα έλεγα λογική που χαρακτηρίζει την αιτιολογική έκθεση. Και εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα της Ευρωμεσογειακής Ζώνης. Και κοιτάξτε, εδώ δεν θα πρέπει να είμαστε όμοιροι ε, των ιστορικών συγκρούσεων που δεν μας αφήνουν να σημειώσουμε πρώτα, πώς έγινε με την ε, Βαρκελόνη. Πολύ σύντομα, τώρα από το εξή. Στο β της αιτιολογικής έκθεσης, δεν ξέρω κατά πόσον το μήνυμα, το μήνυμά μας είναι ότι δεν μας απασχολεί το θέμα της μετανάστευσης. Όχι, η μετανάστευση πρέπει να μα απασχολήσει στι ε, ευρωμεσογειακέ σχέσει και δεν νομίζω ότι είναι σωστό να πούμε ότι μέχρι στιγμή αυτό το οποίο μα ε, απασχόλησε ε, βασικά ήταν η ασφάλεια ή η μετανάστευση. Α είμαστε ρεαλιστέ. Από τι τρει-τέσσερι συμβάσει διαπραγμάτευση σε θέματα επανεισδοχή με τι μεσογειακέ χώρε και εδώ σκέφτομαι την Τουρκία, το Μαρόκο ή την Αλγερία. Έξι-εφτά χρόνια διαπραγματευόμαστε αυτέ τι συμφωνίε και δεν έχουμε ολοκληρώσει όπω με το Πακιστάν, με την Ουκρανία ακόμα και με τη Ρωσία. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό. Ούτε καν είναι το κατάλληλο μήνυμα το οποίο θα πρέπει να εκπέμψουμε. Άλλο συγκεκριμένο θέμα. Στο 2. Βεβαίω τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι θεμελιώδει ε, ελευθερίε ε, και η πρόθεση δημοκρατία είναι βασικά σημεία. Σα υπενθυμίζω το άρθρο 8 τη Νέα Συνθήκη τη Ένωση ε, τονίζει ε, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, σε σχέση μα με τι γειτονικέ χώρε. Κοιτάξτε, στην ισπανική μετάφραση αναφέρεται ότι ε, όλα αυτά θα πρέπει να αποτελέσουν το βασικό, τον κεντρικό στόχο, ε, τον κεντρικό άξονα. Όχι ένα κεντρικό άξονα, αλλά όχι τον κεντρικό άξονα, γιατί με απασχολούν και άλλα θέματα που έχουν να κάνουν σχέση με τη, Μεσογεία, με τη Μεσόγειο. Η ευημερία, για παράδειγμα, η χρηστή διακυβέρνηση, οι συνολικέ παγκόσμιε προκλήσει. Το να πούμε λοιπόν ότι το επίκεντρο βασικό άξονα είναι η μετανάστευση, νομίζω ότι δεν είναι σωστό. Τρίτο σχόλιο και τελειώνω, Πρόεδρε. Στο 10. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό το εναρμόνιση των θέσεων σε, σε, στον αγροτικό τομέα. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να περάσουμε το μήνυμα ότι θα πρέπει να θεσπίσουμε κάποια ελάχιστα κοινωνικά, περιβαλλοντολογικά πρότυπα, φυτογειονομικά κτλ. όσον αφορά τη γεωργική παραγωγή. Αυτό θα πρέπει να είναι κοινό. Αυτά και Πρόεδρε και ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Κόπα, ε, ε, ξέρω ότι τα πάτε πολύ καλά, είστε πολύ σύντομοι πάντα. Πρόεδρε, θέλω να συγχαρώ τον ε, συνάδελφο Πηγιών για την εξαίρετη έκθεσή του, που πιάνει το νήμα της περσινής έκθεσης Ναπολιτάνο, που συντάχθηκε μετά τη σημαντική απόφαση του Παρισιού για τη μετεξέλιξη της συνθήκης της, της διαδικασίας Βαρκελόνης. Θέλω να επισημάνω τρία σημεία πάνω στα οποία έχω σκοπό και να καταθέσω κάποιες τροπολογίες. Πρώτο σημείο είναι ότι αμέσως μετά τα τραϊκά γεγονότα στη Γάζα ε, είχαμε καταδικάσει την εισβολή ως ε, σοσιαλιστές και δημοκράτες και την παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και είχαμε τονίσει ότι η Ένωση για τη Μεσόγειο οφείλει να συμβάλλει στο διάλογο και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης με στόχο πάντα την επίλυση του μεσανατολικού προβλήματος. Ε, γι' αυτό το λόγο είναι σημαντικό που επαναλαμβάνεται η Εκκλησία μας στο άρθρο 3 του κειμένου που συζητάμε σήμερα επειδή όμως όλοι γνωρίζουμε τις δυσκολίες που περνάει η προσπάθεια να ξαναρχίσει η διαδικασία και ε, της επανέναρξης διαλόγου στη Μέση Ανατολή, θα ήθελα να προσθέσουμε κάτι που να υποδηλώνει τη σαφή στήριξή μας σε αυτά τα πολύ δειλά βήματα που γίνονται και με όλες δυσκολίες. Δεύτερο σημείο είναι ε, θα ήθελα να υπάρξει μεγαλύτερη προσοχή για τα ζητήματα ισότητας και δικαιωμάτων γυναικών ε, όπως ξέρετε τον περασμένο νοέμβρη στο μαρακές έλαβε χώρα η δεύτερη ευρωμεσογειακή υπουργική διάσκεψη σχετικά με την ενδυνάμωση των γυναικών στην κοινωνία με αποτέλεσμα να υπάρξει δέσμευση όλων των συμμετεχόντων υπουργών ότι θα προωθήσουν de jure και de facto την ισότητα. Πιστεύω λοιπόν ότι θα έπρεπε να εκφράσουμε τη στήριξή μας σε αυτή τη δήλωση και γιατί όχι να ζητήσουμε και την υιοθέτηση ενός προγράμματος στήριξης της γυναικείας επιχειρηματικότητας αλλά και της παρουσίας του στο δημόσιο βίο. Τρίτο και τελευταίο μου σημείο είναι πάλι στο θέμα των προγραμμάτων. Ε, πιστεύω ότι πρέπει να εκφράσουμε σαφώς τη δυσαρέσκειά μας για την καθυστέρηση έναρξή του και να υπογραμμίσουμε ότι αυτά αποτελούν την πεμπτουσία και την προστιθέμενη αξία της Ένωσης για τη Μεσόγειο. Θα ήθελα επίσης να υπάρξει μια αναφορά που να δείχνει τη σημασία των περιβαλλοντικών προγραμμάτων, όπως αυτό για την απορρίπανση της Μεσογείου, στα πλαίσια του ορίζοντα 2020, και αυτό για τη διάδοση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Σε σχέση με το τελευταίο θα μπορούσαμε να καλωσορίσουμε και τα δύο συνέδρια που διοργανώνονται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Ισπανική Προεδρία σε υπουργικό επίπεδο για τον ερχόμενο Μάιο σε σχέση με το Μεσογειακό Πλάνο Ηλιακής Ενέργειας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να εκφράσω την ικανοποίησή μου από την πρώτη τοποθέτηση και το κείμενο που περιλαμβάνεται για την Ένωση για τη Μεσόγειο. Είναι ιδιαίτερα σημαντική η προσπάθεια επαναδραστηριοποίησης της Ένωσης για τη Μεσόγειο και ελπίζω ότι με όσα έχουν αναφερθεί ότι θα υπάρχει και ανάλογη χρηματοδότηση και ενίσχυση ιδιαίτερα από τους αρχηγούς των κρατών ούτως ώστε να είναι αποτελεσματική στο τέλος της ημέρας και να μην περάσουμε πάλι κάποια χρόνια αδράνειας αυτής της τόσο σημαντικής επιτροπής. Θα ήθελα να σημειώσω δύο-τρία σημεία στα οποία θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικά στην έκθεση. Πρώτον το θέμα της μετανάστευσης, το οποίο είναι σημαντικό για τις νότιες αρτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης λαμβάνοντα υπόψη ότι τα κράτη της, της Μεσογείου αριθμούν σχεδόν ένα δισεκατομμύριο πληθυσμών. Άρα τα θέματα της μετανάστευσης δεν μπορούν παρά να απασχολήσουν την Ένωση για τη Μεσόγειο όπως επίσης και διάφορα θέματα τα οποία αποτελούν προβληματικές περιοχές στη λεκάνη της Μεσογείου. Στο Μεσανατολικό, ασφαλώς η Ένωση για τη Μεσόγειο δεν θα λύσει το Μεσανατολικό, αλλά οφείλει και πρέπει να παίρνει σταθερές ε, θέσεις σε σχέση με την ανάγκη ενίσχυσης του διαλόγου για να μπορέσουμε τουλάχιστον να παρατηρήσουμε κάποια έναρξη προσπάθειας επίλυσης του Μεσανατολικού και μέσα από την άποψη ότι θα πρέπει μέσα από το κείμενο αυτό να διεκδικηθεί μια ανάλογη συμπαράσταση από τις διάφορες κυβερνήσεις που συμμετέχουν ούτω ώστε πραγματικά να δοθεί η δυνατότητα οικονομικής ενίσχυσης και πραγματικής ενίσχυσης της Επιτροπής αυτής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Επόμενος συνάδελφος, Κύριε Σομπιόλ, σας παρακαλώ να είστε σύντομα, διαφορετικά θα αναγκαστώ να ε, σας διακόπτω στις παρεμβάσεις σας. Κρίμα που είμαστε αναγκασμένοι να συζητήσουμε αυτή την έκθεση τόσο βιαστικά. Γιατί η ευρωπαϊκή πολιτική είναι μία από τι βασικέ προτεραιότητε τη εξωτερική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσα από τι 5-6 βασικέ προτεραιότητε. Αλλά από άποψη κινδύνων, από άποψη κινδύνων είναι η πρώτη από τις προτεραιότητες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πραγματικά θα έπρεπε να ζητήσουμε από την Προεδρία ε, να, αυτά τα θέματα να τα προβλέπει προς συζήτηση κάποια χρονική στιγμή όπου να έχουμε κάποια προσωπική άνεση. Θα περιοριστώ λοιπόν και θα αρκεστώ σε τρία σημεία. Πρώτα απ' όλα συμφωνώ με, την έκθεση, με το σχέδιο έκθεσης ε, του συναδέλφου. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικό έγγραφο, σαφέστατο. Νομίζω ότι εδώ, όπω ακούσαμε από τον συναδέλφο, χαρακτηρίζεται από καρτεσιανή λογική. Ναι, πράγματι, συμφωνώ. Αποτελεί μια άριστη βάση εργασία και ε, συμφωνώ επί τη ουσία με του προσανατολισμού και τι προτεραιότητε που αναφέρετε. Δεύτερον, ίσω θα πρέπει να αναφέρουμε ε, την, ε, την αραβο-ισραηλινή διένεξη. Υπάρχει μια συγκεκριμένη αναφορά στην 11η Σεπτεμβρίου και στον πόλεμο του Ιράκ και βεβαίω και το, και το αναφέρθηκε πολύ καλά η αιτιολογική σχέση, χωρί να αναφέρουμε ότι μόνο σημειωθεί η πρόοδο ε, στην ε, ειρηνευτική διαδικασία, θα υπάρξει αυτή η πολιτική κτλ. Ναι, χωρί να πούμε αυτό, ε, πάντω είναι σαφέ ότι και προ τη μία κατεύθυνση και προ την άλλη υπάρχει άμεση σχέση. Η σωστή πολιτική ευρωμεσογειακή θα μπορούσε κατά κάποιο τρόπο, έστω και σε μετροεπαθέ επίπεδο, να συμβάλλει προ την προώθηση τη αποκατάσταση των διαπραγματεύσεων, τη επαναφορά των διαπραγματεύσεων και σε μια πιο θετική προσέγγιση τη άραβο-ισραηλινή διένεξη. Δεύτερον, Ίσως αυτή η έκθεση θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελεί... Ε, εντάξει, σταματώ. Θα το συζητήσω με τον εισηγητή κατηδία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εμένα με λυπεί περισσότερο που σας αφαιρώ το λόγο, αλλά καταλαβαίνετε... Όχι, όχι. Εντάξει, ε, Πρόεδρε, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Και ε, όταν μου, λέ, όταν μου λένε να μην μιλήσω, επειδή δεν μου αρέσει και πολύ να μιλάω, σα ευχαριστώ πολύ που μου παίρνετε το λόγο. Δεν αισθάνομαι ιδιαίτερα άνετα. Λοιπόν, ευχαριστώ του συναδέλφου. Ε, θα υπάρξει περαιτέρω ε, περιθώριο για συζήτηση και όταν θα έχουμε τι τροπολογίε. Και θα συζητηθούν και οι τροπολογίε. Ε, προθεσμία 27 Απριλίου 2010. Άρα έχουμε ε, ε, χρόνο για συζήτηση και τότε. Ο κύριος Αγκουράκης έχει το λόγο. Από την ΚΟΕ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, καταρχήν έχετε δίκιο, πρέπει να είμαστε σύντομοι, αλλά να με συγχωρέσει ο εισηγητή, μίλησε πάρα πολύ, κατά τη γνώμη μου, το κείμενο το είχαμε, δεν ήταν ανάγκη να μιλήσει τόσο πολύ. Τώρα, στι παρατηρήσει μου. Πρώτη παρατήρηση κύριε Πρόεδρε, νομίζω όταν συζητάμε τέτοιου είδου ε, κείμενα, καλό είναι, θα έλεγα ότι είναι υποχρεωτικό, να έχουμε και την άποψη τη άλλη πλευρά. Δεν θέλετε να έχουμε την άποψη των κυβερνήσεων. Ωραία, Α έχουμε την άποψη των κοινοβουλίων, των χωρών ε, της ευρωμεσογειακής ε, ε, συνεργασίας. Θα ήταν πάρα πολύ ωφέλιμο για μας για να έχουμε μια πιο αντικειμενική εικόνα. Δεύτερο ζήτημα, βλέπω έναν τόνο κάπως συναγερμού, δηλαδή γίνεται κάπως λόγος ότι αυτή η σύνοδος της Βαρκελόνης θα είναι η τελευταία ευκαιρία για να σωθεί η Ένωση για τη Μεσόγειο. Εγώ βέβαια είμαι αντίθετο για ιδεολογικού και πολιτικού λόγου με την Ένωση για τη Μεσόγειο, δεν είναι το θέμα να το συζητήσουμε τώρα, αλλά με ενδιαφέρει αυτό ο τόνο κάπω ε, ε, ο επιτακτικό. Υπάρχει τέτοιο ζήτημα, υπάρχει ζήτημα δηλαδή να μα τελειώσει αυτή η διαδικασία. Και τρίτο ζήτημα, δεν θεωρώ επαρκή τι εξηγήσει τη έκθεση γιατί βάλτωσε η διαδικασία. Δεν μπορεί να πηγαίνουμε έτσι. Σταμάτησε και τώρα είμαστε σε μια καινούργια αρχή και άντε να δούμε να προχωρήσουμε. Δεν δεν, δεν είναι στο, στο επίπεδο των ευθυνών που ε, παίρνουμε και έχουμε. Χρειάζεται περισσότερη εμβάθυνση. Και τέλος, Βεβαίω δεν μπορεί να προχωρήσει αυτή η Ένωση εάν δεν αντιμετωπιστούν σωστά, ισότιμα, δίκαια τα πολιτικά ζητήματα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γιαννάκου έχει το λόγο. αλήθεια είναι ότι η έκθεση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία και θα έπρεπε να υπάρχει πολύ περισσότερο χρόνος για να τη συζητήσουμε. Ας μου επιτραπεί να κάνω μερικές πολύ σύντομες παρατηρήσεις. Η αλήθεια είναι ότι έχει ατονίσει η εστίαση στα ανθρώπινα δικαιώματα και στη δημοκρατία σε σχέση με την ε, ευρωμεσοδιακή διαδικασία και διεργασία. Δεύτερον, το σύστημα έχει αποπολιτικοποιηθεί. Αυτό αποθαρρύνει δημοκρατικές δυνάμεις πιθανών των άλλων χωρών ε, να συνδεθούν μαζί μας. Η Ευρώπη έχει χάσει το βάρος ως πολιτισμικό στοιχείο αναφορά στη Βόρεια Αφρική, κύριε Πρόεδρε. Άλλες δυνάμεις αυτή τη στιγμή παρεμβαίνουν στον χώρο της Βόρειας Αφρικής. Η σχέση με τις χώρες αυτές πρέπει να είναι ισότιμη καταρχήν, υποχρεωτικά. Απ' την άλλη πλευρά, ένα είδος ρήτρα για τα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, ισότητας των γυναικών και μη εξαίρεσή τους από τον κοινωνικό ιστό θα πρέπει να υπάρχει. Εγώ θα κάνω τροπολογίες, θέλω να συγχαρώ τον συνάδελφο για την προσπάθειά του, αλλά νομίζω ότι πρέπει ο ρόλος των γυναικών να περιγραφεί σε ιδιαίτερη παράγραφο. Ε, ποιος θα είναι πιθανόν ο ρόλος στην επίλυση της Ισραηλινοπαλαιστινιακής διαμάχης, αν μπορεί να υπάρξει κάποιος ρόλος να γίνουν κοινέ προσπάθειες για την τρομοκρατία και την παράνομη μετανάστευση. Αυτό δεν μπορεί να καταληφθεί τελείω. Είναι ζήτημα πολύ σοβαρό. Και δεν υπάρχει και καμία αναφορά στα Βαλκάνια, δηλαδή τα Βαλκάνια της Αδριατικής που έχουν μπει στην Ευρωμεσογειακή. Αυτά είναι σημεία στα οποία εγώ ήθελα να πω ότι θα προβώ σε τροπολογίες στην έκθεση αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Bene, allora il collega Agi Giorgio. Ευχαριστούμε. Το λόγο έχει ο κύριος Χατζηγεριέου. Καταρχήν ότι δυσκολεύομαι να καταλάβω πώς αυτή η Ευρωμεσογειακή Ένωση θα μπορέσει να αποφύγει τη συζήτηση πολιτικών ζητημάτων. Όση προσπάθεια και αν καταβληθεί, νομίζω ότι στο τέλος η προσπάθεια αποφυγής να αγγίξουμε τα ζητήματα που καίνε ε, μπορεί να μην βοηθήσει στο τέλος και τους ευρύτερους στόχους που έχει η, Ευρωμεσογειακή Ένωση. Το δεύτερο μου ερώτημα. Υπήρχε μια συζήτηση για το ρόλο της Τουρκίας σε αυτή την Ένωση. Υπήρχε δηλαδή μέχρι και συζήτηση αν αποδεχόταν τη συμμετοχή της σε αυτήν την ένωση. Θυμούμε ότι έγιναν και μερικές συναντήσεις ή και τηλεφωνήματα μεταξύ του κυρίου Σαρκοζή και του κυρίου Ερτογάν και θέλω να ξέρω αν υπάρχει εικόνα για το που έχουν καταλήξει τα πράγματα. Το τρίτο θέμα, θέλω να εντοπίσω και εγώ το ενδιαφέρον μου σε θέματα ισότητας ανδρών και γυναικών που πρέπει να αναδειχθούν σε αυτή την Ευρωμεσογειακή Ένωση σαν μεγάλη σημασία ζήτημα για προφανείς λόγους. Κλείνω με το εξής. Ξέρω ότι τα κράτη της Βόρειας Αφρικής ε, που περιβρέχονται από τη θάλασσα της Μεσογείου ζήτησαν οικονομική στήριξη από την Ευρώπη προκειμένου να στρατολογήσουν αστυνομικούς για να ελέγχουν την μετανάστευση που γίνεται από σημεία όπου δεν λαμβάνει η χώρα κρατικός έλεγχος. Υπάρχει κάποια εξέλιξη σε αυτό. La, Ο εισηγητής έχει το λόγο, ο κύριος Πεγιόν. Ευχαριστώ συνάδελφοι για τις παρατηρήσεις σας. Θα προτιμούσα να είχαμε περισσότερο χρόνο, να έχω εγώ το χρόνο να ακούσω περισσότερο από τους συναδέλφους. Εν πάση περιπτώσει ε, ακούστηκαν πολλά και για τις σχέσεις μας με το Μαγκρέμπ. Υπάρχει εμπειρογνωμοσύνη σε αυτή την αίθουσα και ελπίζω ότι η επόμενη συνάντηση και η επόμενη συζήτηση θα επιτρέψει να γίνει μια συζήτηση αντίστοιχη χρονικά με τη σημασία του θέματος. Δεν ήξερα, μακρηγόρησα και εγώ, έκανα λάθος και στέρισα χρόνο από πολλούς από εσάς. Η Ένωση για τη Μεσόγειο λοιπόν είναι μια διαδικασία η οποία είναι ανεξάρτητη και δεν αντικαθιστά τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στις χώρες του Νότου. Η Ένωση για τη Μεσόγειο δεν έχει έρθει δηλαδή για να ρυθμίσει όλα τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν ανάμεσα στην Ένωση και τις υπόλοιπες χώρες. Αν το βλέπαμε έτσι τότε θα ήταν ο καλύτερος τρόπος για να την καταδικάσουμε αν ζητήσουμε από την Ένωση να ρυθμίσει τα προβλήματα της μετανάστευσης σαν παράδειγμα. Αν ζητήσουμε από την Ένωση να ασχοληθεί με θέματα με τα οποία ασχολούνται άλλα ευρωπαϊκά όργανα ή να ασχοληθεί με το μεσανατολικό ειδικά, τότε πραγματικά διαρωτώ ποιο θα είναι το μέλλον της. Εμείς θέλουμε συγκεκριμένα προγράμματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οικοδομήθηκε πάνω στην ε, Ένωση ε, για τον Άνθρακα και το χάλιβα, σε συγκεκριμένα προγράμματα λοιπόν. Πρέπει να βασιστούμε σε αντίστοιχα συγκεκριμένα πράγματα. Αν δεν το κάνουμε αυτό θα την καταδικάσουμε την Ένωση αυτή και δεν θα ακουστεί και η φωνή μας γιατί θα θεωρηθεί ότι δεν ασχολούμεθα σοβαρά με το θέμα. Πρέπει να είμαστε λοιπόν προσεκτικοί στις θέσεις τις οποίες θα λάβουμε και δεν ξεκινάει η συζήτηση εκ νέου. Έχουμε κάποια σορευμένη εμπειρία από το τι συνέβη τα δύο περισσότερα χρόνια. Αν κάποιος πιστεύει ότι θα τα λύσει όλα αυτά τα προβλήματα τώρα, θα μπλοκάρει τη διαδικασία. Και τη στιγμή κατά την οποία προσπαθήσαμε να ξεμπλοκάρουμε τα πράγματα και με την Τουρκία, τότε θα πρέπει η Ευρώπη να μην κάνει τα λάθος να, να, να γύρει καινούρια εμπόδια. Βέβαια το θέμα της μετανάστευσης δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε, απλά έχουμε βρει ένα τρόπο να το κάνουμε, λέγοντας ότι οι συζητήσεις με τον νότο της Μεσογειακής Λεκάνης δεν μπορούν να περιορισθούν στη συζήτηση του θέματος του μεταναστευτικού. Γιατί έτσι θα αγνοήσουμε τα συγκεκριμένα προγράμματα και τους συγκεκριμένους τομείς τους οποίους μπορεί να υπάρξει πρόοδος. Θα πρέπει επίσης να εμβαθύνουμε το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είναι κάτι στο οποίο επανερχόμεθα συστηματικά, δεν εκπλήσει αυτό κανέναν και ταυτόχρονα εμείς δεν θα πρέπει να θεωρήσουμε το συγκεκριμένο θέμα τον βασικό άξονα της Ένωσης για τη Μεσόγειο. Η οικονομική ανάπτυξη, οι πολιτιστικές εξελίξεις, η συνεργασία, είναι θέματα συγκεκριμένα και πάνω σε αυτά θα οικοδομηθεί η πορεία μας. Για την ισότητα ανδρών γυναικών προφανώς και πρέπει ε, να την τονίσουμε, αλλά δεν είμαστε στα πλαίσια της πολιτικής γειτονίας όπου θέτουμε περιορισμούς και προϋποθέσεις. Είμαστε στα πλαίσια μιας διμερούς συνεργασίας δεν βάζουμε προϋποθέσεις. Λέμε ότι θα πρέπει να αναπτύξουμε κάποιες συγκεκριμένες πολιτικές, αλλά δεν βάζουμε τις προϋποθέσεις που βάζουμε στις υπόλοιπες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τέλος, θα πρέπει να επιβεβαιώσουμε την πολιτική μας βούληση σύμφωνα με την οποία η διαδικασία της Ένωσης για τη Μεσόγειο θα πρέπει να συνεισφέρει στην ειρήνη στη Μέση Ανατολή Υπάρχουν και άλλες βέβαια τέτοιου είδους συγκρούσεις τις οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε σε κάποια άλλη φάση αλλά εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί έτσι ώστε να μην βαρύνουμε τη βάρκα με τέτοιο τρόπο που θα την εμποδίσει να προχωρήσει. Αυτά. Για τα γεωργικά θέματα συμφωνώ μαζί σας, θα πρέπει να διευκρινίσουμε καλύτερα αυτά τα οποία λέγουμε και όπως σας είπα προηγουμένως θα ήθελα ο καθένας από εσά να νιώσει απόλυτα άνετα να συνεισφέρει στην έκθεση αυτή θα πρέπει να έχουμε περισσότερο χρόνο τις επόμενες εβδομάδες για να συζητήσουμε τις τροπολογίες που καταθέσατε ή θα καταθέσετε. Προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών είναι 24η Μαρτίου στις 12 το μεσημέρι. Ευχαριστώ. Ah ouais.